So, Kolleginnen und Kollegen, wir fangen an. Ich begrüße, ich begrüße zwei Σας καλημερίζω άλλους δύο, α, τους δύο συναδέλφους που είναι εδώ. Πρέπει να αρχίσουμε. Έχουμε ένα αρκετά πυκνό πρόγραμμα και θέλω να σας ανακοινώσω ότι εκτός από τα εσθονικά και τα μαλτέζικα έχουμε όλες τις γλώσσες, διερμηνίες και για τα απόγευμα. Δεύτερον, στις 28 του μηνός, δηλαδή σήμερα, στις 11 η ώρα, Υπάρχει ένα σεμινάριο από τις 12.30 μέχρι τις 4 παρατέταρτο στην αίθουσα PAS 12.07 από τον Κλάινος Βίρμαρτ και τον Άλαος Πέτερ και έχουμε και μια ομάδα επισκεπτών στην αίθουσά μας, 8 δημοσιογράφους που θα έρθουν το απόγευμα από τις 3 ε, με τις 6.30 τους έχει καλέσει η Ιολάντα Χίπνερ και αύριο έχουμε φοιτητέ του 3ου και 4ου έτους της ε, εφηρμοσμένης επιστήμης του Πανεπιστημίου Λιβάν της Ολλανδίας. Έχουμε και εκπροσώπους της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας της ΣΑΝΚΟ από την Κομισιόν. Τέταρτη ανακοίνωση. Η αντιπροσωπεία του ΕΛΚ για την Νότια Ασία μας κάλεσε αύριο στις 29 Δεκάτου, στις 11.30 μέχρι τις 12.30 να συμμετάσχουμε σε μία συνεδρίαση για την COP18 ανταλλαγή απόψεων και αύριο έχουμε μία ψηφοφορία βεβαίως το ξέρω και ίσως από όλες τις ομάδες μπορεί να έρθει ένας. Ελπίζω από κάθε ένας, ένας να μπορεί να συμμετάσχει. Τώρα, <clears throat> προχωράμε στην έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Δεν υπάρχουν ε, αλλαγές, τροποποιήσεις, ίσως αύριο να υπάρχει κάτι, σήμερα δεν έχουμε. Ε, έγκριση των πρακτικών και εκεί δεν υπάρχει τίποτα καινούριο και φτάνουμε ήδη στο 4, προετοιμασία της COP16. ΣΥΤΕΣ. Εδώ έχουμε σήμερα ένα προσκεκλημένο τον Ζων Σανκλόν, ο οποίος θα μας μιλήσει για την τρέχουσα κατάσταση και δεν θέλω να σας καθυστερήσω περισσότερο, αλλά θέλω να του δώσω το λόγο για να μας ενημερώσει για τη σύμβαση. Thank you very much, Chair, and good morning all. And... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που με προσκαλέσατε στη συζητήση σας σήμερα το πρωί. Να ευχαριστήσω και την, από πλευράς τη γραμματείας τη ΆΕΤΗΣ και της όλης κοινότητα για τη στήριξη που μας έχετε δώσει ως Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να υλοποιηθεί η σύμβασή μα, όπου συμμετέχετε με τα 27 κράτη-μέλη αλλά και συλλογικά, με την εντολή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Μάρτιο του χρόνου θα έχουμε τη 16η συνάντηση τη Σύμβαση των Μερών και θα γιορτάσουμε και τη 40 ε, επέτειο από την υιοθέτηση της ε, Σύμβασης το Μάρτιο του 1973 στην Ουάσιγκτον ε, των Ηνωμένων Πολιτειών. Η επόμενη συνεδρίασή μας το Μάρτιο θα είναι εξαιρετικά σημαντική για την τύχη πολλών ειδών του πλανήτη και τις ε, δυνατότητες που θα έχουν να επιβιώσουν. Έχουμε τις με πιο σοβαρές περιπτώσεις ε, λαθροθυρίας τα τελευταία 10 με 20 χρόνια κατά πολλών ειδών και στην παράνομη θανάτωση ελεφάντων και ενοκαίνων έχουμε πολλές σοβαρές περιπτώσεις με 550 περιπτώσεις ε, προστασίας φέτος. Η λαθροθυρία πρέπει να αναχαιτιστεί εάν θέλουμε τη βιωσιμότητα. Και τώρα έχουμε περάσει στην, ε, στο επαγγελματικό κυνήγι των ειδών αυτών με θανάτωση αγελών με 10 περιπτώσεις μόνο φέτος στην Κένια. Υπάρχει διαφορά των τοπικών υπαλλήλων, των λαών και όλα αυτά με διοχέτευση χρήματος. Θα υπάρξει λοιπόν μια σημαντική προσπάθεια στην COP16 ε, να αντιμετωπίσουμε αυτές τις αυξητικέ τάσει λαθροθυρία των απειλούμενων ειδών. Υπάρχουν όμω και άλλα ζητήματα που βρίσκονται στην ημερήσια διαταξή, ιδίω για κάποια θαλάσσια είδη, είδη καρχαριών, τα οποία καλό θα ήταν να περάσουν από τον έλεγχο της σύμβασης και κάποιων ειδών για είδη, είδη ξυλίας όπου θα μπορούσε να λάβει δράση η σύμβαση και να δούμε τι γίνεται με του διεθνού οργανισμού που προστατεύουν ε, κάποια είδη δέντρων. Για τα καρχαρίε τώρα, κάποια είδη καρχαριών, ε, για το διαβολόψαρο και για ε, κάποια είδη δέντρων θα μπορούσαμε να λάβουμε νέα μέτρα σε ό,τι αφορά την, τα θαλάσσια είδη. ο ορισμός της εισαγωγής από τη θάλασσα, όπως λέγεται, θα πρέπει να περατωθεί πλέον ώστε να εξασφαλίσουμε την προστασία κάποιων ειδών καρχαριών, τα οποία αυτή τη στιγμή ψαρεύονται στα ανοιχτά. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν σε αυτή την κόπα αν θα μπορέσουμε πραγματικά να υλοποιήσουμε πραγματική προστασία θαλάσσιων ειδών και ιδίω κάποιων καρχαριών. Θα πρέπει επίσης να δούμε το όργανο ε, για την προστασία του περιβάλλοντος, ένα ταμείο για το περιβάλλον, το οποίο ε, για την ώρα δεν καλύπτει την site Δεν μπορούν τα μέρη, τα συμβαλόμενα μέρη στην site να ζητήσουν ε, προσφυγή στο ταμείο αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να διευκολυνθεί η πρόσβαση στα μέρη της ε, site και να διευκολύνονται τα μέλη στην υλοποίηση τη σύμβασης. Επίσης θα πρέπει να δούμε κάποια θέματα σχέσεων συνεργασία, να ξαναδούμε την όλη μα στρατηγική και να δούμε και ποιοι είναι οι στόχοι της ε, σύμβαση για τη Βιοπικιλότητα και πώς μπορούμε και αυτού να τους ε, υλοποιήσουμε. Επίση μεγάλη έμφαση θα δοθεί στο, διεθνές, στο διεθνή όμιλο για την καταπολέμηση του οικολογικού εγκλήματο. Θα δούμε πώ μπορούμε να συνεργαστούμε με όσου αντιμετωπίζουν την αργονομανή εγκληματικότητα, την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, τι τελωνιακέ απάτε και γενικότερα όλες τις οργανωμένες εγκληματικές ομάδες που εμπλέκονται στη διακίνηση προστατευόμενων ειδών. Πρόεδρε, είναι πολλές οι προτάσεις για νέα είδη που θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην ε, σύμβαση. Πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά το πλαίσιο εντός του οποίου λειτουργεί η σύμβαση. Και βεβαίως πρέπει να θυμόμαστε τις αρνητικές τάσεις αύξησης της λαθροθυρία και παράνομου εμπορίου για κάποια είδη που έχουν συμβολική αξία για την ε, διεθνή κοινότητα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Σκάνλον. Τρεις με 14 Μαρτίου θα γίνει η συνάντηση στο, στην Μπανκόγκ. Πολλά πρέπει να γίνουν μέχρι τότε και το Συμβούλιο θα θέσει ένα ερώτημα προς το Συμβούλιο και στην Κομισία και θα προετοιμάσει και ένα ψήφισμα και η συνχορηγή θα λάβουν το λόγο. Ο Ρίχαρτ Ζέιμπερ θα πάρει το λόγο που εκπροσωπεί τη συνάδελφο κυρία Έστερ Λάγκε. Ε, δυστυχώς η κυρία Λάγκε ε, δεν είναι, μπορεί να είναι παρούσα σήμερα και μιλώ εκ μέρους της. Ευχαριστώ για τις προσπάσεις και το Γενικό Γραμματέα διότι όλοι ξέρουμε, άμα δούμε τα αριθμητικά στοιχεία, αναγνωρίζουμε ότι πάρα πολλά είδη κινδυνεύουν και έχουμε μια μεγάλη ανάγκη προστασίας αυτών των ειδών. Γι' αυτό ε, αυτή η διάσκεψη του χρόνου θα πρέπει να καταλήξει σε συγκεκριμένα συμπεράσματα και όχι μόνο σε υποσχέσεις συμπεράσματα τα οποία θα μπορούν να ε, υλοποιηθούν. Πρέπει ακριβώς να πούμε ποια κράτη θα πρέπει να περιληφθούν σε αυτό τον κατάλογο και αυτός ο κατάλογος να είναι δημόσιος ε, για να μην μας κατηγορήσουν ότι διεξάγουμε μυστικές ψηφοφορίες όλη η διαδικασία να είναι διαφανής και δημόσια. Ε, θα πρέπει να κάνουμε έναν κατάλογο ξεκάθαρο έτσι ώστε να ονομάζονται και να ντροπιάζονται τα κράτη εκείνα τα οποία δεν ενεργούν σωστά ή παραβιάζουν τις ε, διατάξεις. Γι' αυτό θα πρέπει ακριβώς να έχουμε και τις αναγκαίες πιστώσεις για να μπορέσουμε να εκτελέσουμε το έργο μας Παραδείγματο χάρη την εκτέλεση του προγράμματος Monitoring ε, the Killing of Elephants, ε, εποπτεία παρακολούθηση της φαγής των ελεφάντων, και θα πρέπει επίσης ε, να περάσει, να αντισταθούμε, να μην δεχθούμε την μεταφορά του θέματος αυτού από το προσάρτημα 1 στο προσάρτημα 2 και είναι πολύ σημαντικό να υιοθετήσουμε κοινούς ε, κανόνες για την προστασία των θαλασσίων ειδών, των καρχαριών, των ψαριών κλπ. Διότι όπως ξέρουμε η ζωή προήλθε από το, τους και γι' αυτό χρειάζεται το υψηλότερο επίπεδο προστασίας και ο Γενικός Γραμματέας θα προσπαθήσει να μεταδώσει το νήνυμα στα κράτη-μέλη ότι χρειάζεται η ύψιστη προστασία για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τα ίδια αυτά και για τις μέλους γενιές και για τα παιδιά μας. Ευχαριστώ κύριε Ζήμπερ για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες η κυρία Κράμπαχ. Ευχαριστώ και εγώ θερμά όλους τους ε, χορηγούς, τους συνεργάτες θα ήθελα να συμπληρώσω και εγώ τις απόψεις της Έστερ. Ε, πρέπει να πω ότι αντιμετωπίσαμε μεγάλες πιέσεις από τα λόμπι και το ψήφισμα αυτό έχει και μεταφραστικά προσκόμματα δεδομένου ότι στο πλαίσιο των τροπολογιών θα υπάρξουν πολλές προσθήκες και αλλαγές. Έχουμε προθεσμία μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου για να υποβληθούν όλα αυτά ώστε να μπορέσει να γίνει και το μεταφραστικό έργο έτσι, που χρειάζεται το ψήφισμα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Πρόεδρε για την ε, εισαγωγή σας. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε για την επεξεργασία του ψηφίσματός μας. Και Κυρίως να ευχαριστήσω τη Γιάννη για την ε, μεγάλη της συνεισφορά στο ψήφισμα που έχουμε μπροστά μας. Δεν θα επαναλάβω όσα είπε ο κύριος Κάνλον και κάποιοι από τους συναδέλφους. Είναι πολύ σημαντική η συνάντηση της ΚΟΠ στην Πανκόκ του χρόνου, ιδίω για κάποια είδη ξυλίας και κάποια θαλάσσια είδη. Για σκοπούς διαφάνειας επίσης, το κύριο Σέμπερ ανέφερε ότι όλα αυτά θα είναι ζωτική σημασία. Θέλω να αναφέρω όμω και κάτι ακόμη συγκεκριμένα. Ότι το, λαθρεμπόριο, το αυξάνεται παγκοσμίω. Αναφέρθηκαν οι Ρινόκερ από τον κύριο Σκάνλον. Από τους 15 το 2007 περάσαμε σε εκατοντάδες πλέον είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα πλέον. Θα λέγαμε ότι στο παρελθόν στο λαθρεμπόριο υπήρχαν ε, ε, κάποιοι μεμονωμένοι κυνηγοί και τώρα μιλάμε για οργανωμένες ομάδες. Διεθνές εμπόριο. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε με διεθνώς οργανωμένο έγκλημα, με ε, μια αγορά που παγκοσμίως έχει εισόδημα 10 δις ε, δολάρια, με εντυπωσίασε μια ομιλία πριν από τρεις εβδομάδες της Χίλαρη Κλίντον ε, που δεν προήλθε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος η ομιλία αυτή αλλά από την ίδια τη Χίλαρη Κλίντον η οποία μίλησε με μεγάλο, ε, με μεγάλο πάθος για την ε, λαθροθυρία στο διεθνές προσκήνιο και για τους αντικτύπους της. Για πολλές περιοχές του κόσμου είναι θέμα ασφάλειας, είναι θέμα υγείας. Το πρόβλημα ξεπερνάει το θέμα της ε, εξάλληψης κάποιων ε, ειδών ζώων. Είναι λοιπόν κέρια σημασία και η Ευρώπη να εντείνει τις προσπάθειές της. Και δεν είναι μόνο ευθύνη του Επιτρόπου Ποτότσνικ να καταπολεμήσει το διεθνές έγκλημα, τι οργανωμένες ομάδες, αλλά και άλλοι όπως η Βαρόνι Άστον. Να κάνουν ό,τι μπορούν για να το καταπολεμήσουν ως φαινόμενο. Μετά τους επένους για τη Χίλαρη Κλίντον, θα έπρεπε βέβαια να πω και κάποια στοιχεία επικριτικά για τις Ηνωμένες Πολιτείες διότι μετά την εμπορία ειδών ε, που έχουν να κάνουν με τα άγρια ζώα, ε, είπε η Χιλερ Κλίντον ότι είναι ένα από τα θέματα που μετά την ε, διακίνηση ναρκωτικών και την διακίνηση όπλων είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα. Βέβαια, το, τα κέρδη των 15 δις δολαρίων σε σχέση με τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια που δίνει η διακίνηση άλλων ειδών Σίγουρα είναι πολύ, μικρό, πολύ μικρότερες οι διαστάσεις του φαινομένου. Οι Ηνωμένε Πολιτείε λοιπόν, αλλά και η Ευρώπη, θα πρέπει να δώσουν κονδύλια εκεί που υπάρχει το πραγματικό πρόβλημα. Διότι στόχος δεν είναι να καταπολεμηθεί μόνο το διεθνώς οργανωμένο έγκλημα, αλλά και να προσπαθήσουμε να πείσουμε την Κίνα ιδιαιτέρως και τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, να αντιμετωπίσουν τη ζήτηση κεράτων ρινοκέρου ή άλλων ειδών που μπορεί να προέρχονται από τίγρης και ούτω καθεξής. Το πρόβλημα είναι ότι κάποιοι γίνονται πλουσιότεροι ή αισθάνονται ότι γίνονται πλουσιότεροι. Ε, είναι δείγμα στάτους, ε, ένδειξη στάτους για, κάποιες, ε, για τις μέσες τάξεις κάποιων χωρών το να έχουν κάποια τρόπαια από ρινόκερο ή από άλλα αγριαζόα. Θα ήθελα λοιπόν ο κύριο Κάνλον να μου πει εάν θα μπορούσε ο ΣΑΙΤΕΣ κάτι να κάνει και γι' αυτό. Την πρόληψη, δηλαδή που ίσως να είναι και σημαντικότερη από την πραγματική καταπολέμηση των ε, εγκληματιών εδώ. Και η Ιντερπολ διδραματίζει σημαντικό ρόλο, αλλά η σχετική τους ε, δυνατότητα είναι πολύ περιορισμένη. Πριν από ένα ή δύο χρόνια νομίζω ότι μίλησα με τον μόνο επιφορτισμένο να ασχολείται με την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματο αυτού του τύπου στην Νοτιοανατολική Ασία. Σω ο κύριος Κάνιλα να έχει περισσότερε πληροφορίε σχετικά. Αλλά εδώ το προσωπικό που διατίθεται είναι ένα τεράστιο πρόβλημα σχετικά. Και το ερώτημά μου προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι τι σχεδιάζει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώ θα εντείνει τι προσπάθειέ τη κατά των εγκλημάτων, ε, κατά των αγρίων ζώων. Η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, ή άλλες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπουν κάτι, μπορούμε να συνεργαστούμε με τις ΗΠΑ για να αντιμετωπίσουμε αυτό το μεγάλο φαινόμενο και να δώσουμε σοβαρά κίνητρα ώστε να, το να λάβουμε δραστικά μέτρα. Ευχαριστώ. Ε, τώρα για τους πράσινους. Ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Σκάνλοντ, λέει ο κύριος Έλκουτ. Λυπάμαι που άργησα λιγάκι, αλλά είμαι βέβαιος ότι κάνετε μια θαυμάσια εισαγωγή, εισήγηση για την σημασία του ΣΑΙΤΕΣ ε, και το Κοινοβούλιο έχει παίξει ένα σημαντικό ρόλο εκφράζοντας τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή ότι πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι, πιο δυναμικοί στη διεθνή σκηνή. Δεν θα επαναλάβω αυτά τα οποία είπαν ή προλαλήσαντε συνάδελφοι διότι πιστεύω ότι σε αυτό το κοινοβούλιο υπάρχει μία ε, συνεργασία μεταξύ των ομάδων, των πολιτικών ομάδων και πιστεύω ότι η διάσκεψη της Μπαγκόκ θα, είναι, θα έχει φιλόδοξους στόχους. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη θα παίξει το ρόλο που της αρμόζει στη Μπαγκόκ. Αυτή είναι και ερώτησή μου προς την Κομισιόν. Θα ε, έχουμε προετοιμαστεί καιρός αυτή τη φορά για να εξασφαλίσουμε ότι όταν υπάρχει διαφανής διαδικασία ψηφοφορίας, όταν θα υπάρχει λοιπόν ψηφοφορία, θα έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμάχους στην ε, προηγούμενη COP ε, του ΣΑΙΤΗΣ ήμουνα στην Τόχα και ήταν πολύ απογοητευτικό να διαπιστώνουμε ότι η Ευρώπη οθούσε και πίεζε για πρόοδο στην προστασία της κλωρίδας, της πανίδας κλπ. Αλλά όλες τις προτάσεις μας τις χάσαμε. Γιατί χάσαμε σχεδόν σε όλα, διότι όλες οι άλλες χώρες του κόσμου ήταν καλύτερα προετοιμασμένες. Ξέρουμε βεβαίως ότι η Ευρώπη ε, έχει μεγάλες δυσκολίες να καταλήξει σε κοινή θέση για τον τόνο για τον βόρειο τόνο με γαλάζια αλλά το θέμα είναι ότι όταν οι διαπραγματευτές της Κομισιόν πήγαν στην Τόχα την ημέρα που άρχιζε η διάσκεψη τότε μπόρεσαν να ενημερωθούν ε, δηλαδή ήταν κατά κάποιο τρόπο ε, δυσάρεστο να δεις αυτό το γεγονός της καθυστέρησης και βεβαίως λόγω της ανεπαρκούς προετοιμασίας απέτυχαν τώρα γιατί δεν, μπόρεσαν, ε, δεν μπόρεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταλήξει σε μια κοινή θέση. Δεν ξέρω. Οι άλλες χώρες μπόρεσαν να ενερμονίσουν τη θέση τους παραδείγματος χάρη και να ακολουθήσουν τη γραμμή της Κίνας. Εμείς δεν μπορέσαμε. Και όταν φτάσαμε εμείς στην Τόχα ψηφίσαμε με το σωστό τρόπο, έτσι όπως θα έπρεπε δηλαδή, αλλά οι άλλες χώρες δεν ψήφισαν έτσι. Λοιπόν, αυτή τη φορά να ρωτιέμαι, θα είμαστε προετοιμασμένοι, θα έχουμε συμμάχους που θα υποστηρίξουν τη θέση μας, πέραν δηλαδή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι το ερώτημά μου σήμερα και είμαι πολύ περίεργο να μάθω από την Κομισιόν τι, τι στρατηγική θα ακολουθήσει. Έχει βελτιώσει τη στρατηγική της, έχει μάθει από, τα, το προηγούμενο πάσημα της ε, Ντόχα. Αυτή είναι η βασική μου ερώτηση. Για όλα τα υπόλοιπα, βεβαίω θα προσπαθήσουμε να υποβάλουμε τροπολογίε που να αναφέρονται σε πιο συγκεκριμένα είδη στο ψήφισμα, αλλά πρέπει να πω ότι γενικά εμείς στο Κοινοβούλιο έχουμε μια καλή προσέγγιση και έτσι θα καταλήξουμε σε καλό ψήφισμα. Το πρόβλημα δεν είναι το ψήφισμα, το πρόβλημα είναι εάν μπορέσουμε το ψήφισμα αυτό να το περάσουμε, να τύχουμε υποστήριξη περισσότερων κρατών από τα κράτη-μέλη μα. Ο Πρόεδρος. Βεβαίω, το ψήφισμα πολλέ φορές είναι η θεωρία, η ψηφοφορία είναι η πρακτική υλοποίηση, πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε να μεταφέρουμε στην πρακτική εφαρμογή τη θεωρία μας. Ο κύριος Πίτερ Φοντάν είναι ο επόμενος ομιλητής. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Πραγματικά τα προβλήματα αυτά είναι πολύ σημαντικά και θα πρέπει να καταπολεμήσουμε. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ όλο αυτό το ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με την λαθροθυρία, ιδίως όσον αφορά τους ελέφαντες. Το πρόβλημα είναι ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό προσπαθούμε να εξαλείψουμε το φαινόμενο αυτό, αλλά χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Στις αρχές του έτους είχα πάει στην Νότιο Αφρική και είδα ότι υπάρχουν εκεί κάποιες ε, ομάδες ελεφάντων που πραγματικά προστατεύονται. Δεν γίνεται όμως το ίδιο για τους ρινόκερους, για τους οποίους η λαθροθυρία συνεχίζεται πάρα πολύ έντονα. Και βλέπουμε ότι πολλές φορές οι επιτόπου φύλακες δεν μπορούν να κάνουν σπουδαία πράγματα. Τι μπορεί λοιπόν να γίνει στο μέλλον. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να επικεντρωθούμε πραγματικά στους στόχους μας. Πολύ συχνά συντάσσουμε γενικόλογια ψηφίσματα με πάρα πολλά σημεία θεωρώ ότι το δικό μας το ψήφισμα θα πρέπει να επικεντρωθεί αυτή τη φορά σε ένα ή δύο συγκεκριμένα σημεία. Δηλαδή, να επικεντρωθούμε στο ζήτημα της ε, λαθροθυρίας, στο ζήτημα της διακίνησης των ε, κεράτων ε, ρινοκέρων και είναι πάρα πολύ σημαντικό το 2003 να αποτελέσει το έτος αυτό κατά το οποίο θα αναλάβουμε πραγματική πολιτική δράση και αν δούμε τα πράγματα από πολιτική πλευρά, θα πρέπει να μα απασχολήσει επίση και η χρηματοδότηση των προγραμμάτων που θέλουμε να προωθήσουμε. Θα δούμε επίση αν θα έχουμε κάποιου πολιτικού συμμάχου στον αγώνα μα αυτό. Αναφερθήκατε στι Ηνωμένε Πολιτείε. Θα πρέπει όμω να γνωρίζετε ότι πολύ συχνά μα δίνονται γενικόλογε αόριστες υποσχέσει από τι Ηνωμένε Πολιτείε. Δίνονται επίση ε, κάποιες ε, χρηματοδοτήσεις οι οποίες όμως τελικά δεν ε, καταλήγουν σε συγκεκριμένα προγράμματα και συγκεκριμένες πράξεις. Πρέπει να γίνουμε πολύ πιο συγκεκριμένοι αυτή τη φορά, προκειμένου πραγματικά να διεξάγουμε ένα σημαντικό αγώνα το 2013. Και μια ερώτηση να θέσω προς το Γενικό Γραμματέα. Μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν θετικές επιπτώσεις από τον αγώνα αυτό, από τη μάχη αυτή, κατά της λαθροθυρίας και της θανάτωσης ή του ακροτηριασμού πολλές φορές των ειδών αυτών Υπάρχει πραγματικά μία ελπίδα, διαφαίνεται κάπου μία ελπίδα για το μέλλον. Δεν νομίζω, είμαι κάπως απεσιόδοξο ενδεχομένω. Thank ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ με το ψήφισμα αυτό. Όντως το πρόβλημα της λαθροθυρίας ε, παρουσιάζει όλο και μεγαλύτερη ανάπτυξη και επίσης πρέπει να μας απασχολήσει και το ζήτημα της αποκοπής των πτερυγίων των καρχαριών, ζήτημα το οποίο έχουμε ήδη αντιμετωπίσει στις σχέσεις που έχουμε με τους Κινέζους. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένα σημείο το οποίο απουσιάζει από το ψήφισμα. Ένα ζήτημα ασφαλείας. Σε ορισμένε περιπτώσεις εγκληματίες ή τρομοκράτες έχουν φύγει πλέον από την Αφρική και σκοτώνουν ελέφαντες σε άλλες περιοχές και προσπαθούν να χρηματοδοτήσουν κατά αυτόν τον τρόπο τις α, δραστηριότητές τους. Υπάρχουν ακόμα και περιοχές ή χώρες που έχουν πάρα πολλούς φύλακες, αλλά τελικά δεν καταφέρνουν να ανταποκριθούν στο γεγονός ότι υπάρχουν πλέον ολόκληρες παραστρατιωτικές οργανώσεις, οι οποίες προχωρούν σε δραστηριότητες ε, λαθροθυρίας. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να επικεντρωθούμε και στο ζήτημα αυτό. Να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή την τελευταία διαθέσιμη τεχνολογία προκειμένου να βοηθήσουμε τους ε, φύλακες οι οποίοι επιτόπου προσπαθούν να καταπολεμήσουν το φαινόμενο της λαθροθυρίας. Και επίσης προσπαθούν να βοηθήσουν και να σώσουν τις ζωές των ανθρώπων που καταπολεμούν τα φαινόμενα. Ευχαριστώ κύριε Σούτερ. Και ε, δίνω το λόγο τώρα στον εκπρόσωπο της Επιτροπής, την Κομισιόν. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον που δείχνετε για την site της. Πράγματι, ΣΥΤΕΣ είναι μια πάρα πολύ σημαντική σύμβαση και ένα διασνές μέσο προστασίας ε, ειδών αλλά και προώθησης ε, βιώσιμου εμπορίου. Είναι πολύ σωστό να λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υποστηρίξει σερμά αυτή τη σύμβαση και πρέπει να συνεχίσουμε την υποστήριξη διότι έχουμε μεγάλη κρίση να αντιμετωπίσουμε ιδίως στη λαθροθυρία. Η Κομισιόν, όπως ξέρετε, αυτή τη στιγμή προετοιμάζει μια απόφαση του Συμβουλίου και πρόσφατα ξεκινήσαμε την εσωτερική διαβούλευση για αυτή την απόφαση του Συμβουλίου η οποία στο τέλος θα καθορίζει την στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ΚΟΠ είναι νωρίς ε, να μιλήσουμε για αυτή την πρόταση. Μόλις ξεκίνησε η εσωτερική διαδικασία και είναι υπό διαβούλευση. Αλλά θα ήθελα να τονίσω δύο στοιχεία τα οποία έχουμε ενσωματώσει σε αυτό το σχέδιο απόφασης. Ε, το πρώτο είναι ότι θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι η σύμβαση θα χρησιμοποιηθεί πλήρως για την προστασία των θαλασσίων ειδών. Ήδη έχετε αναφέρει τους καρχαρίες πιστεύουμε ότι αυτή είναι μια σημαντική ευκαιρία να τονίσουμε το πρόβλημα αυτών των ειδών, συγκεκριμένων ειδών και θα πρέπει επίσης να συνεργαστούμε με τις λατινοαμερικές χώρες δεδομένου ότι ε, έχουμε επιτύχει κάποια πρόοδο πριν από, σχετικά με το τι υπήρχε πριν από μερικά χρόνια, ιδίως στους φυροκέφαλους καρχαρίες. Το δεύτερο στοιχείο που θέλουμε είναι να εδραιώσουμε μια μεγαλύτερη διαφάνεια. Ήδη ακούσαμε τις μυστικές ψηφοφορίες που γίνονται και πιστεύουμε ότι είναι δυσανάλογη, δυσανάλογο το φαινόμενο αυτό που συμβαίνει στους κόλπους της ΣΑΙΤΙΣ και πιστεύουμε ότι δεν είναι σωστό να υπάρχουν αυτές οι μυστικές ψηφοφορίες και θα πρέπει τουλάχιστον να, να προβάλλουμε προσκόμματα ως προς αυτό το φαινόμενο. Ε, ε, έχουμε μια υποστήριξη και από την πλευρά του Μεξικού παραδείγματο χάρη, αν και δεν είναι τόσο φιλόδοξοι ως εμείς. Το επόμενο θέμα είναι να αποφύγουμε τη σύγκρουση συμφερόντων στις επιτροπές του ΣΑΙΤΙΣ. Αυτή τη στιγμή ε, δεν υπάρχει καμία διαδικασία η οποία να ε, αμβλύνει, να μπορεί να ξεπεράσει τη σύγκρουση συμφερόντων. Και τέλος, η τρίτη προτεραιότητα είναι υλοποίηση και εφαρμογή. Ε, εκεί έχουμε μεγάλα, μεγάλες ελλείψεις, τις ανέφερε ο κύριος Σκάνλον και άλλοι. Το βασικό πρόβλημα στην ε, εφαρμογή και υλοποίηση και να το πω λίγο απλά τα πράγματα, ε, άσπρο σε μαύρο δηλαδή, ε, δεν θα μπορέσουμε, αν δεν έχουμε σωστούς καταλόγους, να υλοποιήσουμε τα μέτρα που αφορούν συγκεκριμένα είδη. Ελπίζω λοιπόν η ΚΟΠ στην Ταϊλάνδη να τονίσει ιδιαίτερα το θέμα της ε, εφαρμογής, της υλοποίησης. μας ε, ε, τέσει το ερώτημα τι κάνουμε για την, ε, τα εγκλήματα κατά της άγριας πανίδας. Έχουμε 2 εκατομμύρια ευρώ, υπολογίσει 2 εκατομμύρια ευρώ για την καταπολέμηση αυτού του εγκληματικού φαινομένου και μπορώ να σας ανακοινώσω με μεγάλη ικανοποίηση, δεν είναι μόνο ο, Πύρο, ο κύριος Ποτόσκι ή ο Γενικός Διευθυντής ε, Περιβάλλοντος, αλλά είναι και οι συνάδελφοι από την Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης που είναι και οι ταμείες που έχουν τα χρήματα, ότι μας υποστηρίζουν σε αυτή τη χρηματοδότηση. Εν συνεχεία ο κύριος Σέρκαρτ ρώτησε τι κάνουμε ή ε, εάν, προσπα... εάν προσπαθούμε να συμπεριφερθούμε πιο έξυπνα ή πιο οργανωμένα για να ε, μας υποστηρίξουν και άλλοι. Όπως σας είπα υπάρχουν και άλλες χώρες οι οποίες ε, έχουν προτάσεις που θα υποβάλουν τις οποίες μπορούμε να υποστηρίξουμε. Παραδείγματος χάρη Καρχαρίες έχουμε μία σύμπνοια απόψεων, δεδομένου ότι είναι ένα θέμα που παγκόσμιο ενδιαφέροντος και σίγουρα θα αναπτύξουμε περαιτέρω αυτή τη σύμπνοια και με τα άλλα κράτη-μέλη θα αναπτύξουμε μία συνεργασία προς τρίτους η οποία θα είναι πιο συντονισμένη και πιο οργανωμένη οι Ηνωμένε Πολιτείε που συνήθως είναι στο πλευρό μας ε, όταν συζητούμε τα θέματα του ΣΑΙΤΙΣ, όχι τόσο στο περιβάλλον, αλλά τουλάχιστον στα θέματα της ΣΑΙΤΙΣ έχουμε μια υποστήριξη από εκεί. Θα έρθουμε σε επαφή και με άλλους ε, ενδιαφερόμενους, με άλλους παίκτες στη διεθνή σκηνή, με τους οποίους έχουμε τα ίδια ενδιαφέροντα, ίδιες έννοιες και απόψεις. Ε, ε, έχουμε λοιπόν δραστηριοποιηθεί όσο μπορούμε περισσότερο για να συνεργαστούμε με άλλους εταίρους. Αυτά είχα να πω, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας. Και τέλος δίνω το λόγο στο Γενικό Γραμματέα για να απαντήσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ όλους σας για την υποστήριξη που δίνετε στην ε, σύμβαση COP16 της ΣΑΙΤΙΣ. Ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η ΣΑΙΤΙΣ, γιατί χωρίς αυτήν το διεθνές εμπόριο δεν θα ρυθμιζόταν στα άγρια είδη. Θα μπορούσε να γίνει ένα οποιοδήποτε εμπόριο ανάμεσα σε οποιαδήποτε χώρα, χωρίς να υπάρχει καμία υποβολή αναφοράς. Ακριβώς επειδή έχουμε τη ΣΑΙΤΙΣ, έχουμε και ένα ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο υποχρεώνει τα κράτη να υποβάλουν αναφορές σε σχέση με τα ίδια αυτά τα οποία καλύπτονται από την site της. Κατά αυτόν τον τρόπο το εμπόριο είναι βιώσιμο. Χωρίς τη site ουσιαστικά δεν θα υπήρχε κανένας απολύτως έλεγχος. Η πρόταση της Τανζανίας για την πώληση του ελεφαντόδοντου, το οποίο θα εξετάσουμε στην Κόπ τον επόμενο Μάρτιο, ουσιαστικά βρίσκεται εκτός οποιοδήποτε πλαισίου προτείνει να πουλήσει οποιαδήποτε ποσότητα ελεφαντόδοντου σε οποιαδήποτε χώρα χωρίς κανέναν έλεγχο. Αυτό το πλαίσιο ελέγχου, αυτό το ρυθμιστικό πλαίσιο θέλουμε να δημιουργήσουμε και να επιβάλλουμε σε όλες αυτές τις χώρες οι οποίες συμμετέχουν στην ΣΑΕΤΙΣ. Έχουμε πει ότι για συγκεκριμένα απειλούμενα είδη θέλουμε να υπάρχει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο ελέγχου. Για συγκεκριμένα είδη τα οποία βρίσκονται στα προσαρτήματα 2 και 3 δεν θέλουμε να υπάρχει καθόλου εμπόριο, να είναι περιορισμένο ρυθμισμένο το εμπόριο. Στην συνδιάσκεψη Ρίο η οποία έλαβε χώρα πρόσφατα, αναγνωρίστηκε η σημασία της ΣΑΙΤΙΣ ως σύμβαση η οποία βρίσκεται πραγματικά στο σταυροδρόμι ανάμεσα στην ανάπτυξη, το περιβάλλον και πραγματικά τονίστηκαν οι επιπτώσεις που μπορεί να έχει τόσο στην οικονομία όσο και στο περιβάλλον. Επίσης, ε, με τη site ασχολείται και η ε, Υπουργό Εξωτερικών Χίλαρη Κλίντον. όλε οι Ηνωμένε Πολιτείε, στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο ασχολούνται με την site της, ιδίως για την εφαρμογή της ε, στην Αφρική. Στο... Υπάρχουν ομάδε ανθρώπων που έρχονται από το Σουδάν στο βόρειο Καμερούν, σκοτώνουν ελέφαντε, παίρνουν το ελεφαντόδοτο και το πουλάνε στη συνέχεια προκειμένου να αγοράσουν όπλα για τι τοπικέ διενέξει, του τοπικού πολέμου βλέπουμε ότι σε πέντε χώρες της Αφρικής υπάρχουν πλέον ομάδες, ακόμα και στο Καμερούν, που θέλουν να προστατεύσουν την άγρια πανίδα. Δεν μπορούν όμως οι άνθρωποι αυτοί να αντιμετωπίσουν τις παραστρο... αυτές οργανώσεις. Είναι εξοπλισμένες, έχουν όπλα σκοτώνουν τους ελέφαντες και οι τοπικοί φύλακες δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Πρέπει λοιπόν να καταφέρουμε να ασχοληθούμε με την Τσάιτης όχι μόνο σε περιβαλλοντικό αλλά και σε πολιτικό πλέον επίπεδο. Δεν μπορούμε μόνο μέσω των Υπουργών Περιβάλλοντος να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό. Θα πρέπει να έχουμε και τη συνεργασία του στρατού, της αστυνομίας, των τελωνιακών αρχών. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι άπτονται πλέον πολύ διαφορετικοί τομείς. Η Υπουργό Εξωτερικών λοιπόν Κλίντον μίλησε πολύ ένθερμα για την Σάιτις και ο επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ αναφέρθηκε επίσης στη σημασία της ΆΙΤΙΣ και στο πώς μπορεί να συμβάλλει για την προστασία των ειδών πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται. Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχουν πάρα πολλέ επιπτώσει μέσω τη που οι οποίε θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σε πολιτικό επίπεδο και να δούμε επίση τι μπορεί να γίνει σε τοπικό επίπεδο. Το γεγονό ότι πολλέ φορέ έχουμε και φαινόμενα διαφθορά κάποιων τοπικών πολιτικών σε χώρε όπου προσπαθούν να προστατεύσουμε κάποια είδη. Στι 15 Νοεμβρίου διάβασα μια επιστολή που πήγε στην Επιτροπή Ασφαλεία των ΗΠΑ όσον αφορά τα όσα γίνονται στη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό. Χρησιμοποιείται εκεί το ελεφαντόδοτο προκειμένου να αγοραστούν όπλα. Επομένως τίθεται ένα ζήτημα ασφαλείας για την ίδια τη χώρα αυτή. Υπάρχει ένα εμπόριο σε ορυκτά και το εμπόριο τώρα αυτό έχει απλωθεί ακόμα και στο ελεφαντόδοτο. Τι κάνουμε προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση αυτή. Δημιουργήσαμε ένα consortium καταρχάς, αναγνωρίσαμε ουσιαστικά ότι υπάρχει μία απειλή από εξοπλισμένες οργανωμένες εγκληματικές ομάδες, από παραστρωτικές οργανώσεις και είπαμε ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση αυτή. Δημιουργήσαμε λοιπόν ένα consortium, αναφέρθηκε σε αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ουσιαστικά έχουμε την Interpol, την αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ, την γραμματεία της ITIS και τη βοήθεια επίσης της Παγκόσμιας Τράπεζας και προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε τις μυστικές μας πληροφορίες καθώς επίσης και τη βάση δεδομένων και τις δυνατότητες ε, δημιουργίας ικανοτήτων που έχουμε προκειμένου να καταφέρουμε να εμπλέξουμε αστυνομικές τελωνιακές δυνάμεις με το ζήτημα αυτό της προστασίας δηλαδή των ειδών χλωρίδας και Πανίδα. Βλέπουμε ότι εμπλέκονται όλο και περισσότεροι τομεί. Υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται από τη Σουηδική κυβέρνηση, ονομάζεται Gapen, που ουσιαστικά εκπαιδεύονται τελωνιακοί για να καταφέρουν να αντιμετωπίσουν αυτές τις ε, εγκληματικέ ε, ε, δραστηριότητες λαθροθυρίας. Το ίδιο γίνεται και σε άλλες οργανώσεις, όπως για παράδειγμα στην Interpol. Στις Ηνωμένε Πολιτείες επίσης Έχω έρθει σε επαφή με τον ε, επικεφαλής ε, αντιμετώπισης πώλησης διακίνησης ναρκωτικών, ο οποίος ε, θέλει και αυτός να συνεργαστεί στα πλαίσια της ΣΑΙΤΙΣ. Βλέπουμε λοιπόν ότι Ομάδε οι οποίε ασχολούνταν στο παρελθόν μόνο με τη διακίνηση παράνομων αγαθών, αυτή τη στιγμή ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για την παράνομη λαθροθυρία. Και βλέπουμε ότι αυτό γίνεται στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο. Είτε πρόκειται για τον τομέα τη πολιτική, είτε πρόκειται για τον τομέα τη δικαιοσύνη, είτε τον τελωνιακό φορολογικό τομέα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί η δραστηριότητα αυτή, μα λένε όλοι αυτοί οι θύνοντε, πρέπει να σταματήσει αυτό το φαινόμενο. Αν είμαι αισιόδοξο, ναι, έχω κάποιε ελπίδε. Θεωρώ ότι η κατάσταση αυτή τη στιγμή δεν είναι βιώσιμη. Θα πρέπει να σταματήσουν όλα αυτά τα φαινόμενα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια αυξητική τάση όσον αφορά την ε, λαθροθυρία, κυρίω του ελέφαντε και του ε, ρινόκερου. Αν δεν σταματήσουμε τα φαινόμενα αυτά, θα οδηγηθούμε ουσιαστικά στην εξαφάνιση αυτών των ειδών και θα εξαφανιστούν σε ορισμένε περιοχέ Αφρική ακόμα και οι τοπικοί πληθυσμοί. Πολλά πράγματα πρέπει να γίνουν επίση και για την εφαρμογή των νομοθεσιών, για την επιβολή των νομοθεσιών. Έχουμε επίσης απειλούμενα είδη, όπως για παράδειγμα οι τίγρεις, οι οποίες είναι πλέον 3.000 μόνο. Έχουμε συγκεκριμένα είδη ρινοκαίρονα στην Ινδονησία, για παράδειγμα, που απειλούνται πάρα πολύ έχουμε μόνο 780, 780 γορίλες των βουνών, έχουν μείνει πάρα πολύ λίγοι ουσιαστικά. Πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα για να αναχαιτήσουμε την τάση αυτή και θα πρέπει να αλλάξει η κοινοτροπία τελικά των ανθρώπων. Όσον αφορά τους ε, ρινόκερους, είχαμε μια κάποια επιτυχία. Υπάρχει ένα παραδοσιακό κινέζικο φάρμακο το οποίο χρησιμοποιούσε κέρατα από ρινόκερο, το οποίο έχει σταματήσει πλέον να χρησιμοποιείται. οι θεραπείες αυτές οι οποίες χρησιμοποιούντουσαν στο παρελθόν έχουν σταματήσει, από την άλλη έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούνται όμως τμήματα του ρινόκυρου αυτή τη στιγμή ως αφροδυσιακά και πρέπει να σταματήσει βέβαια και η τάση αυτή. Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να απευθυνθούμε στις χώρες στις οποίες βρίσκονται περισσότερες καταναλωτές, οι περισσότεροι καταναλωτές των ειδών αυτών. Πρέπει να καταφέρουμε να μειώσουμε τη ζήτηση στα προϊόντα αυτά. Θα πετυχεί βέβαια χρόνος και θα πρέπει να καταβάλουμε τι απαραίτητε προσπάθειε προκειμένου να μειωθεί η ζήτηση. Έχουν μείνει όμω τόσα λίγα ήδη πολλέ φορέ, απειλούνται τόσο πολύ που πραγματικά πρέπει να προχωρήσουμε πάρα πολύ γρήγορα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ε, χρηματοδότησή τη στα προγράμματα παρακολούθηση λαθροθυρία των ε, ε, ελεφάντων. Πραγματικά είχαμε την καλύτερη παρακολούθηση που υπήρξε ποτέ για οποιοδήποτε είδο. Και πραγματικά η πρακτική τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί ένα παράδειγμα προ μίμηση για το μέλλον. Έχουμε πλέον τα απαραίτητα δεδομένα, έχουμε τι απαραίτητε αναλύσει και θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τι μεθόδου αυτέ και για άλλα είδη. Να ευχαριστήσω λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για όλη την υποστήριξή τη. Όντω τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν, υπάρχει ελπίδα, αλλά θα πρέπει να υπάρχει συνεχή χρηματοδότηση, εμπλοκή του πολιτικού τομέα σε ανώτατο επίπεδο. Χωρί χρηματοδότηση δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Θα πρέπει να διατηρηθεί η γραμματεία, θα πρέπει να καταφέρουμε να εμπλέξουμε περισσότερους ανθρώπους και φορεί στα πλαίσια τη σάιτης και να έχουμε υποστήριξη στο υψηλότερο δυνατό πολιτικό επίπεδο. όσον αφορά την εισαγωγή από τη θάλασσα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να επιληθεί το ζήτημα αυτό. Ζήτημα το οποίο συνδέεται με τις προτάσεις που έχουν γίνει για την καταχώρηση συγκεκριμένων θαλασσίων ειδών, κυρίως για τους καρχαρίες. Αλληλοσυνδέονται τα ζητήματα αυτά, καρχαρίες και εισαγωγή από τη θάλασσα και είναι πάρα πολύ σημαντικό να συζητηθούν στην COP16 και να επιληθούν αυτά και άλλα εκρεμή ζητήματα. Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι απάντησα στις ερωτήσεις που μου απευθύνθηκαν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε ένα από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υποστήριξη που μας έχουν δώσει. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σκάνλον, για τις απαντήσεις σας και πρέπει να πω ότι οι συνάδελφοι που λείπουν σήμερα έχασαν πραγματικά. Και οι συνάδελφοι που είναι παρόντες κέρδισαν και πληροφορήθηκαν ότι έχουν ακόμα να κάνουν πολλή δουλειά για να προετοιμαστούμε όλοι για τη διάσκεψη του Μαρτίου. Είναι πολύ σημαντικό για όλους να διατηρηθούν ε, εν ζωή τα 35.000 ε, είδη και πρέπει να πείσουμε και τα άλλα κράτη που μας ανταγωνίζονται. Γι' αυτό είμαι βέβαιος και αισιόδοξο και με την υποστήριξη της Κομισιόν ότι θα μπορέσουμε να έχουμε μια σωστή τεκμηρίωση για τα στοιχεία που αφορούν τους ελέφαντες και τα άλλα είδη. Χωρίς τη σωστή τεκμηρίωση δεν μπορούμε να πείσουμε τους ε, άλλους συμμετέχοντες οι οποίοι δεν έχουν ακόμα διαμορφώσει μια συγκεκριμένη άποψη μας ε, θυμήσατε βεβαίως ξανά ότι έχουμε ένα νομικό πλαίσιο, ένα νομοθετικό πλαίσιο. Εμείς δεν θέλουμε την μετα... τη μεταφορά από το παράρτημα 1 στο παράρτημα 2 και αυτή είναι μία από τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε στην COP16. Για τους συναδέλφους λέω ότι Παρασκευή 13 Νοεμβρίου είναι η προθεσμία την υποβολή τροπολογιών. Εδώ στην Επιτροπή Περιβάλλοντος θα ψηφίσουμε τις 23-24 Ιανουαρίου και το Φεβρουάριο του χρόνου θα υπάρχει το ψήφισμα στην ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας Εγκαίρως λοιπόν διαμορφώσαμε το χρονοδιάγραμμα για να είμαστε έτοιμοι για το Μάρτιο. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Έμαθα πολλά και, διαπιστώσαμε ότι είσαστε απολύτως δεσμευμένος στην επίτευξη των στόχων μας. Ευχαριστώ πολύ για την επίσκεψή σας. Wir kommen jetzt zum και προχωρούμε στο σημείο της ημερήσιας διάταξης 5 και 6 για την ανακύκλωση των πλοίων. Και το σημείο 6 ε, είναι περισσότερο νομοθετικό και προτείνω να τα συζητήσουμε μαζί τα δύο θέματα δίνω καταρχά το λόγο στην Επιτροπή, στην Κομισιόν. Εν συνεχεία θα μιλήσει ο εισηγητής και θα παρουσιάσει και ένα βίντεο τριών λεπτών για να έχουμε μια πρώτη αντίληψη πώς γίνεται όλη αυτή η διαδικασία της διάλυσης στην πραγματικότητα. Εγώ προέρχομαι από μια παράκτια περιοχή, αλλά όσοι δεν ζουν κοντά σε ακτές μπορεί ίσως να μην έχουν μια εικόνα ε, στο μυαλό τους για την όλη διαδικασία. Δίνω λοιπόν το λόγο στην Κομισιόν. Good morning, Mr. Chair, honorable members. Thank you very Καλημέρα, αξιότιμα μέλη. Ευχαριστώ που δίνετε καταρχάς το λόγο στην Κομισιόν για να παρουσιάσω αυτή τη σημαντική πρόταση. Και είναι σημαντική διότι σήμερα περίπου χίλια μεγάλα πλοία διαλύονται κάθε χρόνο ε, παγκοσμίω και τα μέταλλα ανακυκλώνονται ως πολύτιμες πρώτες ύλες. Η διάλυση αυτή γίνεται συνήθως σε μακρινές περιοχές στην Νότια Ανατολική Ασία κάτω από απαράδεκτες, απάνθρωπες και λίαν επικίνδυνες συνθήκες διότι τα περισσότερε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επειδή τα περισσότερα πλοία δεν έχουν τη σημαία των νέων κρατών μελών, Πρέπει να βρούμε μια διεθνή λύση για αυτό το πρόβλημα και ε, αυτή η λύση μπορεί να βρεθεί μόνο σε διεθνέ επίπεδα. Γι' αυτό ακριβώ η επικύρωση τη σύμβαση του Χονγκ Κόνγκ για την ανακύκλωση των πλοίων είναι σημαντική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως πρέπει να αποτελέσει το παράδειγμα και γι' αυτό η Κομισιόν έχει προτείνει ένα νέο κανονισμό για την ανακύκλωση των πλοίων και πιστεύουμε ότι πρέπει να τεθεί ενισχύει το συντομότερο. Επίσης η Κομισιόν έχει προτείνει ένα σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που θα ζητήσουν από όλα τα κράτη-μέλη να επικυρώσουν τη σύμβαση του Χονγκ Κόνγκ το ταχύτερον. Η Κομισιόν θέλει να εξασφαλίσει ότι στην κοινοτική νομοθεσία, στην ενωσιακή νομοθεσία, τα πλοία τα οποία έχουν σημαία νέου κράτους μέλους θα διαλύονται με τις κατάλληλες ε, συνθήκες υπό συνεχή εποπτεία και τεκμηρίωση. Τα βασικά στοιχεία της ε, πρότασης της Κομισιόν στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο είναι πρώτον ότι τα τα πλοία τα οποία θα έχουν τη σημαία νέου κράτους μέλους θα είναι υποχρεωμένα να διατηρούν έναν κατάλογο των επικινδύνων ουσιών που έχουν. Δεύτερον, τα πλοία αυτά θα πρέπει να ανακυκλώνται μόνο υπό ασφαλείς και περιβαλλοντικά φιλικές συνθήκες έτσι όπως βάσει ενός καταλόγου εγκαταστάσεων που θα έχει η Κομισιόν. Για να υπάρχει αυτό, για να δημιουργηθούν αυτές οι συνθήκες, θα καθιερώσουμε ένα καθεστώς αυστηρών ε, ποινών και κυρώσεων. Οι εγκαταστάσει διάλυσης μπορεί να είναι οπουδήποτε στον κόσμο βάσει των διατάξεων της Σύμβασης του Χονγκ Κόνγκ. Όμως θα πρέπει να είναι πιστοποιημένες και θα πρέπει να, να πιστοποιείται ε, ότι λειτουργούν υποσφαλίσεις και υγιείς υγιεινές συνθήκες. Αυτή τη στιγμή η τα πλοία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ε, μπορούν να σταλούν σε ε, χώρες που δεν ανήκουν στον ΟΣΑ. Αυτή είναι η μετάφραση της απαγόρευσης εξόδου επικίνδυνων αποβλήτων υπό την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Όμως, αυτή η απαγόρευση εξαγωγής ε, επικινδύνων αποβλήτων δεν έχει μπορέσει να εφαρμοστεί σωστά. Πρέπει εμείς να εξασφαλίσουμε ότι όλα τα πλοία τα οποία έχουν αυτές τις σημαίες ε, διαλύονται με ασφαλή τρόπο και ελεγχόμενο βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει την εποπτεία και τον έλεγχο και γι' αυτό ακριβώς δημιουργήθηκε και η σύμβαση του Χονγκ Κονγκ. Δυστυχώς όμως δεν έχει ακόμα τεθεί ενισχύ και θα χρειαστεί κάποιος χρόνος μέχρι ότου τεθεί ενισχύ. Ο στόχος της πρότασης της Κομισιόν είναι να ε, προωθήσει την ταχεία επικύρωση αυτής της σύμβασης. Έχουμε χώρες οι οποίες ήδη εφαρμόζουν την σύμβαση της Hong Kong. Όμως η επικύρωση θα οδηγήσει ε, στην ενδυνάμωση των ε, κατάλληλων συνθήκων για τη σωστή διάλυση των πλοίων. Αυτή η πρόταση έχει ως στόχο να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα όχι μόνο στην Ένωση Εφοπλιστών αλλά και στην όλη βιομηχανία ανακύκλωσης πλοίων όσοι, και να υποστηρίξει όσους ήδη έχουν επενδύσει στη βελτίωση των εγκαταστάσεών των. Έφτασε η ώρα επιτέλους να επενδύσουν ε, στις, ε, στη βελτίωση της εγκατάστασης και των συνθήκων εργασίας εάν θέλουν να συνεχίσουν ε, την διάλυση των πλοίων. Και θα καταλήξω με μία πρόταση, Πρόεδρε. Η Κομισιόν έχει ως στόχο να κάνει την ανακύκλωση, την διάλυση των πλοίων, συγγνώμη, βιώσιμη μέσα σε ένα πλαίσιο ασφάλειας και φιλικό προς το περιβάλλον. Ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε σεμιτές και δίκαιες συνθήκες έτσι ώστε να μην αποστέλλονται τα πλοία στις εγκαταστάσεις στη, για διάλυση στην Νοτιοανατολική Ασία μόνο για, την, για πρόσκαιρο κέρδος και να αποβαίνει όλη οι διαδικασίες βάρος των εργαζομένων και τη υγείας τους. Ο πρόεδρος, πολύ σύντομα ο κύριος Σλούτερ. Για πολλούς το ζήτημα αυτό ενδεχομένω να είναι εντελώς καινούριο. Θα ήθελα να σας πω πραγματικά πώς έχει η κατάσταση και τι προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε. Για το λόγο αυτό θα σας δείξω ένα πολύ μικρό απόσπασμα, ένα φιλμ από το Μπαγκλαντές το 2009, Αντίστοιχε όμω καταστάσει έχουμε δει ακόμα και φέτο. Η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί τα τελευταία δύο χρόνια. Αυτό το οποίο θα δείτε πραγματικά είναι αντιπροσωπευτικό του πώς γίνεται η διάλυση των πλοίων στις χώρες αυτές. Θα δείτε επίσης ε, ότι υπάρχει και ένας εργαζόμενος ο οποίος σχεδόν ε, πλακώνεται από τα τμήματα του πλοίου ενώ δουλεύει για τη διάλυση του πλοίου αυτού. Χρησιμοποιείται ουσιαστικά ο νόμος της βαρύτητας προκειμένου να διαλυθούν αυτά τα πλοία και δεν υπάρχει καμία προστασία για τους εργαζομένους. Θα τη δείτε όλα αυτά στην ε, ταινία, στο φιλμ. Σας ευχαριστούμε πολύ μπορούμε να ξεκινήσουμε το βίντεο. As you can see, the situation is really dark. Θα πρέπει να ξαναρχίσουμε. Γιατί κάναμε ένα δοκιμαστικό χθε και είχε πετύχει. Αλλά αυτή τη φορά δεν είναι τόσο απλό.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 power up the engines and in high tide drive the ship onto the beach. Αυτή είναι η πρακτική της προσάραξης, όπου κατά την, ε, το φούσκωμα της παλήριας οδηγείται στην παραλία το πλοίο. Αμάρ, μπορείτε να δοκτώρ, μπορούν το τσάκι. Αντώντα,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 Βάστι. sing to walk in the same pace everybody because it's Περπατάνε όλοι με τον ίδιο βηματισμό και με τον ίδιο ρυθμό γιατί είναι πολύ βαρύ το φορτίο. Και αν τους πέσει θα πέσει μισός τόνος στα πόδια τους, γι' αυτό προσπαθούν να βαδίζουν ταυτόχρονα. Ευχαριστούμε πολύ. Είδαμε λοιπόν το φιλμ αυτό και θα δώσουμε πάλι στον εισηγητή το λόγο. Ζητάμε, συζητάμε το ζήτημα αυτό γιατί υπάρχει, όπως είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμβαση του Hong Kong. Αυτό το οποίο ισχύει όμως αυτή τη στιγμή είναι η σύμβαση της Βασιλείας, η οποία απαγορεύει όλες τις εξαγωγές επικίνδυνων αποβλήτων. Εδώ και 14 χρόνια ισχύει η σύμβαση της Βασιλείας, ότι όμως υπάρχει η σύμβαση αυτή, ένα 90% των πλοίων που έχουν ευρωπαϊκές εταιρείες διαλύονται τελικά παράνομα, δηλαδή σε χώρες εκτός όσα. Οι πιο σημαντικές χώρες για τη διάλυση είναι τον Μπαγκλαντές όπως είδαμε και στο φιλμ, η Ινδία και το Πακιστάν επίσης. Και στις τρεις αυτές χώρες η κατάσταση είναι πάνω κάτω παρόμοια. Είδατε επίσης στο φιλμ αυτό ότι ε, χρησιμοποιούν διάφορες τεχνικές διάλυσης ε, του πλοίου. Και ξέρετε ότι ε, αν πρέπει να διαλυθεί για παράδειγμα ένα δεξαμενόπλιο, τότε θα πρέπει να προηγηθεί μια διαδικασία καθαρισμού, καθαρισμού του, προκειμένου να μην απομείνουν κάποια έφλεκτα υλικά πάνω στο πλοίο. Αυτό όμως δεν γίνεται, με αποτέλεσμα τα υλικά να υπάρχουν και διάφορα ατυχήματα με πυρκαγιές. Βλέπετε σε ορισμένε περιπτώσει ότι υπάρχουν κάποια πλοία, τμήματα του πλοίου, τα οποία τελικά φλέγονται και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για του εργαζομένου. Γίνεται επίση αυτή η μέθοδο τη προσάραξη όταν υπάρχει το φαινόμενο τη παλήρεια. Όταν υποχωρούν όμω τα νερά, τελικά όλα τα τοξικά απόβλητα, οι τοξικέ ουσίε παραμένουν πάνω στο πλοίο και στη συνέχεια περνάνε στη θάλασσα. Επίση, τα πλοία κανονικά καλύπτονται από τη Σύμβαση της Βασιλείας όσον αφορά τα επικίνδυνα απόβλητα και αυτό γιατί υπάρχουν καύσιμα πάνω στο πλοίο βέβαια, καθώς επίσης και αμίαντος. Όλα επίσης ε, τα πλοία έχουν ε, PVC, πολυβινοχλωρίδιο, καθώς επίσης και άλλα υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται για την προστασία τους από πυρκαγιές. Επίσης ε, υπάρχουν κάποια πολλά τοξικά, πολλές τοξικές χημικές ουσίες που προστατεύουν πάλι το πλοίο από την φθορά. Υπάρχουν γενικά πάρα πολλές επικίνδυνες ουσίες, αμίαντος όπως είπαμε. Σε ορισμένε περιπτώσεις θάβουν τον αμίαντο στην γη και τον καλύπτουν με χώμα. Σε άλλες περιπτώσεις επιστρέφει πάλι στην αγορά και χρησιμοποιείται ως οικοδομικό υλικό σε διάφορες παραγκουπόλεις. Η κατάσταση είναι δραματική, επηρεάζει τη δημόσια υγεία, δεν υπάρχει καμία ασφάλεια και τελικά βλέπουμε ότι πάρα πολύ τοξικές χημικές ουσίες περνάνε στη θάλασσα όταν υποχωρήσει η παλήρια. Για ποιο λόγο όμως τα πράγματα εξελίσσονται κατά αυτόν τον τρόπο. Είδατε ότι ο μισθό των ανθρώπων αυτών είναι 2 δολάρια την ημέρα, και είναι πολύ πιο φτηνό βέβαια η διάλυση των πλοίων να γίνει στις χώρες αυτές, στο Μπαγκλαντές, την Ινδία ή το Πακιστάν. Σε αυτούς τους χώρους διάλυσης, αν μπορούμε να τους πούμε έτσι, στις παραλίες αυτές τελικά καταβάλουν οι εταιρείε αυτές προς τους πλειοκτήτες μεγαλύτερη τιμή ακριβώ επειδή το κόστος εργασίας είναι πάρα πολύ χαμηλό για τις εταιρείε αυτές. Όπως σας είπα, τα τελευταία χρόνια προσπαθούμε να επιβάλλουμε τη σύμβαση της Βασιλείας τα τελευταία 14 χρόνια. Δεν το καταφέρνουμε όμως ακριβώς επειδή το δίκαιο της θάλασσας είναι πάρα πολύ πολύπλοκο. υπάρχουν ε, πάρα πολλοί κανόνες που έχουν να κάνουν με τον πλειοκτήτη, με τον ιδιοκτήτη του πλοίου. Οι κανόνες όμως, αυτοί διαφέρουν από τη μία περιοχή στην άλλη και πάρα πολύ συχνά τροποποιούνται. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι ε, οι ε, πλειοκτήτες ουσιαστικά δεν μπορούν να ε, πουλήσουν τα πλοία τους αν τα πλοία αυτά έχουν φτάσει στο τέλος του κύκλου της ζωής τους και ουσιαστικά θα πρέπει τελικά να διαλυθούν. Ουσιαστικά προσπαθούν να παρακάμψουν τη με νομοθεσία προκειμένου να καταφέρουν να πουλήσουν τα πλοία τους αυτά σε κάποιους χώρους διάλυσης. Είναι πάρα πολύ δύσκολο όμως να αποδείξουμε τα φαινόμενα αυτά. Και μόνο στο 1% των περιπτώσεων καταφέρνουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Αρχίσαμε να συζητάμε τη σύμβαση του Χονγκ Κόνγκ ακριβώ επειδή τα πρότυπα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι απαράδεκτα. Αλλά παρόλα αυτά και η σύμβαση του Χονγκ Κόνγκ δεν απαγορεύει τη μέθοδο τη προσάραξη, απλώ θέτει κάποιε προποθέσει. Η σύμβαση του Χονγκ Κόνγκ θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι έρχεται σε αντίφαση με τη σύμβαση της Βασιλείας γιατί επιτρέπει την εξαγωγή σε χώρες εκτός όσα για τη διάλυση των πλοίων. Κάτι τέτοιο είναι πραγματικά παράδεκτο. Αλλά και η φυστάμενη κατάσταση είναι απαράδεκτη. Αυτό που προσπαθώ λοιπόν να κάνω με την εκθεσή μου είναι να δημιουργήσω ένα καθεστώ το οποίο θα λειτουργεί σωστά. Δηλαδή θα πρέπει τα πλοία αυτά να διαλύονται με ένα σοβαρό και σωστό τρόπο. Επί του παρόντος, οι βασικές χώρες παραγωγής πλοίων είναι η Νότια Κορέα, η Κίνα και η Ιαπωνία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα μόνο 2,5% της συνολικής παραγωγής. Η Ρωμανία 0,6%. Δεν είμαστε λοιπόν πλέον σημαντικές χώρες δημιουργίας πλοίων. Θα πρέπει να απευθυνθούμε κυρίω λοιπόν στι χώρε εκείνε που έχουν τα υψηλά ποσοστά κατασκευή πλοίων, όπω για παράδειγμα η Κίνα, η οποία όμω δεν ανήκει στον ΩΣΑ. Η σύμβαση λοιπόν του Hong Kong νομιμοποιεί τη μέθοδο, αυτό, τη μέθοδο αυτή και Μολονότι έχουμε τη σύμβαση της Βασιλείας, όπως σας είπα υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να παρακάμψει κανείς την υφιστάμενη νομοθεσία. Προσπαθήσαμε λοιπόν να επιβάλλουμε ένα πρόστιμο στους ε, πλειοκτήτες, στους τελευταίους πλειοκτήτες ενός ε, πλοίου, όταν αυτοί προσπαθούν να πουλήσουν το πλοίο τους για διάλυση. Εγώ θεώρησα ότι θα πρέπει να προβλέπεται μια χρονική περίοδος δύο ετών και να μην έχει να κάνει μόνο με τον ε, τελευταίο, αλλά πολλές φορές και με τον πρώτο τελευταίο διοκτήτη του πλοίου. Τα πρόστιμα όμως και οι κυρώσεις δεν πρόκειται τελικά να μας βοηθήσουν. Αν δεν συμμορφωθούν οι πλειοκτήτες και ο τομέας της ναυτιλίας με τη Σύμβαση της Βασιλείας δεν πρόκειται να συμμορφωθούν ούτε με τη Σύμβαση του Χονγκ Κονγκ. Αυτό το οποίο προτείνω λοιπόν είναι αυτό το οποίο είπε και ο κύριο Μπλόκλαντ στα δύο προηγούμενα ψηφίσματα τα οποία ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και στι δύο περιπτώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε πει ότι μπορούμε να, θα μπορέσει να λειτουργήσει το σύστημα μόνο αν δημιουργηθεί ένα ταμείο. Δηλαδή, να υπάρχει μία πρημοδότηση για τους ε, φορείς εκείνους οι οποίοι θα λειτουργούν με τρόπο νόμιμο. Ακριβώς αυτό μπορεί να γίνει και με τα πλοία, πιστεύουμε. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δώσουμε τα απαραίτητα κίνητρα προκειμένου η διάλυση του πλοίου να γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ουσιαστικά το ταμείο αυτό θα καλύπτει την διαφορά η οποία προκύπτει από το να πουλήσει ο πλειοκτήτης το πλοίο σε έναν χώρο διάλυσης ο οποίος ακολουθεί συγκεκριμένα πρότυπα. Μπορεί ο πλειοκτήτης να μην κερδίσει πάρα πολλά χρήματα αλλά τουλάχιστον η διαφορά αυτή θα καλυφθεί από το τομείο αυτό το οποίο θέλουμε να δημιουργήσουμε. Η χρηματοδότηση του ταμείου αυτού θα γίνεται με την, με την προσάραξη των πλοίων κάθε φορά που πηγαίνουν σε ένα λιμάνι. Κάθε φορά που πλοία προσαράζουν σε κοινοτικό λιμένα θα πρέπει να πληρώνουν ένα μικρό τέλος, το οποίο μπορεί να είναι 0,03 ευρώ ανατόνο, και κατά αυτόν τον τρόπο μπορεί να χρηματοδοτηθεί το ταμείο αυτό. Δεν ξέρω αν θα καταλήξουμε τελικά στο ποσό αυτό, μπορούμε να το συζητήσουμε. Πιστεύω ότι θα πρέπει να καλύψουμε τουλάχιστον το 10% της διαφθοράς, της διαφοράς με συγχωρείτε, η οποία προκύπτει ανάμεσα στο να διαλύσει κανείς ένα πλοίο σε νόμιμο χώρο διάλυσης και στην τιμή η οποία θα μπορούσε να κερδίσει αν διέλυε το πλοίο του σε έναν παράνομο χώρο διάλυσης. Πιστεύω λοιπόν ότι ε, η καταβολή του τέλους αυτού θα χρηματοδοτήσει το ταμείο αυτό, προκειμένου τελικά να μπορεί να λειτουργήσει. Το κόστος ε, για τον τομέα της ναυτιλίας δεν θα είναι υψηλό, γιατί τα χρήματα από το ταμείο αυτό τελικά θα επιστρέψουν στον τομέα της ναυτιλίας κάθε φορά που τα ε, πλοία θα διαλύονται με σωστό τρόπο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να καταφέρουμε να έχουμε και έναν κατάλογο, έναν ευρωπαϊκό κατάλογο χώρων διάλυσης που θα ακολουθούν συγκεκριμένα πρότυπα τα οποία θα εξασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρχουν χημικές ουσίες οι οποίες θα περνάνε στα θάλασσες, στα νερά του ωκεανού μετά την διάλυση του πλοίου και ότι θα υπάρχει και απαραίτητη υποδομή προκειμένου να γίνεται κάτι τέτοιο. Αν συμμορφώνεται λοιπόν κανείς με τα κριτήρια αυτά, τότε θα μπορεί να χαίρει και τις χρηματοδότηση, η οποία θα προβλέπεται. Σύμφωνα με τη σύμβαση πρέπει να καλύψουμε τα πλοία εκείνα τα οποία φέρουν ευρωπαϊκή σημαία. Αν όμως αρχίσει να λειτουργεί το σύστημα αυτό, τότε θα καταφέρουμε πραγματικά να βελτιώσουμε την κατάσταση. Σήμερα ένα ίμιση των πλοίων που φέρουν ευρωπαϊκή σημαία χάνουν αυτή την ευρωπαϊκή σημαία, ουσιαστικά αλλάζουν σημαία λίγο πριν τη διάλυση, ακριβώς για να παρακάμψουν την φυστάμενη νομοθεσία αν καταφέρουμε να δημιουργήσουμε το νέο αυτό σύστημα, θα καταφέρουμε να καταργήσουμε την πρακτική αυτή. Θα δώσουμε και ένα κίνητρο προκειμένου ο πλειοκτήτης να διατηρήσει την ευρωπαϊκή σημαία μέχρι το τέλος του κύκλου ζωής του πλοίου. Ακριβώς επειδή θα καταφέρει να χρηματοδοτηθεί σωστή διαλυσή του από το ταμείο το οποίο θέλουμε να δημιουργήσουμε. Πιστεύω ότι η πρόταση αυτή μπορεί να λειτουργήσει στην πράξη. Έχει πολύ χαμηλά ποσοστά γραφειοκρατίας και θεωρώ ότι ε, η εναλλακτική τελικά του να διατηρήσουμε το φυστάμενο σύστημα είναι κάτι το απαράδεκτο, γιατί έχουμε μόνο παράνομες δραστηριότητες τελικά. Παραβιάζουμε τη σύμβαση της ε, Βασιλείας και δεν μπορώ καν να δεχθώ το επιχείρημα της ανταγωνιστικότητας. Δεν μπορούμε να μιλάμε για την ανταγωνιστικότητα μέσω της παραβίασης νομοθεσίας. Θεωρώ λοιπόν ότι θα καταβάλουμε μέσω της πρότασής μου ένα ελάχιστο κόστο προκειμένου τελικά να καταφέρουμε να εφαρμόσουμε τη σύμβαση της Βασιλείας και στο μέλλον τη σύμβαση του Χονγκ Κονγκ και θα καταφέρουμε κατά αυτόν τον τρόπο με ασφάλεια να διαλύουμε τα πλοία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρθηκε επίση σε έναν κατάλογο και αυτή η ιδέα είναι πολύ θετική. Εγώ επέφερα τουλάχιστον κάποιε θετικέ τροποποίησει στην ιδέα αυτή και είπα ότι θα πρέπει να αναφερθούμε και συγκεκριμένε χημικές ουσίες οι οποίες βρίσκονται πάνω στα πλοία και όπως σας είπα ένα 20% του παγκόσμιου στόλου προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ πάντως ότι θα καταφέρουμε να έχουμε την απαραίτητη χρηματοδότηση προκειμένου να προωθήσουμε την σωστή ασφαλή διάλυση των πλοίων. Πιστεύω ότι με τη δημιουργία του Ταμείου αυτού η κατάσταση στο μέλλον θα είναι πάρα πολύ καλύτερη. Και πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να βοηθήσουμε και τις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να προχωρούν στις ίδιες θετικές πρακτικές. Ο αντίκτυπος λοιπόν της πρότασης θα είναι παγκόσμιος τελικά. Τώρα, διερωτάστε ενδεχομένω για ποιο λόγο έκανα μία πρόταση για τον κανονισμό αυτό και όχι για την σύμβαση αυτή καθ' αυτή. Θεωρώ ότι η αποδοχή της σύμβασης και η προσχώρηση σύμβαση θα πρέπει να συνδεθεί με τον κανονισμό. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να έχουμε μια σύμβαση του Χονγκ Κόνγκ η οποία στην πράξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μην εφαρμόζεται. Όπω ακριβώ έχουμε δει και με τη σύμβαση τη Βασιλεία. Στην περίπτωση αυτή α διατηρήσουμε τη σύμβαση τη Βασιλεία και α προσπαθήσουμε να τη βελτιώσουμε. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να προχωρήσουμε πρώτα με έναν ευρωπαϊκό κανονισμό και συνέχεια να δούμε πώς θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την σύμβαση του Χονγκ Κονγκ. Ευχαριστώ με τον κύριο Σλούτερ. Και τώρα δίνουμε στην Κρίστα το λόγο. Ε, θα δώσουμε στην Κρίστα το λόγο στον κύριο Φιέλνερ πρώτα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λίτερ παρουσίασε πολύ εύλογα το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Είναι απαράδεκτη κατάσταση. Η διάλυση παλιών πλοίων ή τέλος πάντων ο σωστός όρος που χρησιμοποιείται είναι ανακύκλωση. Η ταινία, δεν ξέρω ποιον όρο έπρεπε να χρησιμοποιήσει, ποιος είναι ο δόκιμος, αλλά ακούσαμε και την παρουσίαση της Επιτροπής. Μας είπε ότι υπάρχουν ε, τρόποι να επιδιώξουμε μια σωστή υλοποίηση διεθνών υποχρεώσεων μέσω της σύμβασης του Χονγκ Κονγκ. Ο κ. Χίλτερ προτείνει πέντε διαφορετικές λύσεις. Πρώτα απ' όλα θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για έναν φόρο για τα πλοία. Ένα δασμό Κάτι τέτοιο νομίζω ότι περιγράψατε. Έπειτα υπάρχει ο κατάλογος των χώρων διάλυσης, η ανακύκλωση και το σχέδιο ανακύκλωσης και τέλος τα πρόστιμα για τις διάφορες παραβιάσεις. Σε ό,τι αφορά τον κατάλογο και τις απαιτήσεις για, τις, ε, για τους χώρους διάλυσης, τις εγκαταστάσεις διάλυσης, νομίζω έχει δίκιο ο εισηγητής. Όμως, ο δασμός ή φόρος ή όπως αλλιώς τον ονομάσουμε για τα πλοία είναι κάτι που μου προκαλεί ερωτηματικά. Εάν επιβάλλουμε τέτοιο φόρο σε όλα τα πλοία που προσαράζουν ή αγκυροβολούν ε, στην Ευρώπη ασχέτως της σημαίας που φέρουν και συλλέξουμε όλα αυτά τα ποσά, αυτό θα είναι μια ένα πρώτο βήμα. Όμως θα επιδοτούμε τα ευρωπαϊκά πλοία. Έπειτα, μπορεί να υπάρξει μαζική αποχώρηση και αλλαγή σημεών σε αυτή την περίπτωση. Οι Ηνωμένε Πολιτείε τι ε, θα μπορούσαν να κάνουν παρομοίω. Να πούν ότι θα φορολογήσουμε τα ευρωπαϊκά πλοία και να χρησιμοποιήσουμε τα έσοδα ω ε, ε, χρηματοδότηση για να επιδοτήσουμε αμερικάνικα σκάφη. Θα αλλάξει τελείω το σύστημα νεολόγηση των πλοίων τα ευρωπαϊκά σκάφη θα περάσουν σε Αμερικανούς ε, πλειοκτήτες. Αυτό δεν το θέλουμε φαντάζομαι. Επιπλέον το πρόβλημα με αυτό το είδος των φόρο ή δασμό ή τη δημιουργία ενός μεγάλου ευρωπαϊκού ταμείου είναι κάτι που έχει να κάνει γενικότερα με το σχέδιο ε, ανακύκλωσης με τα σχέδια ανακύκλωσης, τα οποία θα μπορούσαν και να λειτουργήσουν, αλλά θα υπάρχει και μια γραφειοκρατική διαδικασία και τα έπαχθες. Όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να τα εγκρίνουν, να τα ε, καταρτήσουν από κοινού και μετά να υπάρχει και μια κοινή διαχείριση. Για αυτού τους λόγους, Καλ, ε, θα έλεγα ότι το πρώτο σημείο είναι λίγο προβληματικό. το υπόλοιπα να τα συζητήσω και να γίνει Ευχαριστώ ο κύριος Μπρόντι. Μπρόντι. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για, ε, για το έργο του στο θέμα αυτό. Βεβαίως, η πρόταση αυτή προκαλεί σύγχυση για τους διάφορους ενδιαφερομένους. Είναι κάπως παράξενο να βλέπουμε μη κυβερνητικέ οργανώσεις από τη μια να παραπονούνται για την κακή υλοποίηση της σύμβασης και από την άλλη οι εφοπλιστές να είναι ικανοποιημένοι. Ας δούμε τα πράγματα μας από την αρχή. Εξ όσων κατάλαβα, η αιτιολόγηση για αυτόν τον νέο κανονισμό είναι η ελλειπής ε, υλοποίηση της σύμβασης της Βασιλείας και της, ε, του κανονισμού για την ανακύκλωση. Εγώ πρώτος θα παραδεχτώ ότι τα ε, εργαλεία αυτά, τα μέσα, τα νομοθετικά δεν είναι αρκετά για να αντιμετωπιστεί η προσάραξη των πλοίων. Υπάρχουν σοβαρές ε, πιέσεις που ασκούνται έτσι στις ε, χώρες του τρίτου κόσμου. Όμω, οι ευγενεί αρχέ που μα οδήγησαν να αγωνιστούμε για την ε, σύμβαση τη Βασιλεία και τι αρχέ τη τώρα μπορεί να είναι τόσο πραγματιστικέ ώστε να μα οδηγήσουν να αναγνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει κανονισμό ή σύμβαση που να, μας μπορεί, που να μπορεί να μα επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε περιβαλλοντικές καταστροφές και παραβίαση ανθρώπινων δικαιωμάτων που προκαλούνται από τη διαχείριση των ευρωπαϊκών σκάφων. Είναι δυνατόν και μπορεί να παραδεχτεί κανείς ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί θα ε, αναγνωρίζουν ότι δεν γίνονται σεβαστοί οι ίδιοι οι δικοί τους κανόνες. Στη χώρα μας ο Πρωθυπουργό ήταν τόσο ρεαλιστής ώστε να δέχεται ότι πολλοί Ε, ανοίγουν λογαριασμού στο εξωτερικό προκειμένου να μπορούν να μετακυλίουν ε, τη φορολόγηση στα τραπεζικά τους. Εδώ λοιπόν, ε, Πρόεδρε, θα πρέπει την αρχή αυτή να την ε, σκεφτούμε, εάν μπορεί να εφαρμοστεί στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και εάν τα πράγματα συνεχιστούν προς αυτή την κατεύθυνση, θα έχουμε νομικό ασύμβατο και κενό που θα μας οδηγήσει σε ένα χάος και για τις ευρωπαϊκές και για τις αναδυόμενες οικονομίες, εάν επανεληφθεί η περίπτωση της σύμβασης της Βασιλείας. Και εδώ μην ξεχνάμε ότι έχουμε στην ε, Ευρώπη ναυπηγεία. Αυτοί απευθύνουν μια έκκληση για βοήθεια προς το μέρος μας. Θα πρέπει λοιπόν στους όλους κανόνες για το τέλος ζωής των σκαφών να λάβουμε υπόψη και τη συνιστόσα της τεχνολογίας, τις τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά και τις περιβαλλοντικές ανάγκες. Τα στοιχεία αυτά καθορίζουν ένα υψηλότερο πολιτιστικό επίπεδο και θα πρέπει να μας οδηγήσουν σε υψηλότερες περιβαλλοντικέ απαιτήσει. Εγώ ανησυχώ για το εξή. Πώς θα μπορούσαμε να τονώσουμε την ευρωπαϊκή και μεσογειακή ναυτιλία, τα ναυπηγεία σε τέτοιου καιρού κρίσης προωθώντα ταυτόχρονα την υγιή και φιλική προ το περιβάλλον ανακύκλωση των πλοίων. Ο εισηγητή έχει προτείνει τη δημιουργία ενό ταμείου για να παροτρύνουμε συγκεκριμένα είδη συμπεριφορά μεταξύ πλειοκτητών και εφοπλιστών στην Ευρώπη. Εγώ νομίζω ότι οι Ευρωπαίοι θα περάσουν στα κινέζικα ναυπηγεία, χωρί να ασχοληθούν με την προστασία του περιβάλλοντο. Οι κινέζικε ενώσει και συλλογοί έχουν παραδεχτεί ότι ναι, έχουν τη δυνατότητα να ναυπηγήσουν σκάφη για μα, αλλά δεν μπορούν να ασχοληθούν με το θέμα των επικίνδυνων ουσιών, όπως τα PVC και ούτω καθεξής. Θα πρέπει λοιπόν να μην ε, περάσουμε σαν μπαλάκι το πρόβλημα σε εκείνους. Θα πρέπει να αναζητήσουμε μια άλλη λύση ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν τω μεταξύ, θα πρέπει να αναλυφθούν πρωτοβουλίε ε, και κυρίω να απευθυνθούμε στην νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου για να δούμε κατά πόσο είναι συμβατή η σύμβαση τη Βασιλεία με την προτινόμενη σύμβαση του Χονγκ Κόνγκ. Ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι υπάρχει νομικό κενό. Θα μπορούσε να προκύψει τέτοιο κενό εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρήσει ότι ισχύει η σύμβαση της Βασιλείας και η σύμβαση του Χονγκ Κόνγκ ε, είναι ανοιχτή μόνο για συγκεκριμενα κάτι κράτη-μέλη, δηλαδή με περιορισμένο αριθμό συμβαλωμένων. Αυτά όλα θα χρειαστούν χρόνια για να ισχύσουν το σελος Τι θα κάνουμε στο μεταξύ. Οι εγκληματίες του εργατικού χώρου συνεχίζουν να εγκληματούν. Ξέρουμε ότι κάποια κράτη χρειάζονται ευρωπαϊκό έλεγχο προκειμένου να περιοριστεί αυτό το είδους το έγκλημα στα εργασιακά και προκειμένου να εξασφαλίσουμε τη σωστή υλοποίηση των συμβάσεων. Φοβούμε λοιπόν ότι η κατάσταση απλώς θα επιδεινωθεί εντωμεταξύ. μεταξύ. Κατά κύριο λόγο πρέπει να βρούμε μέτρα που να υποχρεώνουν τα ευρωπαϊκά σκάφη να διαλύονται σε ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις ώστε να προστατεύεται το περιβάλλον, τους, να προστατεύουμε τους εργαζομένους μας και να μπορέσει να ανακάμψει και η οικονομία του όλου τομέα. Νομίζω λοιπόν ότι όλα αυτά θα πρέπει να τα σκεφτούμε σοβαρά. Θεωρώ ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλες λύσεις. I Εγώ νομίζω ότι ο κύριος Σλάιτερ μας ε, έκανε μια θαυμάσια ε, χειρονομία βάζοντας το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη για να συζητήσουμε ακριβώς τις χείριστες πρακτικές ε, και τους κινδύνους της διάλυσης πλοίων. Και ο στόχος μας είναι βεβαίως να ενισχύσουμε την ε, διάλυση των πλοίων σε, στην ευρωπαϊκή επικράτεια. Όμως ε, όλες αυτές οι συμβάσεις και οι συμφωνίες αυτή τη στιγμή έχουν τόσα πολλά κενά, τόσα πολλά παρασυράκια που δεν προσφέρουν και πολλά. Προσφέρουν πολύ λίγα. Εγώ μου αρέσουν οι ιδέες τις οποίες προέβαλε ο Καρλ. Βεβαίως βλέπω και τις αντιρρήσεις, ε, κόστος, δαπάνες, δεν είναι ο κατάλληλος χρόνος αυτός. Όμως το, οι ιδέες οι οποίες ε, μας εξέσεσε οδηγούν στην ε, ελαχιστοποίηση του κόστους. Ε, μπορούμε να επιτύχουμε ελαχιστοποίηση του κόστους χωρίς να βασιζόμαστε στις χείριστες μεθόδους, την πολύ κακή μέθοδο διάλυσης των πλήρων. Μπορούμε και να βελτιώσουμε τη διάλυση αλλά και να μειώσουμε, να συγκρατήσουμε το κόστος. Εγώ θα έλεγα προς το Συμβούλιο, εάν δεν μπορέσετε να υποστηρίξετε αυτές τις προτάσεις, ελπίζω να μπορέσουν, μπορείτε εσεί στο Συμβούλιο να μας παρουσιάσετε εναλλακτικέ λύσεις, να μας πείτε τι καλύτερο μπορείτε να κάνετε ώστε να κλείσουμε τα παρασυράκια που υπάρχουν. Δεν νομίζω να μπορέσουν να βρούνε τέτοιες εναλλακτικέ λύσεις και γι' αυτό ακριβώς προσβλέπουμε προς την Κομισιόν η οποία μας παρουσίασε όχι μόνο τη δική της θέση αλλά ανταποκρίνεται και στις ιδέες, δηλαδή θέλουμε να δούμε αν ανταποκρίνεται στι ιδέε του Καρλ, ο Πίτερ Βαντάλερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή διότι μπορέσαμε πραγματικά να κάνουμε μια πολύ καλή ανταλλαγή ε, απόψεων για αυτές τις μεθόδους ε, διάλυσης και χαίρομαι ιδιαίτερα που προέβαλε αυτή την ιδέα και ο Hans Blockland είχε ήδη παρουσιάσει αυτό το θέμα. Είχαμε κάνει και ένα ψήφισμα για το, την έκθεση Blockland. Όπως σωστά είπε ο κ. Σλούτερ, δεν είναι δυνατόν να κινδυνεύει η ζωή των ανθρώπων ε, για, τη διάλυση, όταν εκτελούν αυτή τη διάλυση πλοίων υπό απαράδεκτες συνθήκες. Τα, τον, πέρσι, τα τελευταία χρόνια, καμία αλλαγή δεν έγινε και ακόμα ε, διαλύονται πλοία εκτός χωρών ΩΣΑ. 90% των πλοίων υπό, υπό ευρωπαϊκών κρατών διαλύονται έτσι. Και η σύμβαση της Βασιλείας παραμένει μία σύμβαση επιχάρτου και τίποτα περισσότερο. Ε, τι θα γίνει τώρα το 2020, θέλουμε να εδρώσουμε ένα ε, νέο σύστημα και ελπίζουμε να λειτουργήσει καλά, αλλά δεν το ξέρουμε. Ελπίζω, Πρόεδρε, να καταλαβαίνουν όλοι ότι η παρούσα κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν μπορούμε να, έχουμε, να κάνουμε ασκήσεις επί χάρτου και να μην έχουν καμία ουσιαστική σημασία αυτές οι συμβάσεις. Πρέπει να ασχοληθούμε σοβαρά με τη με τις μεθόδους διάλυσης. Ποια είναι λοιπόν η βασική προσέγγιση. Καταρχάς θα πρέπει να κλείσουμε τα παρασυράκια και τα διάφορα κενά της ελλείψης που υπάρχουν, δεδομένου ότι η πρόθεση είναι να γίνει με το φτηνότερο τρόπο η διάλυση στο Μπαγκλαντές. Υπάρχει λοιπόν μια τεράστια, ένα τεράστιο χάσμα μεταξύ του κόστου στην Νοτιοανατολική Ασία ε, και στα ευρωπαϊκά, στις ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν αν υπάρχουν δυνατότητες να γίνουν οι διαλύσεις αυτές στην ευρωπαϊκή επικράτεια. Ε, μήπως ε, πρέπει να επιβάλλουμε ε, κάποια εισφορά μαζί με την, τις εισφορές για τους λιμένες που ήδη ισχύει, μπορούμε να αποφύγουμε ενδεχομένω γραφειοκρατικά εμπόδια κλπ. Λοιπόν υπάρχουν διάφοροι τρόποι που μέσω της υπάρχουσας διαδικασίας να μπορέσουμε να επιβάλλουμε μια ισφορά, μια ειδική εισφορά. Δεν μπορούμε απλώς να απορρίπτουμε κάτι χωρίς να προτείνουμε μια εναλλακτική λύση. Οι δύο αυτές συμβάσεις του Χοκόν και της Βασιλείας αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα, έχουν όση αξία όσο και το μελάνι με το οποίο έχουν γραφτεί. Λοιπόν, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε αυτή την κατάσταση. Και τι, γίνεται τώρα με τα ε, πλοία τα οποία παραμένουν σε ευρωπαϊκούς λιμένες αλλά δεν έχουν ευρωπαϊκή σημαία και απλώς τα εγκαταλείπουν. Ε, το πλήρωμα δεν μπορεί να πληρωθεί πλέον, ε, το εγκαταλείπουν το πλοίο και τα πλοία αυτά παραμένουν αραγμένα στα ευρωπαϊκά λιμάνια. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο αυξάνεται και έχει ξεκινήσει εδώ και 10 χρόνια, ε, παραδείγματο χάρη στο Άμστερνταμ υπάρχουν πλοία τα οποία έχουν εγκαταληφθεί στο λιμάνι του Άμστερνταμ ε, πολλά χρόνια και τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πιστώσεις, παραδείγματο χάρη που εισπράττονται από τις εισφορές που καταβάλλονται στους, στα λιμάνια. και δεν αφορά μόνο πλοία με σημαία τρίτων χωρών και ευρωπαϊκά, ευρω, σημαίες ευρωπαϊκών κρατών ε, διαπιστώνουμε ότι εγκαταλείπουν τα πλοία αυτά. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε το, το θέμα αυτό συνολικά και να δούμε εάν μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο ταμείο και όχι να το απορρίπτουμε εξ αρχής λέγοντας ότι είναι πολύ δύσκολο, αδύνατο να γίνει κλπ. Εάν συνάδελφοι ε, ε, ειδικοί απορρίπτουν τις λύσεις που προτείνουμε, τότε θέλω να ακούσω από το στόμα τους τι λύσεις προτείνουν αυτοί. Και τέλος για το σχέδιο της Κομισιόν, για την διατήρηση του άρθρου 23 και την συμπλήρωση του άρθρου αυτού με πολλές άλλες λεπτομέρειες για τη λεπτομερή διαχείριση του προβλήματος και την επιβολή κυρώσεων και ποινών. Το, το βρίσκω υπερβολικά λεπτομερές αυτό το άρθρο και θα υποβάλω σχετικές τροπολογίες. Όμως πιστεύω ότι θα πρέπει εμείς να υποστηρίξουμε τις ιδέες του συναδέλφου, διότι ε, μη ουσιαστικέ συμβάσεις δεν ωφελούν ε, κανέναν. Πρέπει να βοηθήσουμε τους, ε, τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι κινδυνεύουν καθημερινά στον Μπαγκλαντές. Ευχαριστώ. Η κυρία Βίλς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή για τις ε, προτάσεις του και η πρόταση της Κομισιόν έχει πολύ ενδιαφέρον. Δεδομένου ότι αγνοείται εντελώς, αγνοούνται εντελώς οι διατάξεις της ε, Βασιλείας. Ε, το οι επικίνδυνες ουσίες ε, ε, δηλητηριάζουν ε, και το περιβάλλον και τους ανθρώπους που επιτελούν αυτή τη διάλυση στην Νότια-Ανατολική Ασία και ο Καρλ Σβίτερ μας τα εξήγησε όλα πάρα πολύ σωστά. Η, η εξαγωγή πλοίων με επικίνδυνα απόβλητα τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις της Βασιλείας πρέπει να απαγορευτεί. Και επίσης ε, πρέπει να απαγορευτεί η εξαγωγή πλοίων με ευρωπαϊκή σημαία. Ε, γι' αυτό ακριβώς ε, πιστεύω ότι η πρόταση του εισηγητή για μια έκτακτη εισφορά, μια ειδική εισφορά η οποία θα δημιουργήσει ένα ταμείο το οποίο να χρησιμοποιηθεί για την τελική διάλυση του πλοίου είναι πολύ σωστή. Επίσης πιστεύω ότι όλα τα πλοία πέραν της ασφάλισης ε, που καταβάλουν οι πλειοκτήτες θα πρέπει να πληρώνουν μία επιπλέον ασφάλιση για την διάλυση. Έτσι ώστε να μην υπάρχει αυτή η μεγάλη διαφορά κόστους μεταξύ ε, ευρωπαϊκών και μη ευρωπαϊκών εγκαταστάσεων διάλυσης. Αυτή η συμπληρωματική ασφάλιση θα απέφευγε ένα περαιτέρω αυξημένο κόστος για τη διάλυση των πλοίων σε ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις ή λιμένες. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε εγκαταστάσεις οι οποίες μπορούν θαυμάσια να διαλύσουν τα πλοία και να ε, να αποθέσουν ε, σωστά, με κατάλληλες συνθήκες δηλαδή, τα επικίνδυνα απόβλητα. Έτσι θα αποφύγουμε και το κλείσιμο ε, περαιτέρω ναυπηγείων και εγκαταστάσεων. Και θα μπορέσουμε να χειριστούμε και τα, τις επικίνδυνες ουσίες όπως τον αμύοντο. Έχουμε τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Thank you, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κάποια ερωτήματα για την ε, Επιτροπή. Εγώ δεν είμαι εδώ εμπειρογνώμονα, όπως ο συγγετής μας και η Όμως θα πω το εξής, Να τη συζήτηση με τον κύριο Μπλόκλαντ πριν από κάποια χρόνια. Φαίνεται ότι έχετε παρατηθεί για τις, ε, ό,τι αφορά τη σύμβαση της Βασιλείας. Λέτε δεν λειτουργεί. Και πάμε σε νέα σύμβαση τώρα, προσπάθεια για νέα σύμβαση, αυτή του Χονκ Κόγκ. Ακούγοντας και διαβάζοντας την έκθεση, ακούγοντας τους συναδέλφους, δεν καταλαβαίνω γιατί πιστεύετε ότι αυτή η σύμβαση θα πιάσει τόπο ενώ η προηγούμενη δεν τα κατάφερε. Δεν φαίνεται τίποτα από την πρόταση. Λέτε μια νέα διεθνή σύμβαση με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, ωραίο είναι αυτό, αλλά ε, δεν έχουν φέρει αποτέλεσμα αυτέ οι συμβάσει ω τώρα. Πώ θα καταφέρατε να προσχωρήσουν στη σύμβαση του Χονγκ τα μελη Με του ανθρώπου από τον Μπαγκλαντέ είδατε τι γίνεται. Δεν βλέπω και να αλλάξει τίποτα με τι προσπαθίε σα. Εάν δεν αλλάζει τίποτα, τι είναι αυτό που πραγματικά προτείνεται. Εάν δεν σα αρέσει η ιδέα του κυρίου Σλίτερ για το ταμείο, τι, τι, τι, τι ακριβώς επιδιώκεται. Σε άλλα πέντε χρόνια θα έρθετε και θα μα πείτε τίποτα δεν έχει αλλάξει το μεταξύ. Η ερώτηση λοιπόν είναι τι αλλάζει. Πώ θα βεβαιωθείτε ότι αυτά θα τεθούν σε ισχύ. Είναι πιο αυστηρό ο νόμο τώρα, θα γίνει πιο αυστηρό. Γιατί κανεί δεν προσάγεται, γιατί που δεν έχουμε πρόβλημα οι πλειοκτήτε παγκοσμίω. Γιατί τελικά δεν μπορεί να κάνει τίποτα η αστυνομία. Αυτό αποδέχεσαι στην πραγματικότητα. Πράγματι, πράγματι το θέμα της ε, διάλυσης ή ανακύκλωσης των πλοίων που είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει σε πολλές χώρες ε, της Ασίας είναι διάλυση πλοίων. Ε, δεν τηρούνται οι κανονισμοί ασφαλείας και δεν τηρούνται και οι περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Απ' την άλλη πρέπει να προχωρήσουμε σε ανακύκλωση των υλικών, αλλά με ασφαλή και περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο. Μπορούμε να σκεφτούμε, σε σχέση με όσα είπε ο Κάρλ που έχει κάνει πολύ καλή δουλειά, ήμουν και στην ημερίδα που οργάνωσε, αλλά έχει κάνει πολύ καλή δουλειά και είναι πολύ σημαντικό το φέρνει το θέμα εδώ. Νομίζω πρέπει να αξιοποιήσουμε λίγο και τις σκέψεις που υπήρχαν όταν μιλάγαμε για άλλου είδου απόβλητα και την έννοια της εκτεταμένης ευθύνης του παραγωγού. Δηλαδή ένας παραγωγός έχει την υποχρέωση να διαχειριστεί και μετά το τέλος ζωής ένα προϊόν π.χ. της συσκευασίας. Άρα εδώ πέρα θα πρέπει να σκεφτούμε ότι μια αντίστοιχη αρχή για τις ναυτιλιακές εταιρείες θα πρέπει να εισαχθεί στη συζήτηση. Δηλαδή ένα πλοίο το οποίο κατασκευάζεται να έχει η ναυτιλιακή εταιρεία την υπευθυνότητα απέναντι στην σωστή επανένταξη στον παραγωγικό κύκλο είτε αλλάζει ενδιάμεσα η ναυτιλιακή εταιρεία, είτε πάει σε άλλη σημαία. Αυτό νομίζω είναι ένας κανόνας ο οποίος θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε σε όλο τον κύκλο ζωής ε, το θέμα αυτό με τα πλοία. Τώρα, από την άλλη μεριά, αυτό που συμβαίνει δεν είναι μόνο περιβαλλοντικά ανεύθυνο, έχει να κάνει και με το θέμα της ανταγωνιστικότητας. Επειδή ακριβώς δεν τηρούνται οι προδιαγραφές των ε, συνθήκων εργασίας με ασφάλεια και δεν τηρούνται οι περιβαλλοντικές προδιαγραφές, γι' αυτό Πολλέ από τις δραστηριότητε που θα μπορούσαν να γίνουν σε ευρωπαϊκά ναυπηγεία, σε ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις, πηγαίνουν για λόγους φτηνού κόστου προφανώ σε χώρες που ε, όπου έχουν μια παράδεκτη ε, διαδικασία διάλυσης των πλοίων. Άρα είναι πολύ σημαντικό να βάλουμε κανόνες που θα ισχύουν. Δεν είναι να με τρόπο μη αποδεκτό να ενισχύσουμε τα, τα, ευρωπαϊκά ναυπηγεία, αλλά να βάλουμε ίδιους κανόνες για όπου γίνεται ανακύκλωση πλοίων. Δηλαδή είτε αυτό γίνεται στον Μπαγκλαντές είτε γίνεται στην Ευρώπη να υπάρχουν κανόνες ασφάλειας και περιβαλλοντικές προδιαγραφές ώστε πραγματικά να μιλάμε για σωστές διαδικασίες. Και νομίζω πρέπει να ξεκινήσουμε προφανώ από την Ευρώπη. σω η ιδέα του Κάρλ να έχει ενδιαφέρον σαν ένα ξεκίνημα, δηλαδή μια έκθετη σφορά για να δημιουργηθεί ένα ταμείο στην αρχή με πρωτοβουλία. Δηλαδή ε, με πρωτοβουλία που θα μπορεί μετά να επεκταθεί και σε παγκόσμιο επίπεδο. Και προφανώ χρειαζόμαστε διαδικασίε εφαρμογή των όποιων διεθνών συμφωνιών, γιατί όταν δεν εφαρμόζονται δεν έχουν νόημα. Άρα προφανώ πρέπει η Ευρώπη να δείξει ότι παραμένει στην πρωτοπορία περιβαλλοντικών πολιτικών, που αυτέ μπορούν επίση να δημιουργήσουν και θέσει εργασία και βιώσιμε οικονομικέ δραστηριότητες. Άρα δεν πρέπει κανεί να το δει ότι ε, δημιουργεί οικονομικά προβλήματα, αλλά ίσα ίσα που δημιουργεί νέε ευκαιρίε οικονομική δραστηριότητα και για την επιβίωση ναυπηγείων που σήμερα αντιμετωπίζουν πράγματι μεγάλα προβλήματα. Ευχαριστώ κύριο Τζέμπα. Πρόεδρε, εντυπωσιάστηκα αυτά που μας είπε ο Καρλ. Πράγματι, εδώ πρόκειται για μεγάλο πρόβλημα. Αλλά εξετάζοντας τις προτάσεις αναρωτιέμαι πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα, τις προτάσεις αυτές. Η υλοποίηση λοιπόν. Ε, έχουμε ένα νομοθετικό πλαίσιο, μια νομοθετική βάση. Έχουμε τη Βασιλεία και έχουμε τις προτάσεις του Καρλ. Τώρα, εάν δούμε το σημείο 44 με την πρόταση αυτή για ένα ταμείο που λέει ο Καρλ, είναι μια Πολύ ωραία ιδέα, αλλά εξωπραγματική στον κόσμο μας. Αν θέλουμε να μιλήσουμε ρεαλιστικά, δεν νομίζω ότι η Κομισιόν μπορεί να το εδραιώσει αυτό και δεύτερον δεν νομίζω ότι και πολιτικά θα περάσει μια τέτοια ιδέα. Εγώ πιστεύω ότι πρώτον πρέπει το να αναγνωρίσουμε το πρόβλημα. Αυτό το αναγνωρίζουμε. Δεύτερον να βρούμε μέσα τα οποία είναι εφαρμόσιμα, υλοποιήσιμα ε, το πρόβλημα είναι παγκόσμιο. Ξέρουμε τι δυσκολίες έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, εφαρμόσουμε τα νομοθετήματα. Φανταστείτε τώρα σε διεθνές επίπεδο τι δυσκολία είναι να επιβάλλουμε νομοθετικές ρυθμίσεις. Λοιπόν, μη συζητάμε για ιδέες οι οποίες είναι εξαιρετικά συμπαθητικές αλλά όχι υλοποιήσιμες. Γι' αυτό ακριβώς θέλουμε από την Κομισιόν να εξετάσει με τις αρμοδιότητες και τις δυνατότητες που έχουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Πώς μπορούμε τα, τις δικές μας εγκαταστάσεις, τα δικά μας facilities να τα κάνουμε πιο ελκυστικά. πρέπει να κάνουμε τις δικές μας ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις πιο ελκυστικές για να αξίζει να γίνεται όλη αυτή η διαδικασία στην ευρωπαϊκή επικράτεια. Ίσως με την επιβολή τακτικών ελέγχων, παραδείγματο χάρη προς το τέλος του κύκλου ζωής, ενός πλοίου, ε, ίσως με την ε, επιβολή συμπληρωματικών τραπεζικών εγγυήσεων, ίσως με την ε, ε, υιοθέτηση μέτρων που να βοηθούν στην ε, τον, τελευταία φάση του κύκλου ζωής των πλοίων και την προοπτική της διάλυσης. Ε, βεβαίως υπάρχει μια, ένα μεγάλο ε, οικονομικό χάσμα μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Νοτιοανατολικής Ασίας. Τώρα, εάν εγώ ως κράτος μπορέσω να έχω μία εγγύηση ότι το πλοίο που θα έρθει σε μένα θα διαλυθεί σωστά και ότι υπάρχει η οικονομική κάλυψη, γιατί να μην το δεχτώ. Οι προτάσεις του ΚΑΡ είναι πολύ ωραίες, αλλά έχουν τέτοιες περίπλοκες επιπτώσεις και απαιτούν ε, απραγματοποιητές ε, ε, συνθήκες. Εμείς όλοι θέλουμε, όπως και η Κομισιόν, να εξετάσουμε κατά πόσο μπορούμε να εφαρμόσουμε απλά, απλά ε, χρηματοδοτικά μέτρα. Ίσως με κάποια εισφορά, ίσως με κάποιες επιπλέον εγγύησεις, εισφορές ασφαλιστικές, ε, κάτι να μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να υπάρχει ένα οικονομικό μέσο για τη διάλυση του πλοίου. Αυτά να κοιτάξουμε μέσα στις ρεαλιστικές μας δυνατότητες και πρέπει οι προτάσεις μας να είναι υλοποιήσιμες. Ευχαριστώ τον κύριο Ζέμπερ ο ναυτιλιακός, ο ναυπηγό, υπεσκευαστικός τομέας είναι στην πιο σοβαρή κρίση την οποία έχει περάσει ποτέ. Τρεις, τέσσερα, πέντε, έξι πλοία ε, οι πλειοκτήτες ε, πτωχεύουν καθημερινά και αυτή η ιδέα του Ταμείου ε, και απευθύνουμε πάλι στην Κομισιόν ε, Απευθύνουμε λοιπόν στη Γενική Διεύθυνση ε, μήπως Μήπως αξίζει τον κόπο να εξετάσουμε την ιδέα, να εδραιώσουμε, να δημιουργήσουμε ένα ταμείο. Αυτή τη στιγμή όμως ο εφοπλιστικός κόσμος και οι θα αντιμετωπίζουν ένα τεράστιο πλεόνασμα χωρητικότητας. Και πρέπει να δούμε, υπάρχει αυτή η δυνατότητα να βάλουμε κατάμερα ένα ποσόν πιστώσεις μέσα ενός ταμείου για την διάλυση των πλοίων. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε την ε, πλεονάζουσα χωρητικότητα και δεδομένου το, ότι οι διαλύσεις αυτές των πλοίων αυξάνονται. Γι' αυτό ακριβώς ήθελα να ρωτήσω τη Γενική Διεύθυνση μήπως ε, μπορούμε να επιλύσουμε το πρόβλημα αυτό, δηλαδή ε, οικονομικές, διαφορές κόστους με η πλεονάσα χωρητικότητα με, μια λύση ε, τη δημιουργία ενός ε, χρηματοδοτικού ταμείου ή ενός ταμείου παθεματικού αν θέλετε για τη διάλυση έτσι ώστε να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τον αυπηγοεπισκευαστικό κλάδο και να γίνονται διαλύσεις στην Ευρώπη. Μήπως μπορεί λοιπόν η Κομισιόν να μας απαντήσει, να μας εξηγήσει την προσέγγιση της. Αλλά πριν απαντήσει θα δώσουμε στον Καρλ Χάινς Φλόρενς το λόγο. Ο κύριος Φλόρενς. Ναι, εγώ το βρίσκω πραγματικά πάρα πολύ καλή ιδέα το ότι συζητούμε αυτό το θέμα και η Κομισιόν και ο Σλούτερ. Ε, επειδή η Κομισιόν έχει κάνει καλές προτάσεις και ο Κάρλ επίσης, ο, ο, Ρίχαρτ Τζέμπερ είπε πώς θα τα υλοποιήσουμε όλα αυτά. Όπως παραδείγματο χάρη η οδηγία για τα οχήματα. Εδώ βλέπουμε ότι ε, πολλά κράτη-μέλη κάνουν ό,τι τους κατέβει. Δεν μπορεί να αποφασίσει η Κομισιόν ποιο είναι παλιό όχημα και πότε. Αυτό το αποφασίζει ο διοκτήτης. Λοιπόν, μην μπλέξουμε σε τέτοιες καταστάσεις. Εδώ έχουμε και το πρόβλημα των πρώτων υλών στην Ευρώπη. Εάν λοιπόν είναι αλήθεια ότι κάθε μέρα 4-5 ε, πλειοκτήτες ή ε, πλοία είναι υποπτώχευση τότε θα πρέπει να, να μας βοηθήσει η ευρωπαϊκή βιομηχανία, ο ευρωπαϊκός κλάδος. Πώς μπορούμε να προσανατολίσουμε τον τομέα αυτό στις πραγματικότητες των αγορών. Πρέπει να έχουμε υπόψη πάντοτε την πραγματικότητα των αγορών. Η Βασιλεία, η άλλη σύμβαση, όποια και να είναι. Ε, εντάξει, αυτές υπάρχουν, ε, αλλά δεν, δεν, προσφέρουν και πολλά. Η αγορά έχει το λόγο και οι αγορές ε, ε, πρέπει να πρέπει να, δώσουν το σύνθημα του πώς θα προχωρήσουμε, διότι οι αγορές ενδιαφέρονται για τις πρώτες ύλε που προκύπτουν. Έχω τον κύριο Σκυλακάκη, τελευταίο ομιλητή και τελειώνει κατάλληλος των ομιλητών. Κύριο Σκυλακάκης. Thank you, Mr. President, and Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή για το έργο του και τις ευγενείς του προθέσεις. Όμως, οι ευγενείς προθέσεις δυστυχώς πάντοτε δεν φέρνουν αποτέλεσμα σε αυτό τον τομέα. Άκουσα πολλά για τα ευρωπαϊκά σκάφη. Αυτή είναι μια έννοια νομίζω που θα πρέπει και πάλι να την σκεφτούμε. Δεν ανήκουν τα σκάφη σε χώρες ανήκουν σε πλειοκτήτες και οι πλειοκτήτες μπορούν να αλλάξουν σημαία σε δύο ώρες. Και μπορούν και το κάνουν. Και το κάνουν και μία και δύο και τρεις και τέσσερις φορές αν χρειαστεί. Προκειμένου να διαφύγουν από το χέρι που προσπαθεί να τους επιβάλλει κάτι του νόμου. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός είναι ένας οργανισμός που κινείται με βραδύτητα. Όπως βεβαίως και η Ευρώπη έχει βελτιωθεί πάρα πολύ ε, τα τελευταία χρόνια. Δεν μιλάμε για την ναυτιλία που γνωρίζαμε πριν από 20-30 χρόνια. Η σύμβαση του Χονγκ Κόνγκ που αυτή τη στιγμή δεν έχει κυρωθεί ούτως ή άλλως από κανέναν. Εάν κυρωθεί από τις ε, χώρε στι οποίε κατά κύριο λόγο βρίσκονται εγκαταστάσει, αν μπορούμε να το ονομάσουμε έτσι, για διάλυση, τα πράγματα βαθμιδών ή σταδιακά θα βελτιωθούν λιγάκι. Πάντω θα βελτιωθούν. Μπορούμε να κάνουμε κάτι πολύ περισσότερο όμω. Έχω σοβαρέ αμφιβολίε. Αυτό που συζητούμε είναι εάν μπορούμε να υλοποιήσουμε περιβαλλοντική νομοθεσία στην Κίνα, την Ινδονησία, τον Μπαγκλαντές και το Πακιστάν ενώ δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε την νομοθεσία αυτή, όπως θα δούμε υπό το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δεν βλέπει τι γίνεται στις ε, παραλίες ε, των ευρωπαϊκών χωρών, με τα απόβλητα. Πώς ε, διαχειριζόμαστε τα απόβλητα στην Ευρώπη θα μπορούμε να επιβλέπουμε εγκαταστάσεις που είναι στο άλλο ημισφαίριο του κόσμου. Πώς θα υλοποιηθούν αυτά. Πραγματικά έχω σοβαρούς ενδιασμούς και νομίζω ότι πράγματα μπορούν να γίνουν. Μπορούμε να διευκολύνουμε την υλοποίηση της Σύμβασης του Οι άνθρωποι αυτοί δουλεύουν για 2 δολάρια τη μέρα. Το πρόβλημα δεν είναι ότι ασχολούνται με τη διάλυση και τον μαχισμό μεταλλών, ότι υπάρχει κίνητρο για να δουλέψουν εκεί. Γιατί δεν μπορούν να βρουν δουλειά με 3 δολάρια τη μέρα. Εκεί είναι το πραγματικό πρόβλημα. Αυτό δεν θα αλλάξει με τον κανονισμό που προτείνεται. Ευχαριστώ. Και δίνω τώρα το λόγο στην Επιτροπή για να απαντήσει στα ερωτήματα που προέκυψαν. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ακούσαμε πολύ προσεκτικά τον εισηγητή, καθώς επίσης και τους κοιόδης εισηγητές και όλους τους άλλους που πήρανε το λόγο. Και βέβαια, εκ των προτέρων προτιμάζοντας τη συνεδρίαση αυτή, μελετήσαμε πολύ προσεκτικά την έκθεση του εισηγητή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την εντύπωση ότι όλοι συμμεριζόμαστε εδώ πέρα έναν κοινό στόχο, δηλαδή η ανακύκλωση των πλοίων να γίνει ένα φαινόμενο βιώσιμο σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την εντύπωση ότι ε, συμμεριζόμαστε και τις βασικές ιδέες ε, βάσει των οποίων θα πετύχουμε τον κοινό μας αυτό στόχο, δηλαδή ότι θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένους κανόνες για την ακύκλωση και τη διάλυση των πλοίων, προκειμένου να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε το σύστημα αυτό το οποίο δεν αποδείχτηκε αποτελεσματικό όσον αφορά δηλαδή την υφιστάμενη νομοθεσία για την ανακύκλωση των πλοίων. Εμείς υποστηρίζουμε τη σύμβαση της Βασιλείας και εν προκειμένου δεν λέμε ότι ο κανονισμό Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις μεταφορές των αποβλήτων που αποτελεί ουσιαστικά την ευρωπαϊκή ερμηνεία της σύμβασης της ε, Βασιλείας δεν λέμε ότι θέλουμε να καταργήσουμε αυτόν τον κανονισμό. Αυτό το οποίο λέμε ουσιαστικά είναι ότι η σύμβαση της Βασιλείας ή αν θέλετε ο κανονισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις μεταφορές των αποβλήτων δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το ζήτημα των πλοίων γιατί όπως είπε ο εισηγητής είναι σχεδόν αδύνατο να καταφέρουμε να εντοπίσουμε ένα πλοίο εκείνο το οποίο γίνεται πλέον επικίνδυνο απόβλητο. Γιατί αυτό εξαρτάται τελικά από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη του πλοίου και είναι αδύνατο να δούμε πότε λαμβάνεται αυτή η απόφαση από τον πλειοκτήτη αν η απόφαση ελήφθη επίσης στα χωρικά ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αν τελικά υπάγεται στον κοινοτικό κανονισμό ή όχι. Δύο πράγματα όμως θέλω να τονίσω. Πρώτον, η Σύμβαση της Βασιλείας για τις διασυνοριακές μετακινήσεις επικίνδυνων αποβλήτων θεωρούμε ότι είναι ουσιαστική και επομένως εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι θα πρέπει να επιβάλλεται η σύμβαση αυτή μέσω του δικού μας κανονισμού για τις μεταφορές των αποβλήτων. Και για άλλους τομείς χρησιμοποιούμε τον κανονισμό αυτό και θέλουμε να συνεχίσουμε να το χρησιμοποιούμε και για τομείς όπως για παράδειγμα τα επικίνδυνα ηλεκτρονικά απόβλητα. Βλέποντας τα τελευταία αυτά χρόνια και το πώς εφαρμόστηκε τελικά η σύμβαση της Βασιλείας και ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός που αντιστοιχεί σε αυτήν, Συντοποιούμε τελικά ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί στα πλοία και ότι ουσιαστικά δεν μπορεί να επιβάλλει συγκεκριμένε προδιαγραφέ για την ανακύκλωση των πλοίων. Τα συμβαλώμενα μέρη τη Σύμβαση Βασιλεία ζήτησαν από τον IMO να υπάρχει μια συγκεκριμένη νέα σύμβαση η οποία ασχολείται ακριβώ με το συγκεκριμένο ζήτημα τη ανακύκλωση των πλοίων. Αναγνωρίζει ουσιαστικά ότι έχει, ότι έχει αποτύχει η σύμβαση της Βασιλείας να εφαρμοστεί στην ανακύκλωση των πλοίων. Όλα τα συμβαλώμενα μέρη της σύμβασης της Βασιλείας έχουν πει ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί στα πλοία και γι' αυτό το λόγο θέλουν να εγκριθεί η σύμβαση του Χονγκ Κόνγκ. Άκουσε επίσης ότι ε, υπάρχουν και κάποιες κοινέ ιδέες με τις οποίες συμφωνείτε και οι οποίες ε, υπάρχουν τόσο στην έκθεση του εισηγητή όσο και στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μεγαλύτερη ευθύνη η οποία θα πρέπει να βαρύνει τους πλειοκτήτες καθώς ε, και στην επιλογή που κάνουν για την σημαία όσον αφορά τον κύκλο ζωής του πλοίου, όσον αφορά την δημιουργία του καταλόγου και τις επικίνδυνες ουσίες. Και όλοι συμφωνούμε νομίζω με τον στόχο να καταφέρουμε να εξαλείψουμε εντελώ τις απαράδεκτες αυτές πρακτικές διάλυσης. Καταγράφω λοιπόν τα σχόλιά σας κύριε Σιγητά, καταγράφω τα σχόλια και των άλλων Ευρωβουλευτών και όσον αφορά τώρα κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες για τους χώρους διάλυσης, για τον κατάλογο επικίνδυνων ουσιών κτλ. Καταγράφω και τις σχετικές παρατηρήσεις. Η ανακύκλωση των πλοίων είναι μια οικονομική δραστηριότητα. Τα ναυπηγεία ουσιαστικά προχωρούν σε μια οικονομική δραστηριότητα. Η οικονομική όμως αυτή δραστηριότητα θα πρέπει να γίνεται συμμορφούμενη απόλυτα με την ε, περιβαλλοντική νομοθεσία. Θα πρέπει να σέβεται συγκεκριμένε προδιαγραφέ. Αυτό θα πρέπει να δούμε αν γίνεται ή όχι. Πάντως αποτελεί σε κάθε περίπτωση μια πολύ συμφέρουσα οικονομική δραστηριότητα. Υπάρχουν κάποια πολύ, πολλά μεγάλα πλοία τα οποία έχουν 10.000, πολλές φορές ακόμα και 400.000 τόνους ατσάλι, χάλιβα. Ένας τόνος χάλιβα μετά τη διάλυση είναι 300 περίπου ευρώ. Ένα μόνο πλοίο, ένα και μόνο. 100.000 τόνων για παράδειγμα, που έχει 100.000 τόνους χάλιβα, έχει μία αξία 30 εκατομμυρίων όσον αφορά τον χάλιβα που μπορεί κανείς να πάρει από το πλοίο αυτό μετά τη διάλυσή του. Για τέτοια ποσά μιλάμε. Οι εγκαταστάσει όμως διάλυσης που θα μπουν στο ευρωπαϊκό κατάλογο θα πρέπει να περιλαμβάνουν συγκεκριμένε προεγραφέ και θα πρέπει να τα αποκρίνονται σε συγκεκριμένα κριτήρια. Και ένα από τα κριτήρια αυτά είναι τι γίνεται ακριβώ, πώ διαχειριζόμαστε τα απόβλητα τα οποία απορρέουν από τη διάλυση, τι γίνεται με όλα αυτά τα επικίνδυνα έλεα και το καθεξής. Και θα πρέπει ουσιαστικά να συνάδουν τα κριτήρια αυτά με τη Σύμβαση της Βασιλείας. Δεν εγκαταλείπουμε τη Σύμβαση της Βασιλείας. Το τονίζω ακόμη μία φορά. Και να περάσω τώρα στο κεντρικό σημείο της έκθεσης ε, του εισηγητή, τη δημιουργία δηλαδή αυτού του Ευρωπαϊκού Ταμείου, τις εισφορές που θα πρέπει να συγκεντρώνται σε ένα ταμείο και που θα καταβάλουν οι πλειοκτήτες, οι ναυτιλιακές εταιρείες. Είναι ενδιαφέρουσα η ιδέα αυτή, την έχουμε εξετάσει και στο παρελθόν και έχει απασχολήσει επίσης και τα συμβαλόμενα μέρη της σύμβασης του Χονγκ Κόνγκ και τις διαπραγματεύσεις που έλαβαν χώρα εκεί. Εξετάσαμε και εμείς την ιδέα αυτή επεξεργαζόμενη την πρότασή μας και έχουμε να κάνουμε την ακόλουθη παρατήρηση. Δεν συμπεριλάβαμε την ιδέα αυτή γιατί θεωρούμε ότι ε, στις διαβουλεύσεις που είχαμε με τα ενδιαφερόμενα μέρη και στη δική μας την ανάλυση που κάναμε ήταν πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί στην πράξη δε αυτή γιατί ε, επιφέρει πολλούς, ε, πολλά γραφειοκρατικά εμπόδια. Συμφωνούμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα θετικό κίνητρο. Εμείς λέμε ότι το κίνητρο ενδεχομένω να πρέπει να είναι αρνητικό. Εσείς προτείνετε ένα θετικό κίνητρο, εμείς προτείνουμε ένα αρνητικό κίνητρο. Προσπαθούμε να αποτρέψουμε. Σε κάθε περίπτωση χρειαζόμαστε κίνητρα και θέλουμε να δούμε μαζί σας ποιο είναι το καλύτερο μείγμα κινήτρων το οποίο θα μας επιτρέψει να επιτύχουμε τους στόχους μας. Ο βασικός μας στόχος, το επαναλαμβάνω, είναι όλα τα ευρωπαϊκά πλοία να διαλύονται πακοσμίω με τρόπο ασφαλή και φιλικό προς το περιβάλλον. Τούτων λεγθέντων, θέλουμε να συνεργαστούμε με τον εισηγητή και γενικότερα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να καταλήξουμε σε μια πρόταση αποτελεσματική, η οποία να μπορεί να λειτουργήσει πολύ σύντομα στην πράξη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ίσως μπορέσετε να απαντήσετε και σε μένα. Υπάρχει ανταλλαγή μεταξύ ΕΝΒΗ και της Γενικής Διεύθυνσης ε, για τις επιχειρήσεις. Μήπως υπάρχει δυνατότητα μεταξύ της Επιτροπής μας και της Γενικής Διεύθυνσης ε, να υποβάλουμε μια νέα πρωτοβουλία βασισμένη στην ιδέα του Καρλ για αυτό το ταμείο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι απάντησα στο ερώτημά σα κατά την παρέμβασή μου για την ανακύκλωση των ε, πλοίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, μια, ένα βιομηχανικό κλάδο που γνωρίζει κρίση αυτή τη στιγμή, ξέρουμε ότι τα περιβαλλοντικά πρότυπα ε, γίνονται σεβαστά από τον κλάδο αυτό. Αυτά τα πρότυπα θα ισχύουν και μετά. Όμως εδώ ο κλάδος αυτός είναι ειδικευμένο στην ανακύκλωση άλλου είδους σκαφών, μικρότερων σκαφών που δεν ταξιδεύουν στα νυχτά, στους ωκεανούς και την ανακύκλωση κυβερνητικών και στρατιωτικών σκαφών, κάποιες φορές και πολεμικών. Για τα μεγάλα εμπορικά σκάφη υπάρχει μικρή δυνατότητα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και εντός ΟΣΑ Σκεφτόμαστε ποιε θα είναι οι αναγκαίε επενδύσει σε κεφάλαια και ποιε οι διαδικασίε αδειοδότηση. Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήξαμε και αυτό το μελετήσαμε όχι μόνο με τους συναδέλφους της Γενικής Διεύθυνσης ε, Μεταφορών που είναι συνσυντάκτες της, έκθεσης, ε, πρότασης που έχετε μπροστά σας αλλά και αυτής της Γενικής Διεύθυνσης επιχείρηση, είναι ότι η βελτίωση της δυνατότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα χρειαστεί δεκαετίες. Ε, εάν όχι και περισσότερο γιατί δεν είναι αρκετά οικονομικά ελκυστική. Το πώς οι συνάδελφοι εξετάζουν την πρόταση του συγητή για το Ευρωπαϊκό Ταμείο και με διαλλακτικότητα έχοντας υπόψη ότι όλοι τον ίδιο στόχο επιδιώκουμε δηλαδή την οικοδόμηση δυνατοτήτων εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούμε λοιπόν ότι μια τέτοια λύση θα χρειαστεί ένα πολύ μακρινό ορίζοντα ακόμη και αν επιτευχθεί κάποτε Ευχαριστώ Ευχαριστώ Εδώ νομίζω υπάρχει μια παρανόηση ε, εγώ εννοούσα τους πλειοκτήτες. Τι, συμβαίνει, τι συμβαίνει στα ναυπηγεία θα το δούμε τους ερχόμενους μήνες. Ε, πολλά ναυπηγεία θα πεθάνουν. Ο κύριος Σλούτερ. Ευχαριστώ όλους όσοι ενδιαφέρονται για αυτό το θέμα. Εγώ ενδιαφέρομαι διακαώς ε, τώρα, πολύ περισσότερο από το παρελθόν, διότι είναι τόσο μεγάλο ζήτημα τα χρήματα τα οποία χρειαζόμαστε όταν μιλάμε για τονάζ, για χωρητικότητα, μπορούμε να το ερμηνεύσουμε δύο τρόπους. Είτε το βάρος του πλοίου ε, και τη μετατόπιση του νερού στην οποία οδηγεί το βάρος του πλοίου. Ε, πιστεύουμε ότι 1,5 εκατομμύρια Τονι είναι το όγκος της ε, διάλυσης ευρωπαϊκών πλοίων τα ερχόμενα χρόνια. Ε, το 2015 ίσως 2 εκατομμύρια τόνους. Δεν χρειάζεται να καλύψουμε όλο το ποσό με το ταμείο αυτό, απλώς τη διαφορά μεταξύ του, της υψηλότερης ε, προσφοράς και του κόστους διάλυσης την εγκατάσταση. Έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα, υπολογίζοντας με αυτόν τον τόπο την χωρητικότητα, να έχουμε μια γενική προοπτική του μεγέθους του προβλήματος. Είχα στην αρχή, Κριστόφ, την ίδια προσέγγιση όπως και εσύ. Ας πληρώσουμε όλοι και ας, πληρώ, ας ε, έχουν το δικαίωμα όλοι να έχουν πρόσβαση στο ταμείο. Όλοι καταβάλουν εισφορές, όλοι έχουν πρόσβαση. Αυτό το πιστεύω εγώ ότι ήταν σεμιτό. Τώρα βεβαίως ε, μερικά πλοία εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια μία-δύο φορές μόνο. Οπότε η εισφορά τους στο ταμείο είναι πάρα πολύ μικρή. Τώρα να πληρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση την προστιθέμενη αξία για το παγκόσμιο στόλο, ε, αυτό θα αυξήσει τις απαιτήσει ε, τετραπλάσια ε, οπότε το, η πρότασή μου για το Ταμείο γίνεται πάρα πολύ ακριβή και πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί. Δεδομένου ότι υπάρχει μια εξαιρετικά περίπλοκη διαδικασία ορισμού του πλειοκτήτη. Όπως είπε και ο κ. Κυλακάκη, ο πλειοκτήτη η εταιρεία μπορεί να αλλάξουν σε δύο ώρες και να αλλάξει και σημαία το πλοίο. Παρόλο που κάθε πλοίο είναι καταχωρημένο σε κάποιο νεολόγιο. Γι' αυτό η μόνη μας ευθύνη μπορεί να καλύπτει μόνο τα πλοία με ευρωπαϊκή σημαία. Μόνο για αυτά μπορούμε να μιλάμε. Τότε μπορούμε να πούμε, α, μόνο τα ευρωπαϊκά πλοία ας πούμε θα πληρώσουν. Εγώ πίστευα ότι ο πλούστος τρόπος είναι να πληρώσουν μία φορά όλα τα πλοία, όλα τα πλοία που μπαίνουν σε ένα λιμάνι. Στο δικό μου κράτος μέλος, στη Σουηδία, για να μπορέσουμε να υποχρεώσουμε τους πλειοκτέτες να καθαρίζουν τις δεξαμενές τους, πληρώνουν ένα στάνταρ, μια στάνταρ εισφορά όταν μπαίνουν στο λιμάνι. Είτε καθαρίσεις τις δεξαμενές ούτε όχι, η εισφορά αυτή δεν αλλάζει. Έχουμε λοιπόν μια συγκεκριμένη εισφορά που βασίζεται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες. Είτε κάνεις ε, καθαρισμό είτε όχι. Ρώτησα και την νομική υπηρεσία και για τη σύμβαση της, Βασιλεία της Βασιλείας και για την εισφορά και το πώς μπορεί όλο αυτό το πλέγμα των εισφορών να ε, εδρεωθεί και να καλυφθεί νομικά. Περιμένω ακόμα την απάντηση λοιπόν της νομικής υπηρεσίας στα ερωτήματα αυτά για το ταμείο, τη νομική βάση, τις εισφορές κλπ. Όπως είπατε πολύ σωστά, από πολιτικής απόψεως δεν μπορούμε να κερδίσουμε τη μάχη. Τώρα, στο Βιτόριο απαντώ. Βεβαίω ε, θα μελετήσουμε τι θα απαντήσει η νομική υπηρεσία για τη συμβατότητα της ε, Σύμβασης της βασιλεία. Δεν θέλουμε να διαχωρίσουμε εντελώ ε, το ζήτημα της διάλυσης από τη σύμβαση της Βασιλείας. Οπωσδήποτε θέλουμε να διατηρήσουμε τη σύμβαση. Στην έκθεσή μου κάνω, αναφέρομαι και σε εξαιρέσεις. Λέω, παραδείγματο χάρη, όταν ένα πλοίο, είναι προφανές το ότι χρειάζεται διάλυση όταν οι μηχανές του έχουν πεθάνει, δεν, μπορούν να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω, ε, τότε βεβαίως πρέπει να διαλυθεί. Εν πάση περιπτώσει, περιμένουμε για να δούμε τι, τι διασυνδέσεις μπορούμε να, να διατηρήσουμε με τη Σύμβαση της Βασιλείας όταν μας απαντήσει η νομική υπηρεσία. Τώρα, μια άλλη ερώτηση, σημείωσα, αλλά δεν μπορώ να διαβάσω τις σημειώσεις μου. Κάτι για το Συμβούλιο. Α, το Συμβούλιο δεν έχει ακόμα αρνηθεί, δεν έχει ακόμα απαντήσει αρνητικά. Τα κράτη, μέλη με τα οποία έχω μιλήσει, όλα μου είπαν ενδιαφέρουσα ιδέα, ενδιαφέρουσα ιδέα, αναρωτιέμαι πώς θα λειτουργήσει αυτό το ταμείο. Ε, κανένας δεν μου είπε κατευθείαν όχι το απορρίπτω προς τον κύριο Βαντάλεν. Όπως είπατε, όλη αυτή η αλλαγή θα πάρει χρόνια να εφαρμοστεί και θα έχουμε μία εχμή της διάλυσης πλοίων του 2015 λόγω της πλεονάζωσας χωρητικότητας. Θα είναι καλό λοιπόν να έχουμε ήδη το 2015 ε, κάποιο πλαίσιο υλοποίησης ε, για να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτό την εχμή της διάλυσης το 2015. Ε, αναφερθήκατε επίσης και στα παροπλισμένα, παροπλισμένα πλοία. That's a good idea. Let's see. Ε, τα, τα οποία έχουν εγκαταλειφθεί. Και αυτό θα το εξετάσω. Το άρθρο 23 πράγματι είναι το πιο αμφιλεγόμενο. Όμως, πιο αμφιλεγόμενη είναι η πρόταση της Κομισιόν. Λέει, ε, θα, θα χρησιμοποιήσουμε ένα αρνητικό κίνητρο γιατί είναι πιο εύκολο να κερδίσουμε έτσι. Αλλά εμεί δεν θέλουμε να διευκολύνουμε την αποφυγή των ευθυνών. Ακόμα και αν διατηρήσουμε το άρθρο 23, θα είναι πολύ σπάνια η χρήση του διότι σας συμφέρει οικονομικά να συμμορφώνεστε προς τις διατάξεις παρά να σου επιβάλλουν κυρώσεις, παρά να παρανομείς και να είσαι σήμα, ας πούμε, των κυρώσεων και των ποινών. Δεν σας συμφέρει να παρανομείς, σας συμφέρει να είσαι ένομος. Όσον αφορά την κρίση στην στον ναυπηγό επισκευαστικό τομέα, όντω υποφέρει από τεράστια κρίση. Αλλά η διάλυση, ο όγκος των πλοίων υποδιάλυση αυξάνεται. Εγώ προτιμώ να ε, προχωρήσουμε προς μία αυτοχρηματοδοτούμενη λύση. δυστυχώς ε, πιστεύω και εγώ ότι όταν μπορούν να αποφύγουν τον νόμο οι άνθρωποι δεν ακολουθούν τους νόμους. Προσπαθούν να βρουν παρασυράκια. Αλλά το θέμα είναι ότι όλα αυτά πρέπει να τα εξετάσουμε στο πλαίσιο της πρόταση του Ταμείου. Ρίτσαρτ, εσύ ανέφερες ότι ό,τι λύση προτείνουμε πρέπει να είναι υλοποιήσιμη ε, και ρεαλιστική πιστεύω ακράδαντο ότι η πρότασή μου έτσι είναι. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα θέμα, ένα πλαίσιο το οποίο να βασίζεται στις αρνητικές ε, πρωτοβουλίες. Επειδή η εφαρμογή της βασιλείας είναι ε, αναπερκέστατη, δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αυτό ως δικαιολογία. Εγώ πιστεύω ότι οι λύσεις μου είναι ρεαλιστικές. Ε, δεδομένου ότι καταβάλλονται εισφορές στο λιμάνι με την είσοδο των πλοίων, προσθέτουμε μία γραμμούλα που να λέει ότι ένα μέρος της εισφοράς ή μία επιπλέον εισφορά θα πηγαίνει προς αυτό το ταμείο για τη διάλυση. Εφόσον θα έχουμε ένα κατάλογο ευρωπαϊκών εγκαταστάσεων, που δεν είναι και τόσες πολλές, ε, τα θα διοχετεύονται τα χρήματα αυτά της ειδική εισφοράς στο ταμείο και από εκεί θα πηγαίνουν σε αυτές τις όχι και τόσο πολύ άρισμες εγκαταστάσεις. Ε, άρα το πρόβλημα δεν έχει τόσο τεράστια γραφειοκρατία και ούτε είναι τόσο μεγάλο το κόστος ε, συμμόρφωσης. Για την τραπεζική εγγύηση που και αυτή μπορεί ανήκει στις ε, αρνητικές, στα αρνητικά κίνητρα, οι τραπεζικές ε, πρόσθετες εγγύησεις θα οδηγήσουν σε περισσότερη γραφειοκρατία, διότι το καθεστώς εγγυήσεων που καταβάλει ο πλειοκτήτης αλλάζει κάθε φορά που το πλοίο αλλάζει πλειοκτήτη ή αλλάζει σημαία. Ενώ αυτό το οποίο εγώ προτείνω είναι μία καταβολή μαζί με την εισφορά εισόδου στο λιμένα, η εισφορά και για το ταμείο αυτό, μία φορά θα γίνεται αυτό. Μία διαδικασία, χωρίς επιπλέον γραφειοκρατία. Οπότε, όταν θα έρθει η στιγμή της διάλυσης του πλοίου, τότε θα καταβάλλεται η ενίσχυση. Θα καταβάλλεται το ποσό αυτό από το Ταμείο, στην τελική φάση, στο, στην τελική διαδικασία. Και ο Θόδωρος ναι, βεβαίως δεν μπορούμε να βελτιώσουμε το ημερομίσθιο των 2 δολαρίων με αυτά τα οποία προτείνουμε, δυστυχώς. Όμως αυτό το οποίο προσπαθούμε να δημιουργήσουμε είναι να δώσουμε κίνητρα στις εταιρείες διάλυσης να, να μπουν στον ευρωπαϊκό κατάλογο και να έχουν πρόσβαση σε αυτό το ταμείο. Θα δημιουργηθούν έτσι περισσότερα κίνητρα για, τη βελτίωση των, για τις επενδύσεις, τη βελτίωση των εγκαταστάσεων ε, των ευρωπαϊκών. Ε, ε, είμαι αρκετά αισιόδοξο. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, αλλά το να έχουμε μία μη εφαρμόσιμη, μη λειτουργική σύμβαση του Χονγκ Κόνγκ παράλληλα με τη μειονεκτική σύμβαση της Βασιλείας δεν είναι λύση. Ευχαριστώ και έτσι ολοκληρώνουμε ε, τη συζήτηση των θεμάτων 5 και 6. 7 Δεκεμβρίου θα συζητήσω, είναι οι τροπολογίες, ε, συγγνώμη, 17 Δεκεμβρίου είναι η ε, προθεσμία τροπολογιών, θα ψηφίσουμε ψηφίσουμε στις 19 Ιανουαρίου και θα μπει στην ημερήσια διάταξη του Απριλίου. Ευχαριστώ ε, πολύ. Συγγνώμη, η προθεσμία απολογίου είναι 5 Δεκεμβρίου. Έκανα λάθος, 5 Δεκεμβρίου και Ολομέλεια τον Απρίλιο. Ωραία, προχωρούμε στο σημείο 7. Βελτίωση των ωφελών από τα περιβαλλοντικά μέτρα, οικοδόμηση εμπιστοσύνη μέσω τη βελτίωση τη γνωστική βάση και τη ικανότητα απόκριση των αρχών. Και δίνω το λόγο στον κύριο Ορέστε Ρώση, τον εισηγητή. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω με μία παρατήρηση που ε, έγινε ήδη και για τα πλοία, δηλαδή ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε προσεκτικοί κάθε φορά που εγκρίνουμε μέτρα τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν τελικά σύγχυση, γιατί τότε χάνουμε όχι μόνο ανταγωνιστικότητα, αλλά ενδεχομένω να κλείσουν και κάποιες εταιρείε οι οποίες πηγαίνουν σε πιο εύκολε χώρε. Και όταν λέω εύκολε, ενώ χώρε οι οποίε τελικά δεν ανταποκρίνονται στι ευρωπαϊκέ προδιαγραφέ, ιδίω από περιβαλλοντική πλευρά. Κατά αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, μπορεί να αυξηθεί περισσότερο η μόλυνση και η ρήπανση του περιβάλλοντο. Στην έκθεσή μου, λοιπόν, λέω ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας μεγαλύτερος διάλογος τόσο με τις επιχειρήσεις, με τα κράτη-μέλη, αλλά και εμείς θα πρέπει ενδεχομένω να μιλάμε περισσότερο με τη Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για το Περιβάλλον και με τον Επίτροπο Ταγιάννη. Διακόπτει ο Πρόεδρος, παρακαλώ πολύ, όσοι δεν θέλουν να συμμετάσχουν στη συζήτηση, παρακαλώ να αποχωρήσουν ηρέμως από την αίθουσα για να μπορέσει να ακούσουμε τον εισηγητή. Σας έλεγα λοιπόν ότι στη διαφορετική περίπτωση ενδεχομένω να μην είναι πάρα πολύ εύκολο να εφαρμοστούν τα περιβαλλοντικά μέτρα και κατά αυτόν τον τρόπο απομακρυνόμαστε από το στόχο μας, δηλαδή όλα τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν με τον ίδιο τρόπο τα περιβαλλοντικά μέτρα. Στην ε, προηγούμενη συνεδρίασή μας ε, είχαμε αναφερθεί στην, ε, στο ζήτημα αυτό είναι δεχομένω σύντομη η έκθεσή μου. Υπάρχει ένας περιορισμός όσον αφορά όμως το λέξεις μπορώ να χρησιμοποιήσω. Θα γίνουν προφανώς κάποιες τροποποιήσεις, τροπολογίες από τους συναδέλφους. Ποια είναι τα βασικά σημεία. Τα βασικά σημεία είναι καταρχάς οι επιπτώσεις, οι επιπτώσεις της ε, περιβαλλοντική νομοθεσίας, οι απλοποιήσεις και η μείωση των διοικητικών φραγμών, που μπορούν ουσιαστικά να οδηγήσουν σε μια καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας, μια μεγαλύτερη διαφάνεια και δημοσιότητα των διοικητικών διαδικασιών στον τομέα του περιβάλλοντος, καθώς επίσης και εγγυήσεις πρέπει να δοθούν για ευκολότερη πρόσβαση των πολιτών στην περιβαλλοντική δικαιοσύνη. Όλα αυτά τα προβλήματα ουσιαστικά είναι αλληλένδετα. Πρέπει να γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι πριν και μετά την εφαρμογή των περιβαλλοντικών μέτρων να δούμε επίσης αν εφαρμόζεται η αρχή της επικουρικότητας, της αναγκαιότητας, αν επίσης ανταποκρινόμαστε πραγματικά στην πρόκληση της επικουρικότητας. Βλέπουμε ότι πάρα πολλές παραβιάσεις στην περιβαλλοντική νομοθεσία, μάλλον στην κοινοτική νομοθεσία, έχουν να κάνουν με το περιβάλλον. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι πάρα πολλές καταγγελίες δεν γίνονται γνωστές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να διορθωθεί το πρόβλημα αυτό και θα πρέπει να βρεθούν κάποιες λύσεις. Ποιες είναι οι λύσεις που μπορούμε να προωθήσουμε, που εγώ προωθώ, αλλά θα ακούσω και τους συναδέλφους. Καταρχάς, μια καλύτερη εφαρμογή της περιβαλλοντικής κοινοτικής νομοθεσίας, δηλαδή διορθωτικά μέτρα σε κέριους τομείς με μια καλύτερη διοργανική, διαθεσμική συνεργασία. Μια ένας καλύτερος συντονισμός στον κοινοτικό προπολογισμό για το περιβάλλον, μια καλύτερη ενημέρωση επίσης, δηλαδή να καταφέρουμε να διαχέουμε καλύτερα τις βέλτιστες πρακτικές ανάμεσα στην Ένωση και τα κράτη-μέλη όσον αφορά την περιβαλλοντική νομοθεσία. Επίσης πρέπει να υπάρχει μια καλύτερη διάχυση και ενημέρωση των περιβαλλοντικών προγραμμάτων της Ένωσης. Επίσης μια καλύτερη διοικητική οργάνωση για τη συλλογή δεδομένων, για τη διάχυση αυτών των πληροφοριών, για την πρόσβαση στις πληροφορίες σε όλα τα επίπεδα. Ότι θα πρέπει να έχουμε καλύτερη συνεργασία ανάμεσα στο κοινοτικό, το εθνικό και το περιφερειακό επίπεδο. Καλύτερη ασφάλεια δικαίου επίσης. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να κάνει μια διεξοδική ανάλυση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Θα πρέπει επίσης να αξιολογήσουμε κάποια συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα έχουν ως στόχο να, να μειωθεί το διοικητικό κόστος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον χωρίς όμως να δημιουργούμε περισσότερα διοικητικά περισσότερους διοικητικούς φραγμούς και περισσότερες δαπάνες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε ποιο τομέα θα πρέπει να αποκρίνεται σε ποια περιβαλλοντικά μέτρα. Για παράδειγμα, να πούμε ότι η αυτοκινητοβιομηχανία θα πρέπει να σέβεται συγκεκριμένους, συγκεκριμένα περιβαλλοντικά μέτρα. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια λογική, απλή προσέγγιση σε αυτή την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Επίσης πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια διάχυση των δεδομένων και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Επίσης, θα πρέπει να τονιστεί περισσότερο το ζήτημα της περιβαλλοντικής ευθύνης συγκεκριμένων ε, επιχειρήσεων. Επίσης, θα πρέπει και οι ίδιοι οι πολίτες να έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση όσον αφορά την περιβαλλοντική νομοθεσία. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχουν ε, να καταφέρουμε να εντοπίσουμε τα κατάλληλα περιβαλλοντικά μοντέλα τα οποία θα πρέπει να εφαρμοστούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να δούμε επίσης ε, πώς μπορούμε να επιλύσουμε κάποια προβλήματα τα οποία έχουν ε, προκύψει. Όχι μόνο δηλαδή να έχουμε κυρώσεις, αλλά να καταφέρουμε να πείσουμε τις εταιρείε ότι ε, η εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας είναι προς το συμφέρον όλων. Ότι δεν αποτελεί δηλαδή επιβάρυνση βάρος, αλλά τελικά ότι είναι ένα πλεονέκτημα, ένα συμφέρον. Επίση, είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε τι γίνεται με την περιβαλλοντική νομοθεσία και τι επενδύσει. Θα πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε τι εταιρείε για να εφαρμόζουν την περιβαλλοντική νομοθεσία θα πρέπει να καταφέρουμε να δίνουμε τα απαραίτητα, τα απαραίτητα κίνητρα σε εταιρείε αυτέ προκειμένου να εφαρμόζουν την περιβαλλοντική νομοθεσία και να παραμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να μην πηγαίνουν σε άλλε χώρε όπου θα λειτουργούν χωρί περιγραφέ και τελικά θα μολύνουν περισσότερο. Πιστεύω λοιπόν ότι Όλα αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να εξεταστούν και στο πλαίσιο του θεμητού ανταγωνισμού. Ολοκληρώνω στο σημείο αυτό, ανέφερα τα σημεία αυτά στα οποία θεωρώ ότι θα πρέπει να επιμείνουμε πολύ περισσότερο. Πρώτον, υπάρχει ένα καλύτερο διάλογο σε όλα τα επίπεδα. Αυτό ισχύει για τη δική μα την Επιτροπή, ασχύει επίση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ισχύει και για τι εταιρείε. Από την άλλη, οι επενδύσεις στο περιβάλλον δεν αποτελούν παράλογες δαπάνες ή μία δαπάνη που γίνεται άνευ Θα πρέπει μέσω των επενδύσεων αυτών να καταφέρουμε να βελτιώσουμε την υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία προς το συμφέρον όλων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, σκιώδης εισηγητής, ο κύριος Φλόρενς. Ε, ε, ε, αγαπητέ πρόεδρε, όπως ξέρετε εγώ έχω μια εντελώς αντίθετη άποψη. Στο τέλος είπατε ότι έχετε την μεγάλη ανησυχία, ότι μπορεί η ευρωπαϊκή βιομηχανία να εξαχθεί. Εγώ πιστεύω ότι η έλλειψη ανταγωνιστικότητας μέσα στην Ευρώπη με στεναχωρεί πολύ περισσότερο. Αν δω τι γίνεται στη χώρα μου και στην Ιταλία τι γίνεται, Παραδείγματο χάρη την οδηγία συσκευασία. Ε, τότε βλέπετε στην, ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ιταλία ε, δεν έχει γίνει τίποτα και άλλες χώρες όπως η δικιά μου το παρακάνει. Δεν λέω, ομολογώ αυτό είναι δικό μας πρόβλημα. Κοιτάω προς την Κομισιόν. Πολύ λυπάμαι που η Γενική Διευθύντρια δεν είναι πλέον εδώ, αλλά αν ρωτήσετε τον Επίτροπο μας λέει ότι το βασικό μας πρόβλημα είναι η έλλειψη της ε, μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Και αυτό, αυτό λοιπόν με οδηγεί στο να πω ότι Πού γίνεται τέλος πάντων κάτι σωστό. Συμφωνώ με τη μείωση των ρυθμίσεων και των κανόνων, περισσότερη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων, αλλά ας αρχίσουμε τέλος πάντων αυτά τα οποία είναι εφαρμόσιμα και να μεταφέρουμε αυτά. Η Κομισιόν δεν έχει το δικαίωμα να πάρει δείγμα νερού κοντά στο Στρασβούργο, στο Κέλ, για να διαπιστώσει εάν το εργοστάσιο χρησιμοποιεί τις σωστές πρώτες ύλες ή όχι. Δεν έχει το δικαίωμα λοιπόν να πάρει αυτό το δείγμα. Πρέπει να μπορούμε να έχουμε συγκρίσιμα και μετρήσιμα στοιχεία. Δεν μπορεί να θέτουμε τον πύχη πάντοτε τόσο ψηλά. Γι' αυτό πρέπει να πιάσουμε τα κράτη-μέλη, τα προβληματικά από το λαιμό, από το γιακά, και αν δεν το κάνουμε αυτό δεν θα υπερψηφίσω, δεν συμφωνώ με την πρόταση αυτή και ε, έχω συμφωνήσει και με, τις, με άλλες μεγάλες ομάδες να ενισχύσω αυτή την έκθεση προς τη δική μας κατεύθυνση και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα που μας έχετε δώσει λίγο χρόνο περισσότερο να διαβουλευτούμε. ο κύριος Λάινεν. Η υλοποίηση του κοινοτικού και εκτιμένου φαίνεται ότι είναι πολύ προβληματική για ορισμένους συναδέλφους. Βέβαια, είναι μεγάλο σημώνει αγανακτή κανείς όταν έχει συμβάλει στην νομοθετική, στην νομοθεσία, στη δημιουργία της νομοθεσίας και μετά βλέπει ότι δεν εφαρμόζονται αυτοί οι νόμοι. Όμως πιστεύω ότι ο κύριος Φλόρεντς έχει παρανοήσει την πρόθεση της Κομισιόν. Η πρόθεση της Κομισιόν ε, προέρχεται από την έκθεση για το περιβάλλον και ε, η, έκθεση του κυρίου, η πρόταση του κυρίου Ρώση τονίζει τα μειονεκτήματα της περιβαλλοντικής πολιτικής. Ε, πιστεύω ότι η έκθεση έχει πετύχει σωστά ορισμένα θέματα. Όμως ξεκινάει από μια αρνητική αρχή, από την μια αρνητική βάση. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να αναποδογυρίσουμε την πρόταση αυτή. Δηλαδή, η πολιτική την οποία εμείς ακολουθούμε εδώ στην ΕΝΒΗ να ε, αντανακλάται σε αυτά τα οποία ζητούμε από την Κομισιόν και αυτά τα οποία λέμε στο δημόσιο, στην κοινή γνώμη. Θέλουμε όλοι να συγχρονίσουμε, να εφαρμόσουμε καινοτομίε και ξέρουμε ότι μη εφαρμογή των κανόνων ε, έχει και ε, οικονομικές επιπτώσεις. 500 δισεκατομμύρια ευρώ είναι το ύψος των επενδύσεων που μπορούμε να επιτύχουμε. Αναφέρθηκε ο, ο εισηγητής, ο κύριος Ρώση, στο θέμα της επικουρικότητας, όμως η επικουρικότητα δεν είναι θέμα υλοποίησης, δεν είναι θέμα εφαρμογής. Εμείς είμαστε μια κοινότητα δικαίου και θα πρέπει και στις 27 χώρες να ταυτόχρονα και ισότιμα να μεταφέρεται η νομοθεσία στο το, τοπικό επίπεδο και περιφερειακό είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι μέσα στα πλαίσια αυτά υλοποιείται η νομοθεσία. Όμως πιστώσεις δεν βοηθούν, δεν είναι η μόνη λύση διότι έχουμε και ε, μεγάλες ελλείψεις στις δυνατότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης, ε, γενικά στη διοίκηση. Έχουμε ελλείψεις, έχουμε προβλήματα για τη μεταφορά των κανόνων, την εφαρμογή τους και υπάρχουν ε, τοπικές αυτοδιοίκησεις, παράγοντες, φορείς οι οποίοι μεταφέρουν τις κοινοτικές, το κοινοτικό πλαίσιο πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ σωστά, άλλες όμως τα χάνουν. Ε, κατακλείζονται από μια χιονοστιβάδα κανονισμών και δεν ξέρουν καθόλου πώς να τη χειριστούν και πώς να μεταφέρουν στο εθνικό επίπεδο. η, πρώτη μας προτεραιότητα τα <laughs> επόμενα έξι χρόνια είναι εφαρμογή, εφαρμογή, εφαρμογή και χρησιμοποίηση όλων των μέσων και εφαρμοστικές ε, συνεργασίες αν θέλετε. Είμαι βέβαιη, βεβαίως ότι η Κομισιόν μαζί με όλους τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης θα πρέπει να συνεργαστεί για να τους βοηθήσει στη σωστή και ισότιμη εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου, εκεί που έχουν δυσκολίες. Σύμφωνο ε, με τον κύριο Φλόρεντς και λέω ότι πρέπει να αναδιατυπώσουμε την έκθεση. Θα δούμε τι θα προκύψει από τις τροπολογίες. Κύριε Ρώση, θα ήθελα μια πιο θετική προσέγγιση. Τονίζετε πολύ τις ελλείψεις και τα μειονεκτήματα. Εγώ περισσότερο θέλω να τονίσετε τα πλέον εκτήματα. Ο πρόεδρος. Λοιπόν, βάσει τη σειρά των προηγούμενων <laughs> προέδρων, δίνω το λόγο στον κύριο Σκυλακάκη. I would, uh, first like to start by saying... Να ξεκινήσω λέγοντας ότι έχουμε σοβαρές διαφωνίες με τα συμπεράσματα του συζητή. Εναλλακτικές απόψεις θα τις έλεγα. Για την περιβαλλοντική πολιτική, ένα πράγμα είναι βέβαιο. Δεν την υλοποιούμε όπως θα έπρεπε. Ούτε έχουμε σοβαρούς μηχανισμούς ελέγχου της υλοποίησης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Νομίζω ότι θα έπρεπε να έχουμε περισσότερα κεντρικού χαρακτήρα και ισχυρά εργαλεία και οχήματα για να ελέγχουμε κατά πόσον η υλοποίηση τη νομοθεσία μα επιτυγχάνει του στόχου τη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να δείξει περισσότερη πυγμή και θα συμφωνήσουμε με τον κύριο Φλόρεν ω προ αυτό. Επίση, να επισημάνω ότι χρειαζόμαστε περισσότερη συμμετοχή των πολιτών. Πρέπει να το επιδιώξουμε αυτό, αλλά με συνθήκε υπευθυνότητα. Διότι έχουν προκύψει φαινόμενα όπου οι πολίτε συμμετέχουν αλλά όχι για περιβαλλοντικούς σκοπού με άλλα κίνητρα σε κάποιες χώρες κάποιοι χρησιμοποίησαν την νομοθεσία αυτή για να προσφύγουν δικαστικώς κατά κάποιων επενδύσεων χωρίς ε, σοβαρούς λόγους. Δηλαδή αν κάποιος έχει δίκιο να μπορεί να διακόψει μια διαδικασία. Αλλά αν όχι, να μην ε, λειτουργεί ω τροχοπέδι για όλη την κοινωνία. Χρειαζόμαστε επενδύσει που να είναι φιλικέ προ το περιβάλλον. Και κάποιοι τη χρησιμοποιούν την νομοθεσία μα. Την εκμεταλλεύονται. Και κάτι τελευταίο. Ε, στο παρελθόν, η περιβαλλοντική νομοθεσία έχει χρησιμοποιηθεί για σκοπού βιομηχανική πολιτική. Δηλαδή, προκειμένου να υπάρξει κέρδο για τομείς και κλάδου που έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αυτό δεν θα πρέπει να συμβαίνει στο μέλλον. διότι και αυτό το φαινόμενο υπονομεύει το, τους ισότιμους κανόνες που θέλουμε να έχουμε. Ευχαριστούμε, Κρίστα Κλάφ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Φλόρενς όταν λέει ότι χρειαζόμαστε εναρμονισμένη υλοποίηση σε όλα τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να μπορούμε να διεξαγάγουμε ελέγχους για την περιβαλλοντική νομοθεσία όταν χρειάζεται. Όταν πρόκειται για τα φυτογειονομικά ε, μέτρα, τη νομοθεσία για τα ζεζανιοκτώνα, θα πρέπει να βεβαιωθούμε για σκοπούς ε, προστασίας των εργατών ότι η νομοθεσία υλοποιείται παρομοίως σε όλη την Ευρώπη. Αλλά κάποιες φορές οι ίδιοι υποσκάπτουμε τη θέση μας. Διότι η νομοθεσία μας εξελίσσεται με γοργά, αλλά εμείς μεταξύ δεν έχουμε το χρόνο να την αφομοιώσουμε. Δηλαδή, έχουμε κάποια ευθύνη εδώ. Δεν μπορούμε να σκορπιζόμαστε δεξιά και αριστερά. Θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξασφαλίσει μια σχετική συνοχή μεταξύ των διαφορών κειμένων, ε, κανονισμών και οδηγιών. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν επικαλύψεις. Ε, Α πούμε για την αποψήλωση των δασών. Εδώ απευθύνω έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συχνά κάποια πράγματα που συζητούμε εδώ φαίνονται να είναι ιδιαίτερα θεωρητικά. Πολλές φορές και μαθηματικού χαρακτήρα. Και φαίνεται δύσκολο να γίνουν χειροπιαστά βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Στην κάθε χώρα υπάρχουν ε, διαφορετικά μερικοί βαθμή επιτυχημένης υλοποίηση. αλλά φαίνεται να μην ε, είναι τόσο απλό να αποτιμηθεί η προστιθέμενη αξία νέων νομοθετημάτων. Νέε θέσει απασχόληση λοιπόν, ναι, αλλά θα πρέπει κάποιο να τι πληρώνει. Θα πρέπει να δοθεί λοιπόν μεγαλύτερη αξία στην περιβαλλοντική μα πολιτική. Αυτή είναι μια τεράστια πρόκληση και θα πρέπει να θέσουμε στου εαυτού μα το ερώτημα. Και εμεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώ θα πετύχουμε να πάρουμε την κοινωνία με το μέρο μα. Θα πρέπει η υλοποίηση σε κάθε κατός να δείχνει την αξία ακριβώ αυτή τη πολιτική. Αυτή είναι η πραγματική πρόκληση. Ευχαριστούμε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, thank you, Mr. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε έρθει ιδιαιτέρως που έχετε διορίσει έναν εισηγητή, ο οποίος θα συντάξει έκθεση, συνέταξε έκθεση για τη δική μας ανακοίνωση. Μια-δυο παρατηρήσεις. Η ανακοίνωση αυτή, καταρχάς, καταδεικνύει την προτεραιότητα που ο αρμόδιος επίτροπος δίνει για την νομοθεσία αυτή. Μέσω της ανακοίνωσης αυτής θέλαμε να αφαιρθούμε σε κάποιες βασικές ιδέες που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε με το στόχο αυτό. Όσον αφορά τώρα τα πιο ιδιαίτερα σημεία, νομίζω ότι μπορούμε και στα πλαίσια της ανακοίνωσης να πούμε ότι έχουμε έξι βασικές ιδέες. Πρώτον, γνώση γνωστική βάση. Κάτι το οποίο ακούσαμε στις παρεμβάσεις πριν από λίγο. Το πόσο σημαντικό είναι να καταφέρουν όλοι όσοι εφαρμόζουν την περιβαλλοντική νομοθεσία να έχουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να βελτιώσουμε την ροή των γνώσεων και τη ροή των βέλτιστων πρακτικών. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει περισσότερες πληροφορίες να είναι διαθέσιμες ε, επιγραμμικά, προκειμένου να γνωρίζουν όλο και περισσότεροι πώς εφαρμόζεται επιτόπου η παρβαλλοντική νομοθεσία. Μία άλλη ιδέα έχει να κάνει με τη δημιουργία δικτύων, δικτύων εμπειρογνωμόνων. Αυτό περιλαμβάνει βέβαια πολλά διαφορετικά δίκτυα. Ήδη συνεργαζόμαστε με ένα δίκτυο δικαστών που επιτρέπει στη δικαστική εξουσία παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταλλάσσει πληροφορίε όσον αφορά συγκεκριμένε δίκε ή προσφυγέ που έχουν να κάνουν με την παραβολοντική νομοθεσία. Ένα πολύ καλό πρακτικό τρόπο λοιπόν προκειμένου να καταφέρουν τα κράτη-μέλη και οι δικαστέ αυτά τα κράτη-μέλη να παραμένουν ενημερωμένοι για τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Έχουμε και ένα άλλο δίκτυο ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και θα συνεργαστούμε επίση και με την Επιτροπή των Περιφερειών προκειμένου να καταφέρνουμε να αναφερόμαστε περισσότερο στα ζητήματα εκείνα τα περιβαλλοντικά που απασχολούν πιο που απασχολούν περισσότερο, με συγχωρείτε, την τοπική και περιφερειακή διοίκηση. Αναφέρθηκε και σε όλα αυτά τα ζητήματα ο κύριος Ρώση. Πρόσβαση επίσης σε περισσότερες πληροφορίες, το ανέφερε αυτό και ο κύριος Ρώση και άλλοι ευρωβουλευτές, Επεξεργαζόμαστε το σημείο αυτό περισσότερο, κάναμε κάποιες μελέτες. Το Δικαστήριο επίσης Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αποφανθεί για το ζήτημα αυτό. Το 2003 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μια πρόταση που δεν σημείωσε όμως την απαραίτητη πρόοδο. Έκτοτε όμως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει την απαραίτητη πλέον ε, νομολογία που ε, επιτρέπει σε όλους περισσότερους πολίτες να προσφύγουν στα εθνικά δικαστήρια για παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Και αυτό θα θέλαμε να μας απασχολήσει περισσότερο και να συνεργαστούμε για το ζήτημα αυτό μαζί σας. Άλλα ζητήματα έχουν να κάνουν με μηχανισμούς αντιμετώπισης κάποιων καταγγελιών και σε αυτό αναφέρθηκε ο κύριος Ρώση. Πώς μπορούμε δηλαδή να εξασφαλίσουμε ότι οι πολίτες μπορούν με επικοδομητικό τρόπο να βρουν το δίκαιο τους κάθε φορά που προσφεύγουν ή που κάνουν καταγγελίες στις εθνικές αρχές για παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Τελευταίο σχόλιο. Πολύ μεγάλη σημασία δίνουμε και στο ζήτημα των ελέγχων, των επιθεωρήσεων. Πάρα πολλά από τα προβλήματα τα οποία εντοπίζουμε τελικά απορρέουν από το ότι δεν έχουν γίνει επιτόπιοι απαραίτητοι έλεγχοι. Αυτό το βλέπουμε παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν βέβαια και ορισμένα κράτη-μέλη τα οποία έχουν πολύ καλές προσεγγίσεις στο ζήτημα αυτό, έχοντας ένα πολύ μικρό, γραφειοκρατικό άχθος και καταφέρνουν να κάνουν τους απαραίτητους ελέγχους. Θέλουμε οι βέλτιστες αυτές πρακτικές να γίνουν ένα κοινό πρότυπο παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Πρόεδρε, λοιπόν, βλέπετε ότι προσπαθούμε να επεξεργαστούμε πολλές διαφορετικές πρωτοβουλίες και ελπίζουμε ότι κάποιες από τις πρωτοβουλίες αυτές θα αποτελέσουν τμήμα του εβδόμου προγράμματος δράσης που ελπίζουμε να υλοποιηθεί πολύ γρήγορα. Σας ευχαριστώ. Möchte Μήπως θέλει ο να παρέμβει πάλι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα κυρίως να ευχαριστήσω τους συναδέλφους της Επιτροπής. Ιδίω ο πρόσωπος της Επιτροπής σωστά έκανε κάποιες επισημάνσεις, θα συμφωνήσω μαζί του. Πρόσβαση στη δικαιοσύνη, σεβασμός των δικαιωμάτων πολιτών, Ευαισθητοποίηση, ενημέρωση. Συμφωνώ απολύτω. Σε ό,τι αφορά τώρα τι παρατηρήσει των συναδέλφων. Νομίζω για όσα είπε ο κύριο Φλόρεν ότι πρέπει να βελτιστοποιηθούν οι κανόνε. Σωστό είναι και αυτό και πρέπει να εφαρμόζονται κιόλα. Δηλαδή και εύληπτοι και υλοποιήσιμοι κανόνε. Ε, αυτό μα βρίσκει απολύτω σύμφωνο. Το είπε και η κυρία Κλάσ. Για το πώ θα πρέπει να είναι οι κανόνες υλοποιήσεων με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα κράτη. Αν θέλουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία να λειτουργεί εύρυθμα, θα πρέπει οι κανόνες να είναι ίδιοι για όλους. Για τον κύριο Σκυλακάκη. Είπε ότι υπάρχουν αναλλακτικέ προτάσεις και ότι δεν συμφωνεί και τόσο με τα συμπεράσματα της έκθεσης και ότι θα έπρεπε να είναι πιο ισχυρή παρέμβαση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι η απάντηση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν ακριβώ αυτή που περιμέναμε. Μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών τώρα. Και εγώ το είπα και το επανέλαβε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βεβαίω θα δούμε τι τροπολογίε σα και ελπίζω ότι θα μπορούμε να τι κάνουμε και δεκτέ. Ο κύριο Λάινεν. Ξέρετε ότι τον άφησα τελευταίο γιατί πολλέ φορέ τσακωνόμαστε, βλέπουμε τα πράγματα λίγο διαφορετικά, συνάδελφοι. Παρ' όλα αυτά είπε ότι εκτιμά αρκετά την έκθεση και έκανε μια επισήμανση. Ότι μίλησα περισσότερο για τι αρνητικέ πτυχέ σε αντίθεση με τι θετικέ. Υπάρχουν κάποια θετικά στοιχεία. Τα επανέλαβε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προφανώ εκφράζω την εκτίμησή μου. Όμω, αν θέλουμε να τολμήσουμε και κάπω παραπάνω, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να εξαλείψουμε τα αρνητικά στοιχεία. Γι' αυτό δίνουμε βάρο στα αρνητικά. Προσπαθούμε να επιλύσουμε προβλήματα. Συμφωνώ κατά πολύ μαζί σα λοιπόν ότι πρέπει οι κανόνε που συντάσσονται να εφαρμόζονται. Συμφωνώ και με την έννοια της επικουρικότητας για το πώς ε, μεταφέρονται οι νόμοι στις διάφορες χώρες και το θεωρώ επιτυχία. Επιτυχία που έστω και μέρη. Για μια φορά συμφωνούμε, κύριε Λάιναν. Ευχαριστώ. Πάντα είναι καλό να έχει κανείς μια θετική προσέγγιση και ένα θετικό ντοσία πλουστεύει την υπόθεση. Λοιπόν, μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου προθεσμία τροπολογιών στις 22-23 Ιανουαρίου θα συζητήσουμε την έκθεση πρωτοβουλίας και θα γίνει η ψηφοφορία στην Ολομέλεια Φεβρουάριο ή Μάρτιο. Ωραία, ολοκληρώσαμε και αυτό το σημείο και έτσι προχωρούμε στο τελευταίο του πρωινού που είναι το 8. Ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 88 παράγραφος 2 του κανονισμού, χρήση γαλακτικού οξέας για τη μείωση της μικροβιολογικής επιφανειακής μόλυνσης φαγίων βοηδών. Ε, δεν είναι και συναρπαστικό το θέμα, όμως πιστεύω ότι θα γίνει συναρπαστικό με τη συζήτηση. Και δίνω το λόγο στους συντάκτες καταρχάς αυτής της ένστασης. Η κυρία Λίντα Μακέβαν. Ευχαριστώ. Ο λόγος για τον οποίο έφερα το θέμα αυτό προς συζήτηση είναι διότι με πλησίασαν οργανώσεις καταναλωτών και εργαζόμενοι σε σφαγεία και επιθεωρητές κρεατών, ε, που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα ορίζεται ως υγειονομικό πρόβλημα από την Κομισιόν. Όμως, το θέμα ε, που συζητάμε σήμερα ε, δεν είναι ότι η Κομισιόν θέλει να αλλάξει τους υγειονομικούς κανόνες, αλλά είναι επειδή υπάρχει ε, μια εμπορική διαμάχη με τις Ηνωμένε Πολιτείε όσον αφορά την εισαγωγή βοηδών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν από μερικά χρόνια είχαμε απαγορεύσει την ε, χρήση, την έγχυση ορμονών στο βόλιο κρέας και ως μέρος της συμφωνίας που είχαμε τελικά συνάψει είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιτρέψει την εισαγωγή χιλίων τόνων αμερικανικού βο... βοήου κρέατος το οποίο δεν είχε ορμόνες. Όμως τελικά διαπιστώσαμε ότι είχε χρησιμοποιηθεί γαλακτικό οξύ κατά τη διαχείριση των σφαγίων. και δεν έχει, το, την έγκριση, έχει την έγκριση του FSA ότι είναι, της Αμερικανικής Υπηρεσίας ότι είναι ασφαλές, όμως πολλοί ε, ειδικοί οι οποίοι εργάζονται στην αγορά κρέατος μου είπαν ότι αν χρησιμοποιήσεις το γαλακτικό οξύ κατά τη διάρκεια της διαδικασίας όταν το κρέας είναι πάνω στην ε, στην αλυσίδα παραγωγής, τότε θα αντιμετωπίσει προβλήματα υγιεινής. Εάν το γαλακτικό οξύ χρησιμοποιείται στο τέλος της διαδικασίας Ας πούμε ότι έχουμε ένα σφάγιο, μπαίνει στην αλυσίδα δια σας. Ε, συνεχή επιθεωρητές ελέγχουν το σφάγιο και διαπιστώνουν χρήση γαλακτικού οξέως. Όμως, στα ευρωπαϊκά σφαγεία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μόνο καθαρό νερό, ενώ στις Ηνωμένε Πολιτείε επιτρέπεται η χρήση κατά τη διάρκεια επεξεργασίας του σφάγιου γαλακτικού οξέως. Η Κομισιόν λοιπόν έχει κάνει αρκετές προτάσεις. Στην αρχική πρόταση της Κομισιόν δεν θέλαμε να επιτρέψουμε ε, τη χρήση γαλακτικού οξέως κατά την επεξεργασία του σφαγίου, αλλά να το επιτρέψουμε μόνο στην απολύτως τελευταία φάση. Όμως, όπως σας είπα, στις Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιείται το γαλακτικό οξύ καθ' όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας του σφαγίου και γι' αυτό έχουμε υποβάλει και αυτή την ένσταση είναι μία επίμαχη, ένα επίμαχο θέμα και γι' αυτό ζήτησα να κάνουμε συζήτηση. Στο Συμβούλιο δεν υπάρχει πλειοψηφία για να στηρίξει την πρόταση της Κομισιόν. Μερικά κράτη-μέλη ψήφισαν κατά της, ε, την πρόταση της Κομισιόν στο τελευταίο Συμβούλιο και έχω το κατάλογο των χωρών αυτών που καταψήφισαν την πρόταση της Κομισιόν. Αυτή τη στιγμή οι αντίθετε κυβερνήσει είναι Γαλλία, Αυστρία, Ελλάδα, Λετωνία, Πολωνία. Ψήφισαν κατά της Κομισιόν. Ουγγαρία, Λουξεμβούργο, Φιλανδία απέσχον. Δεν υπάρχει λοιπόν πλειοψηφία. Τις ερχόμενες εβδομάδες οι υπουργοί θα ψηφίσουν και από ό,τι πιστεύω δεν θα υπάρχει πλειοψηφία στο Συμβούλιο υπέρ αυτή τη πρόταση. Εάν δεν υπάρχει στο Συμβούλιο θα παραπεμφθεί στην Κομισιόν προς απόφαση. Με άλλα λόγια, οι Υπουργοί δεν θα λάβουν απόφαση, δεν θα ψηφίσουν και πιστεύω ότι αυτό δεν είναι σωστό για τη δημοκρατία. Αυτά τα θέματα πρέπει να συζητώνται δημοσίως, πρέπει να έχουμε μια ανοιχτή συζήτηση. Το άλλο που θα ήθελα να ρωτήσω την Κομισιόν είναι από απόψεως υγιεινής Εάν η Κομισιόν πιστεύει ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε γαλακτικό οξύ, ε, γιατί δεν μας το έχει πει αυτό στο παρελθόν. Ποια, ποιο είναι το όφελος, το όφελος για τους καταναλωτές, δεδομένου ότι εδώ δεν τίθεται θέμα επισήμανσης, ότι το κρέας δηλαδή που έχει γαλακτικό οξύ, έχει γίνει επεξεργασία με γαλακτικό οξύ, ε, δεν θα το ξέρουν οι καταναλωτές. Οι εταιρείε όμως που χρησιμοποιούν το οξύ αυτό πρέπει να το δηλώσουν στην επεξεργασία των σφαγείων. Άρα λοιπόν ποιο το όφελος για τους καταναλωτές. Ξέρω ότι είναι μέτρο ε, εμπορικό, μέτρο του εμπορίου. και μπορεί η Κομισιόν να επιβεβαιώσει αν υπάρχει ακόμα απαγόρευση εισαγωγής ε, ευρωπαϊκού κρέατος στις ΗΠΑ λόγω της, ε, ε, του BSE, της παλιάς υπόθεσης στον κόδο εγκεφαλοπάθειας. Υπάρχει ακόμα λοιπόν αυτή η απαγόρευση από αμερικανικής πλευράς. Είμαστε λοιπόν ενώπιον ενός μέτρου που προτείνεται που δεν υπάρχει, δεν δημιουργεί όφελος για τους καταναλωτές ε, μια ουσία η οποία δημιουργεί μεγάλες επιφυλάξεις στους ειδικού του τομέα. Και ρωτώ την Κομισιόν, θέλετε να περιμένετε από εμά να πούμε απλώς ναι, ναι, το εγκρίνουμε. Εγώ αντίθετα νομίζω ότι οι συνάδελφοι πρέπει να σκεφτούν πολύ σοβαρά και να δούμε εάν θα επιτραπεί το γαλακτικό οξύ μόνο στο, στην τελευταία φάση επεξεργασίας, εάν επιτραπεί, μπορεί να μην επιτραπεί καθόλου. Το θέμα είναι γιατί να δημιουργήσουμε ένα πρόβλημα το οποίο δεν έχει δημιουργήσει πρόβλημα στην Ευρώπη ποτέ και γιατί να αλλάξουμε τα καλό κείμενα. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ την κυρία Μακέβαν. Η κυρία Ροτ Να προσθέσω κάτι σε αυτά που είπε η κυρία Μακέβαν. Δεν συζητούμε το θέμα της υγιεινής των τροφίμων. Συζητούμε το εμπόριο από εμπορική σκοπιά. Αν κοιτάξουμε τώρα ποιος προσπαθεί να πείσει ποιον και κοιτάξω τα πρόσωπα γύρω μου, Θα ξεκινούσα από τα υψηλότερα κλιμάκια και θα έλεγα ότι δεν βλέπω κάποιος να έχει πιστεί. Τι θέλουμε τελικά. Μια νέα εμπορική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ίσως αυτό είναι το σοβαρότερο σκέλος. Θα θυσιάσουμε το άλλο όμως. Πραγματικά εξεπλάγει όταν είδα ότι στην Επιτροπή της επετροπολογίας ανταλλάσσονταν πολλά έγγραφα, μεταξύ των οποίων μια πρόταση το γαλακτικό να χρησιμοποιείται μετά τους ελέγχους post-mortem και μόνο. Αυτό το αναφέρει η Λίντα Μακέβαν στο τέλος της, ε, του ψηφίσματος, του κειμένου. Δεν είναι όμως αυτή η πρόταση που έχουμε στα χέρια μας τελικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελπίζω να μας εξηγήσει γιατί έγινε αυτή η αλλαγή. Η απάντηση είναι ότι εάν χρησιμοποιείται μόνο μετά του post-mortem ελέγχου, δεν έχει πλέον κανένα συμφέρον για τι ΗΠΑ η χρήση του γαλακτικού ξέου. Δεν είναι ίσονο σημασία λοιπόν να σκεφτούμε ότι υπάρχει και επιστημονική γνωμοδότηση από την ΕΦΣΑ, η οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να επισημάνουμε στην εύσα της ε, ελλείψεις της. Έχουν τεθεί τέσσερα ερωτήματα και η ΕΦΣΑ απάντησε στα δύο. Στα υπόλοιπα είπε δεν έχουμε αρκετά στοιχεία, αλλά φανταζόμαστε ότι κάτι τέτοιο θα πρέπει να γίνει. Το μόνο στο οποίο αναφέρθηκαν είναι η ασφάλεια. Κανεί από εμά δεν λέει όμω ότι το γαλακτικό οξύ είναι επικίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. Όχι, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Δεν είναι ότι είναι επικίνδυνο για την, για την ανθρώπινη υγεία, ούτε τοξικό. Απλώς δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό σε περίπτωση που εξετάζουμε την υγιεινή των τροφίμων. Πρώτα απ' όλα μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Μπορεί να οδηγήσει σε παραμέληση της υγιεινής στα σφαγεία. Μπορεί να σκοτώνει τα μικρόβια τη στιγμή που χρησιμοποιείται, αλλά θα μπορούσε να θανατώνει και βακτήρια τα οποία μπορεί να, να είναι χρήσιμα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μεταφοράς λόγου χάρη. Και στη συνέχεια τη όλη αλυσίδα παροχή δεν θα είναι αξιόπιστε μετά οι δηματοληψίε που θα γίνονται. Όλα αυτά μας οδηγούν σε μια σαφή απάντηση. Εάν θέλαμε το γαλακτικό οξύ, ω Ευρωπαϊκή Ένωση θα είχαμε και από πριν τέτοια νομοθεσία. Κοιτάζω του εκπροσώπου τη Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ, που κάθονται εκεί στα έδρανα αυτά, με τη σοφία που διαθέτουν και την σχετική εμπειρογνωμοσύνη. Αλλά πείτε μα, τι βελτίωση θα προσφέρουν αυτά στην προστασία των καταναλωτών και την ε, υγεία των πολιτών. Δεν θα είχαμε κάποιο τέτοιο μέτρο αν χρειαζόταν. Γιατί πρέπει να θυσιάσουμε αυτέ τις προτεραιότητες στο βωμό τη Εμπορική Συμφωνία με τις ΗΠΑ. Ο κύριος Μαρτή θα είναι ίσως αρμοδιότερος για να μας εξηγήσει τις ε, διαστάσεις των προβλημάτων που εξετάζουμε. Πάντω, θυμάμαι τον αγώνα που είχαμε δώσει για τη χρήση των τεχνητών ορμονών εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση στι ΗΠΑ και θυμάμαι πώ ιτηθήκαμε. Θυμάμαι πώ ε, Ματία, εσύ από την περιοχή που έρχεσαι, αυτοκινητοβιομηχανία, είχε ασκήσει πιέσει. Από την πλευρά λοιπόν ε, της ε, γεννη των καταναλωτών δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Από την πλευρά την εμπορική ίσως δεν γνωρίζω όμω. Αλλά θα ήθελα να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Για κάτι που δεν θέλουμε να εφαρμόσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί κάνουμε θυσίες και το δίνουμε ως αντάλλαγμα για άλλους σκοπούς. Ευχαριστώ, Καλ Σλούτερ. Δεν έχω και πολλά να προσθέσω. Έχουμε εκθέσει τις αντιρρήσεις μας. Και όπως είπε και Ντάγμαρ, στην έκθεση δεν αναφέρονται όλες οι σχετικές πτυχές του θέματος. Η μικροβιολογική πανίδα και ο φυσιολογικός ανταγωνισμός πώς θα αφήσει περιθώριο στους παθογενείς παράγοντες, στους παράγοντες παθογένειας. Μήπως μειώνουμε τις προδιαγραφές υγιεινής και την ποιότητα του κρέατος που φτάνει τελικά στους καταναλωτές. Δεν έχω και πολλά να προσθέσω. Απλώς δεν μπορούμε κάθε φορά που διαφωνούμε με τις ΗΠΑ... να ακολουθούμε την προοπτική, την εμπορική. Είναι εμπορική η διαφωνία και πρέπει να κάνουμε αυτό που μας λένε. Όχι, πρέπει να ακολουθήσουμε τους δικούς μας νόμους, τις δικές μας επιστημονικές γνώσεις και να κάνουμε το σωστό. Και κάποιες φορές μπορεί όντως να υπάρξει και σύγκρουση με τις ΗΠΑ. Εγώ δεν μπορώ εδώ πέρα να άγομαι και να φέρομαι από τις ΗΠΑ. Εάν κάτι είναι σωστό ή λάθος, αυτό θα πρέπει να μας απασχολεί να πράξουμε το σωστό και να δεχτούμε τι συνέπειε. Ανέκαθεν του αποκαλούσαμε φίλου, θα πρέπει να ακούσουν τα επιχειρήματά μα, τα διαφορετική μα κουλτούρα, να μα ακούσουν και να τα αποδεχτούν. Φοβούμαι επίση, μάλλον δεν φοβούμαι ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να πλήξει τι εμπορικέ μα σχέσει. Δεν δικαιολογείται να αφήσουμε κατά μέρο την κοινή λογική για το πώ εξετάζουμε την υγιεινή των τροφίμων, την υγιεινή τη τροφική αλυσίδα και να μην κάνουμε τη σωστή επιλογή. Ευχαριστώ. Έχω έναν κατάλογο μιλητών και θα τον διαβάσω. Μήπω Corinne Chris Μήπως παρέλειψα κάποιον, τον κύριο Μπάκη, και κλείνει ο κατάλογος. Ε, παρακαλώ όλους τους συναδέλφους να είναι σύντομοι. Για να ακούσουμε και την απάντηση της Κομισιόν από τη Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ. Α, και τι έκπληξη και Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. Γι' αυτό παρακαλώ να είστε λίγο σύντομοι. Κυρία Ζόμερ, ευχαριστώ. Έχουμε θαυμάσιες υγειονομικές διατάξεις, όμως κάθε χρόνο έχουμε 320.000 περιπτώσεις ε, μολύνθεων από τρόφιμα. Άρα λοιπόν δεν είναι παράλογο να υιοθετήσουμε ένα επιπρόσθετο μέτρο Συμφωνώ με τη συνάλφο Ροτ Μπέρεντ ότι πρόκειται εδώ και για το εμπόριο και όχι μόνο αποκλειστικά για εμπορικά ζητήματα. Γιατί λοιπόν να μην επιτρέψουμε αυτό το φυσικό οξύ που υπάρχει και σε όλα τα τους μυς μας, εξού και οι κράμπες που πασαίνουμε. Ε, γιατί να μην χρησιμοποιήσουμε λοιπόν αυτή τη φυσική, φυσιολογική ουσία να χρησιμοποιήσει. Ε, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος στην επεξεργασία σφαγείων, με, ε, ιδίως ε, όταν γίνεται κοιμάς να επιμολυνθεί με βακτήρια και να γίνει επικίνδυνος για την κατανάλωση. Στο Συμβούλιο, ναι, δεν υπήρχε συμφωνία. Όμως υπάρχει σαφής πλειοψηφία στο Συμβούλιο, 14 κράτη-μέλη υπέρ της πρότασης και 4 αποχές. Οι αποχές δεν σημαίνει ότι ουσιαστικά είναι απόλυτα αντίθετες, ε, αντίθετα τα κράτη μελιά, μπορούμε να πούμε 18. Δεν μπορώ λοιπόν να πω ότι κατηγορηματικά το Συμβούλιο απέρριψε αυτή την πρόταση. Ε, το Συμβούλιο περιμένει να δει και την άποψη της Κομισιόν και νομίζω ότι αυτή είναι μια καλή εξέλιξη. Θέλω να τονίζω ότι μία από τις προϋποθέσεις στην πρόταση της Κομισιόν είναι ότι το τελικό δείγμα που πηγαίνει για μικροβιολογική εξέταση των σφαγείων ε, εξετάζεται ως προς την τήρηση των υγειονομικών κανόνων. Αυτό λοιπόν το δείγμα λαμβάνεται πριν από την επεξεργασία του σφαγείου με γαλακτικό οξύ. Άρα λοιπόν δεν είναι δυνατόν να έχουμε κακές πρακτικές, να εφαρμόζονται κακές πρακτικές στη φάση εισαγωγής του γαλακτικού οξέως. Άρα λοιπόν εφόσον το δείγμα το λαμβάνονται πριν, εδώ πρόκειται για ένα επιπρόσθετο, ένα συμπληρωματικό μέτρο. Δεν θέλουμε να καλύψουμε τίποτα, να μπουρδουκλώσουμε κάτι ε, και τονίζω ότι Χρειάζεται μία τεκμηρίωση για την επεξεργασία αυτή με γαλακτικό οξύ. Η παραγωγή τροφίμων, οι οποίοι είναι υπέρ της χρήσης του γαλακτικού ε, οξέως, πρέπει να τεκμηριώσουν την επεξεργασία αυτή και όταν προχωράει το σφάγιο στην επόμενη φάση επεξεργασίας να συνοδεύεται και από την τεκμηρίωση αυτή ε, αν η Κομισιόν μπορεί να μας ε, διαβεβαιώσει ότι αυτό θα ισχύει και για τα εισαγόμενα κρέατα και εισαγόμενα προϊόντα, τότε δεν έχω μεγάλες επιφυλάξεις. Δεν ανήκω σε αυτούς που ε, υπακούν τυφλά τις Ηνωμένε Πολιτείε. Πάντα έχουμε εμπορικού καυγάδες για την κλωνοποίηση, για τις ορμόνες, ένα σωρό μάχες έχουμε δώσει και διαφορές έχουν προκύψει, αλλά για μας δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα υιοθέτηση αυτής της πρότασης. Ε, δεν συμφωνώ με την ένσταση και προτείνω την απόρριψη της ένστασης. Ευχαριστώ. Η Κορίν Μπράσο. Σας ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ με τη στάση της Ντάγμαρ ε, και του Καρλ ε, Σλάιτερ. Είναι σαφές αυτή τη στιγμή ότι ασκείται πίεση από τον εμπορικό κλάδο και από την Γενική Διεύθυνση Εμπορίου, οι οποίοι επιθυμούν να τροποποιηθούν οι κανόνες μας. Πιστεύω λοιπόν ότι τα πράγματα είναι απολύτως ξεκάθαρα. Το ζήτημα το οποίο πρέπει να αναλύσουμε αυτή τη στιγμή είναι ποια είναι τα ωφέλη, αν υπάρχουν ωφέλη για τον Ευρωπαίο καταναλωτή. Είναι σαφές ότι το γαλακτικό οξύ δεν είναι επικίνδυνο. Κανείς δεν είπε όμως κάτι τέτοιο το άλλο στο παρελθόν. Αυτό που μας ενδιαφέρει να γνωρίζουμε είναι ποιες είναι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες θα χρησιμοποιηθεί. Το γεγονός ότι μειώνεται η μικροβιολιακή μόλυνση δεν σημαίνει ότι τα πράγματα βαίνουν αισίως. Ενδεχομένως ε, στο μέλλον να υπάρχουν και κάποιες άλλες χρήσεις ή πρακτικές. Να υπάρξουν και άλλες ουσίες που θα αρχίσουν να χρησιμοποιούνται ή που θα μας επιβάλλουν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Και νομίζω ότι όλα αυτά θέτουν κινδύνο όλες αυτές τις, προ... τις προσπάθειες που κάναμε τελευταία χρόνια προκειμένου να βελτιώσουμε τις συνθήκες στα σφαγεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ζήτημα λοιπόν αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να δούμε όμως τι κάνουν η δική μας η παραγωγή και τι γίνεται με το κρέας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάθε φορά στο παρελθόν που έχουμε χαλαρώσει τους κανόνες υγιεινής, πληρώσαμε ένα πάρα πολύ βαρύ τίμημα τόσο σε ανθρώπους όσο όμως και σε οικονομικό, κοινωνικό επίπεδο. Πρέπει λοιπόν αυτά να τα έχουμε κατά νου. Πίτερ Λίζε. Θα μιλήσω αγγλικά γιατί έχω πολλές σημειώσεις μπροστά μου γραμμένες στα αγγλικά. Το γαλακτικό οξύ είναι μια φυσική ουσία και ε, από ό,τι βλέπω η συγκέντρωση του είναι αρκετά χαμηλή σύμφωνα με τα στοιχεία που μας δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τουλάχιστον όσον αφορά τη χρήση που γίνεται στα ζώα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πάντως που γίνεται η συζήτηση αυτή και που ακούμε τα διάφορα επιχειρήματα. Το συζητήσαμε το ζήτημα αυτό και στη δική μου την πολιτική ομάδα, του ΑΕΛΚΑ. Ο πρώην συγητής μας για την βασική νομοθετική πράξη έφεσε ήδη κάποιο ρώτημα γραπτό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την οποία θα ήθελα να σας διαβάσω τώρα. Μας λέει ο κύριος Νέλταρτ, από ό,τι καταλαβαίνω, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χρήση του γαλακτικού οξέου στα σφαγεία επιτρέπεται τελικά μόνο στο τέλος της διαδικασίας της σφαγής, αφού έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες δείγματοληπτικές ε, αναλύσεις και έλεγχοι για την ε, μικροβολογική επιφανειακή μόλυνση. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω αν σωστά ερμήνευσα από ε, την πρόταση της Κομισιόν. Εν συνεχεία στο προσάρτημα ε, της Κομισιόν και ομιλώ τώρα γερμανικά, λέει ότι το γαλακτικό οξύ θα ε, χρησιμοποιείται ε, μετά από την ανάλυση των δοκιμών με μικροβιολογικά κριτήρια. Αλλά στο ψήφισμα λέει κάτι άλλο. Θα ήθελε η Κομισιό να μου διευκρινίσει τι ισχύει ακριβώς. Τι θα πει ε, δοκιμές post-mortem ε, είναι τα, η μισά κομμάτια του ζώου, ε, είναι νεκρά τα ζώα, έτσι δεν είναι, έχουν ψοφήσει, διότι έχουν σφαγεί. Τώρα είτε είναι το μισό ζώο είτε το τέταρτο του ζώου, post mortem είναι post mortem, θα πει μετά τη σφαγή. Λοιπόν, θα ήθελα να με εξηγήσει η Κομισιόν επίσης τι εννοεί με τα εκτιμώντας νη και πι. Τα αιτιολογικές σκέψεις. Ε, λέει ότι θα πρέπει να κατα τα πολεμήσουμε ένα συγκεκριμένο ζωήφιο το οποίο μπορεί να κάτσει πάνω στο κρέας ε, ε, και στο αιτιολογικό πι αναφέρει ότι μπορεί η επιμόλυνση να αυξηθεί και θέλω να μάθω τι εννοεί με αυτό. Το νι και το πι στα αιτιολογικά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ακούσω τι απαντήσει τη Επιτροπή σε αυτά που, είπε, που ρώτησε ο κύριο Λίζε. Και εγώ να κάνω τι παρατηρήσει. Υπάρχουν κάποιε ανησυχίε. Επειδή η βιομηχανία βοήου με τη σπογκόντια κεφαλοπάθεια πέρασε ζωφερέ στιγμέ και δοκιμάστηκε ιδιαίτερα με την εχνηλασιμότητα λόγω των πιέσεων και του Κοινοβουλίου και άλλων. Τώρα μην τους ε, κάνουμε να επιστρέψουν σε κακές πρακτικές ε, με τη χρήση γαλακτικού οξέως που κατά τα άλλα είναι μια φυσική ουσία και που επιτρέπεται από τον κανονισμό το 53 του 2004. Εδώ δεν φαίνεται να είναι βάσιμη η ανησυχία ως αυτό. Το δεύτερο όμως που θέλω να επισημάνω επειδή κάποιοι χάνιζαν ε, όταν μιλούσαμε για τις εμπορικές προτεραιότητες. Δεν θεωρώ ότι το εμπόριο είναι και κανένα παλιόλογο. Και το εμπόριο για τους πολίτες είναι σημαντικό και για τις θέσεις εργασίας. Οπότε, αυτό να το έχουμε υπόψη στη σημερινή μας συζήτηση. Σημαντική είναι και η προστασία των καταναλωτών, αλλά το ίδιο και το εμπόριο. Είναι ζωτική σημασία για τους ε, πολίτες μας. Οπότε, θα συμφωνήσω με την κυρία Σόμα εδώ και με, υπολείπους, ε, με τους υπολείπους. Η ΕΦΣΑ αποφάσισε ότι παλής. Αυτό λέει το πορισμά τη και με την κατάλληλη χρήση επιτρέπει, μπορεί να είναι επιτρεπτή. Θα θέλαμε λοιπόν την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά. Και για την εμπορική διάσταση. Έχει και ωφέλη το εμπόριο για την Ευρώπη και δεν σημαίνει ότι θα υποβαθμίσουμε τις δικές μας προδιαγραφές. Πρέπει να το βλέπουμε και σε αυτό το σκηνικό το θέμα αυτό. Και όντω η συζήτηση αυτή θα έπρεπε να, γίνει και δημοσίω, συμφωνώ εδώ. ο κανονισμό για τη χρήση του γαλακτικού οξέου και δεδομένων των πορισμάτων τη ΕΦΣΑ είναι κάτι που θα πρέπει να στηρίξουμε. Δεν ε, συμφωνώ λοιπόν με το ψήφισμα όπω το έχουμε μπροστά μα. Ο Davis. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ συμφωνούμε ότι είναι μια φυσική ουσία, ένα οξύ, ότι είναι ασφαλές και ότι αν επεξεργαστούμε, το χρησιμοποιήσουμε στην επεξεργασία δεν υπάρχει πρόβλημα. Η ΕΦΣΑ λέει ότι η χρήση του γαλακτικού οξέου βοηθάει στην αποτελεσματική διαχείριση στον απο, αποτελεσματικό έλεγχο των παθογενών μικροβίων δεν ε, δημιουργεί κανέναν κίνδυνο στους καταναλωτές, στην υγεία τους, αλλά μπορεί η χρήση τους να μειώσει σημαντικά την μικροβιολογική απομόλυνση. Γιατί λοιπόν ερωτώ η Κομισιόν, αφού έχει όλα αυτά τα καλά το γαλακτικό οξύ, δεν μας έχει μέχρι τώρα προτείνει νομοθεσία υποχρεωτικής χρήσης του. Μια πρόταση υποχρεωτικής χρήσης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τίθεται το εξής ερώτημα. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλάζει επί της ουσίας την ε, βασική αξία της υγιεινής, της τροφικής υγιεινής και σε ειδικά σε ό,τι αφορά το βόλιο κρέας. Επί... Θεωρητικά μάλλον όχι, γιατί το γαλακτικό οξύ θα μας επιτρέψει να έχουμε πρόσθετα μέσα για να βελτιώσουμε την ε, γηνή των τροφίμων, ιδίω του βοηού. Απλώς βρισκόμαστε σε μια τέτοια οικονομική συγκυρία όπου προκειμένου να μειωθεί το κόστος παραγωγής ίσως να υπάρχει τάση να γίνονται λιγότερες προσπάθειες για την υγιεινή των τροφίμων στην αρχή της όλης ε, αλυσίδας της φαγής, λόγου χάρη, γιατί προς το τέλος της διαδικασίας αυτής μπορεί κανείς να απαλείψει κάποιες αρνητικές διαστάσεις της όλης επεξεργασίας του κρέατος. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη αυτή τη διάσταση του θέματος, την οικονομική κατάσταση, την οικονομική κρίση που κάνει τον ανταγωνισμό να λαμβάνει ιδιαίτερη αξία, καταλαβαίνουμε τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τι βασικέ αρχέ τη υγιεινή των τροφίμων. Αυτό είναι το πραγματικό ερώτημα που πρέπει να θέσουμε στου εαυτού μα. Ακόμη και αν δεν είναι το αντικείμενο του κειμένου που εξετάζουμε. Η είσοδο στην ευρωπαϊκή αγορά κρεάτων που έτυχαν διαφορετικέ επεξεργασία στο αμερικανικό έδαφο από την σκοπιά τη υγιεινή των τροφίμων, όλα αυτά μπορεί να υποβαθμίσουν τι βασικέ αρχέ τη υγιεινή των τροφίμων τη δική μα αγορά, τη ευρωπαϊκή. Αυτό είναι το πραγματικό ερώτημα. Εδώ ε, συμμερίζομαι το αυτό που είπε η συνάδελφο η κυρία Σόμερ, αλλά στη σημερινή ε, οικονομική συγκυρία, μήπω ανοίγουμε έτσι το κουτί τη Πανδώρα και δημιουργούμε κινδύνους για τους συμπολίτε μας. Ερικ Μπάνκι. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, igyekszem elnök úr kérésének megfelelően. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Το όλο ζήτημα είναι πολύ δύσκολο και πολύπλοκο. Σίγουρα ασκείται μία πίεση στην Επιτροπή και σε εμάς. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα το οποίο δεν αναφέραμε ακόμα. Εκτιλήσεται μια ολόκληρη διαδικασία με τη χρησιμοποίηση του γαλακτικού οξέως που ουσιαστικά επηρεάζει και τον χρόνο κατά τον οποίο το προϊόν μπορεί να θεωρείται φρέσκο, νοπό προϊόν. Μπορούμε να πούμε ότι χρησιμοποιούνται κάποια βακτήρια προκειμένου να αυξηθεί η περίοδος χρήσης ενός προϊόντος, εν προκειμένου του κρέατος. Νομίζω ότι και αυτό θα πρέπει πάντως να εξετάσουμε. Την επίπτωση που μπορεί το γαλακτικό οξύ να έχει στην ποιότητα του κρέατος. Θα επιτρέψουμε εμείς μια τέτοια διαδικασία εφόσον στην πράξη υφίσταται. Και κάτι ακόμα. Τα σφαγεία τελικά έχουν το απαραίτητο επίπεδο ασφάλειας χρησιμοποιείται χρησιμοποιούνται απαραίτητα μέσα προκειμένου να είναι ασφαλή, να μην κινδυνεύουν από μολύνσεις. Τι γίνεται με τα σφαγεία αυτά τα οποία χρησιμοποιούν τελικά γαλακτικό γαλακτικόψη. Στη δική μου τη χώρα είχαμε πάρα πολύ σημαντικά προβλήματα ασφάλειας στα σφαγεία. Στην ε, Ουγγαρία βέβαια δεν ελήφθη μια συγκεκριμένη απόφαση, μολονότι αντιμετωπίσαμε προβλήματα. Πρέπει λοιπόν να καταφέρει η δική μας Επιτροπή να δώσει επιτέλους μια απάντηση και πιστεύω ότι τα επόμενα 20 χρόνια όλα αυτά τα ζητήματα ασφάλειας των τροφίμων θα συνεχίσουν να βρίσκονται στην πρώτη θέση ανησυχιών των πολιτών. Σε καμία περίπτωση λοιπόν θα πρέπει να πιστοδρομήσουμε. Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο λοιπόν στην Κομισιόν. Καταρχάς τη Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ είναι ο διευθυντής, ο κύριος Βαν Γκότεμ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Ας ε, διαβεβαίωσω όλα τα μέλη καταρχάς ότι η Ευρώπη έχει πιστεύω το υψηλότερο επίπεδο ε, ασφάλειας ε, τροφίμων στην, στον κόσμο και δεν θα το υπονομεύσουμε ποτέ ούτε θα μειώσουμε το επίπεδο ασφάλειας, ούτε θα παρακάμψουμε από τις ε, θεμελιώδεις αρχές μας, ούτε θα χρησιμοποιήσουμε ε, θα δημιουργήσουμε οποιοδήποτε κίνδυνο με τη χρήση του γαλακτικού οξέως. Πάντοτε θα ακολουθούμε την κείμενη νομοθεσία. Να σας θυμίσω μετά, τι έγινε μετά τη Λευκή Βίβλο για την ασφάλεια των τροφίμων. Διάφορες ε, οδηγίες υγειονομικές υιοθετήθηκαν και τέθηκαν ενισχύ which το 2006 και τώρα υπάρχει μια βασική προσέγγιση από τη φάρμα, από την παραγωγική μονάδα στο πυρούνι, στο στόμα δηλαδή, στο φαΐ. Ας τονίσω λοιπόν ορισμένες αρχές τις οποίες υιοθετήσαμε μα από το Συμβούλιο και ε, το Κοινοβούλιο. Καταρχάς η βασική ευθύνη ανήκει ε, στους, ε, στον παραγωγό, στον εμπορευόμενο και η ασφάλεια θα πρέπει να είναι εξασφαλισμένη καθ' όλη τη διάρκεια παραγωγής του τρόφιμου μέχρι να φτάσει στον καταναλωτή. Έπειτα υπάρχει και η αρχή του HCCP, δηλαδή την ανάλυση των κρισίμων σημείων ελέγχου. Πρέπει να εντοπίσουμε αυτά τα σημεία, τα κρίσιμα, στην τροφική αλυσίδα και να τα ελέγχουμε. Τώρα με τους κανονισμούς που εγκρίθηκαν το 2004, υπάρχει σαφής πλέον νομική βάση, ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγκρίνει και άλλε ουσίε που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό των σφαγείων πέραν των εγκεκριμένων. Έχει λάβει πολλέ αιτήσει σχετικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τουλάχιστον πέντε. Όμω, το γαλακτικό οξύ είναι το μόνο στο οποίο δώσαμε κάποια συνέχεια, διότι για τα υπόλοιπα υπήρξε αρνητική γνωμοδότηση από την ΕΦΣΑ, η οποία αναφέρθηκε πολλέ φορέ στην σημερινή συζήτηση. Το γαλακτικό οξύ δεν παρουσιάζει προβλήματα ασφαλείας ούτε ζητήματα αποτελεσματικότητας και αποτελεσματικό είναι και αυτό φάνηκε από την όλη συζήτηση και η ΕΦΣΑ αναγνωρίζει ότι όντως χρησιμεύει στην ε, περιορισμό της μικροβιολογικής μόλυνσης ε, στην επιφάνεια των σφαγείων. Ούτε λοιπόν ε, για το περιβάλλον υπάρχουν επιπτώσεις, ούτε για την υγιεινή. Και τα τέσσερα κριτήρια για το πληρούνται για το γαλακτικό οξύ. Δεν προκύπτει λοιπόν προφανή λόγο ώστε να μην προτείνουμε τη χρήση του. Όπω είπα, υπήρξαν και άλλε ουσίε για τι οποίε ζητήθηκε να χρησιμοποιηθούν είτε από τα βιομηχανία είτε από κυβερνήσει. σε αυτές δεν δώσαμε συνέχεια, δεν εξετάστηκαν για λόγους ασφαλείας. Νομίζω φάνηκε ξεκάθαρα και από τη συζήτηση ότι το γαλακτικό οξύ ως φυσική ουσία βρίσκεται και υπάρχει και στους μυς του ανθρωπίνου σώματος και στους δικούς σας όταν περπατάτε. Υπάρχει γαλακτικό οξύ εκεί, εκρίνεται και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως πρόσθετο για τα τρόφιμα. Έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΕΦΣΑ συστήνει τη χρήση γαλακτικού οξέω σε πολύ συγκεκριμένε συνθήκε βέβαια. Με συγκεκριμένη συγκέντρωση, θερμοκρασία, όπω αυτά περιγράφονται στο παράρτημα. Του, της πρότασης. Πέραν των απορισμάτων της ΕΦΣΑ, εμείς έχουμε προσθέσει κάποια κριτήρια. Όπως ότι θα πρέπει να χρησιμοποιείται στο σύνολο του σφαγίου των βοηδών, όχι στα μισά, στα τεμάχια Τετάρτου. Δεν θα μπορεί λοιπόν να χρησιμοποιείται σε τεμάχια κρέατος το γαλακτικό οξύ. Πού θα χρησιμοποιείται τώρα το γαλακτικό οξύ, μάλλον πότε θα χρησιμοποιείται το γαλακτικό οξύ. Αυτό είναι το θέμα της συζήτησης. Νομίζουμε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιείται εκεί όπου ο υπεύθυνο της ε, παραγωγής τροφίμων θεωρεί ότι είναι το πλέον αποτελεσματικό. Αυτό μας ενδιαφέρει και από την πλευρά των ελέγχων. Πλέον αποτελεσματικό. Κάθε σφαγείο που έχει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει υπόκειται στο πρόγραμμα HCCP, ε, οπότε υπάρχει και σχετικός έλεγχος από την αρμόδια αρχή, δίνει δυνατότητα στον ε, παραγωγό βάσει των γνώσεων που έχει με το πρόγραμμα HCCP, να καταλαβαίνει πού θα είναι πλέον αποτελεσματικό το γαλακτικό οξύ στη χρήση του. Δεν αντικαθιστά όμως το γαλακτικό οξύ καμία από τις δράσεις που πρέπει να αναλυθούν ούτε εμποδίζει τον έλεγχο της υγιεινής του κρέατος. Η δειγματοληψία στα σφάγια θα συνεχιστεί. Και ο έλεγχος ante και ο έλεγχος post mortem και, τα, και ολόκληρα τα σφάγια θα εξετάζονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το κρέας είναι ασφαλές. Εάν υπάρχει προφανής μόλυνση του σφαγίου, διότι δεν μπορεί να είναι αποστηρωμένα τα σφαγεία, δεν είναι μια αίθουσα χειρουργείου σε νοσοκομείο, σε περίπτωση μόλυνσης δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ούτε κατογαλακτικό οξύ. Τι εννοούμε τώρα με τη μόλυνση επιφανειακή μόλυνση εννοούμε. Βακτηρίδια που δεν είναι ορατά με γυμνόφθαλμο. Πριν αναπτυχθούν. Να θυμίσω στους ε, παρόντες εδώ ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε τουλάχιστον 4, είχαμε, έχουμε 4.000 κρούσματα ή κόλλη ετησίω. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Ξέρετε τι ζημιές προκαλεί και θα θυμάστε τι προέκυψε με τα σχετικά κρούσματα και την όλη κρίση που προέκυψε πέρσι στη Γερμανία. Έχουμε 400, 4.000 συγγνώμη, 4.000 κρούσματα στους ανθρώπους ετησίως. Τουλάχιστον βάσει των στοιχείων του ΑΣΕ. Αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης ότι θα θανατώνονται μαζί και τα καλά ε, βακτηρίδια. Μα δεν υπάρχουν καλά και κακά βακτηρίδια. Κάποια είναι πιο επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία από ό,τι άλλα. Αλλά το γεγονό ότι θα χρησιμοποιείται το γαλακτικό οξύ συνολικά θα περιορίζει τη μόλυνση στο κρέα. Είτε με τα καλά είτε με τα κακά βακτήρια, βακτηρίδια. Όπως ε, είπα και νωρίτερα όμως, δεν ε, υποκαθιστούμε κάτι εδώ. Προσθέτουμε ένα κλιμάκιο ασφάλειας, μια, ένα παραπάνω σκαλοπάτι ασφάλεια για τους καταναλωτές. Είναι μια ουσία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους παραγωγούς τροφίμων, δεν αποτελεί υποχρέωση. Και όπως αναφέρθηκε και στη συζήτηση, η επισήμανση, η ενημέρωση του επόμενου κρίκου στην αλυσίδα της τροφικής ε, παραγωγής προβλέπεται από την πρόταση. Οπότε, Πρόεδρε, μπορείτε να καθησυχάσετε τους συναδέλφους σας ότι η πρόταση αυτή και βάσιμη ήταν και δικαιολογημένη από την πλευρά της υγιεινής των τροφίμων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και δίνω το λόγο στο Γενικό Διευθυντή Trade, στον κύριο Ντεμάρτη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από τη Γενική Διεύθυνση λοιπόν Εμπορίου και εργαζόμενα στο παρελθόν και στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας. Γνωρίζω λοιπόν καλά για τα ζητήματα αυτά. Αυτό που είναι σαφές και δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή να επισέλθουμε σε περισσότερες λεπτομέρειες τεχνικές. Ακούσαμε πολλούς ευρωβουλευτές και όντως ξέρουμε ότι το γαλακτικό οξύ δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι μια κακή ουσία, είναι μια ουσία που χρησιμοποιείται, πρέπει να χρησιμοποιείται με το σωστό τρόπο και ότι αυτό κάνουμε, ακόμη υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις έκολη σαλμονέλα που εμφανίζονται πολλές φορές σε κάποια σφαγεία. Προσπαθούμε όμως με τη χρησιμοποίηση του γαλακτικού οξέους να μειώσουμε τον κίνδυνο που παρουσιάζουν τα βακτήρια αυτά. Πρέπει να σας πω όμως ότι σε καμία περίπτωση δεν υποθάλπτουμε αυτή τη στιγμή την προστασία της υγείας των πολιτών και ότι δεν υποχωρούμε σε καμία περίπτωση σε εμπορικές πιέσεις, σε καμία περίπτωση. Και ουδέποτε θα υπαναχωρούσαμε στους βασικούς μας κανόνες όσον αφορά την ε, υγεία όσον αφορά την υγεία των ζώων. Δεν είναι διαπραγματεύσιμοι οι κανόνες αυτοί για την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν είναι διαπραγματεύσιμοι επίσης και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε μία σαφή επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη η οποία καταδεικνύει, όπως ακριβώς έχει φανεί και στις Ηνωμένες Πολιτείες, πώς έχουν τα πράγματα αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν καταφέρει να προσαρμόσει τον υφιστάμενο καονισμό της με βάση την επιστημονική αυτή εμπειρογνωμοσύνη, καταλαβαίνετε ότι θα προκαλέσουμε αρκετούς αρκετέ αμφιβολίε στι Ηνωμένε Πολιτείε, οι οποίες δεν θα θέλουν να ξεκινήσουν εμπορικές διαπραγματεύσει μαζί μας. Αν δούμε τι έχουν γίνει και σε άλλες επιτροπέ, βλέπουμε ότι 18 κράτη-μέλη έχουν ταχθεί ήδη υπέρ της χρήσης που προβλέπεται στον κανονισμό αυτό. Εν 70% 350 εκατομμύρια, 70% δηλαδή του ευρωπαϊκού πληθυσμού εκπροσωπείται από τις χώρες αυτές. Αν δεν επιληθεί λοιπόν το ζήτημα αυτό, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, τι θα γίνει. Νομίζω ότι οποιαδήποτε πολιτική απόφαση είναι σωστή, αρκεί όλα τα χαρτιά να είναι επιτάπητος. Και πάλι δεν αναφέρομαι εδώ πέρα σε κάποιο παζάρεμα το οποίο λαμβάνει η χώρα. Ξέρετε ότι στην προηγούμενη θέση που είχα έκανα πάρα πολλές διαπραγματεύσεις και είναι σαφές ότι η συμφωνία στην οποία αναφερόμαστε είναι προσωρινή, θα καταγγελθεί όμως και θα επιστρέψουμε τελικά στην παλαιότερη κατάσταση που είχαμε, όπου θα υπάρχουν κυρώσει και ουσιαστικά είναι εμπορικό πόλεμο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωση και Ηνωμένων Πολιτειών. Και καθότι η φυστάμενη συμφωνία λύγει τον Ιούλιο, πρέπει κάτι να κάνουμε γρήγορα. Αυτή θα είναι η πρώτη επίπτωση του να μην αναλάβουμε δράση. Η δεύτερη επίπτωση θα είναι ότι οι προοπτικές να ξεκινήσουν συνολικές εμπορικές διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες ουσιαστικά θα εξαφανιστούν. Και σίγουρα αυτό θα πρέπει να το έχουμε κατά νου κάθε φορά που συζητάμε την απόφαση αυτή. Επαναλαμβάνω πάντω ότι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται εμεί να υπαναχωρήσουμε μπροστά στου βασικού μα κανονισμού. Δεν αποτελούν αυτοί οι κανονισμοί αντικείμενο διαπραγμάτευση στι εμπορικέ διαπραγματεύσει που έχουμε. Ο κανονισμό μα για του γενετικά τροπημένου οργανισμού, ο κανονισμό μα για τι ορμόνε, η απαγόρευση των β ανταγωνιστών δεν πρόκειται επίσης να τεθεί επιτάπητος. Επίσης ο κανονισμός μας για την κλωνοποίηση δεν πρόκειται να ανοίξει σε καμία περίπτωση και δεν θα αποτελέσει αντικείμενο παζαρέματο πραγμάτευσης με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Δεν υφίστανται λοιπόν τα επιχειρήματα αυτά και ούτε υπάρχουν οι σχετικέ ανησυχίε. Σε καμία περίπτωση δεν θέτουμε να αμφιβόλο του παραγωγού, του κτηνοτρόφους βόηου κρέατος, τους παραγωγούς βόηου κρέατος. Μίλησα μάλιστα με μία υπουργό στην αρμόδια επιτροπή, η οποία δεν αναφέρθηκε στις ε, ανησυχίες που έχει για τον καταναλωτή, αλλά περισσότερο στις ανησυχίες που υπάρχουν για τους παραγωγούς βοηού κρέατος. Εμείς πάντως σε κάθε περίπτωση στις διαπραγματεύσεις που θα έχουμε τις ΗΠΑ θα λάβουμε υπόψη μας τα συμφέροντα και τις ανησυχίες που έχουν οι παραγωγοί, οι Ευρωπαίοι παραγωγοί βόηου κρέατος. Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να επιτρέψουμε μια ελεύθερη χαλήνοτη πρόσβαση βόηου κρέατος από τις ΗΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα υπάρχουν συγκεκριμένε ποσοστώσεις. Αυτά είχα να σας πω και θα πρέπει να γνωρίζετε ότι όλα τα επιχειρήματα θα χρησιμοποιηθούν, όλοι οι τομεί θα είναι ξεκάθαροι, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να ληφθεί μια απόφαση η οποία θα θέτει εν κινδύνο συγκεκριμένους τομείς Ευρωπαϊκή οικονομία. Το πιο σημαντικό δεν είναι τόσο πολύ να δούμε αυτή τη στιγμή αν θα μιλάμε για pre-mortem ή post-mortem επιθεωρήσεις, αλλά τι μπορούμε να κάνουμε προκειμένου ουσιαστικά και πραγματικά να προστατεύσουμε τους καταναλωτές μας. Ευχαριστώ. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος ε, της συζήτησης. Κάτι θα πω ακόμα. Ευχαριστώ τους ε, προλαλήσαντες, ε, τέλος πάντων που απάντησαν σε ορισμένες ερωτήσεις, σε ορισμένες της Λίντας δεν απαντήθηκαν. Δεν ξέρω τι θέλετε να δώσουμε άλλα πέντε λεπτά να... Επαναλάβω τις ερωτήσεις. Η Λίντα Μακέβαν. Ήταν η ερώτηση του κυρίου Λίζε για τη φάση ακριβώς, ποια θα είναι η συγκεκριμένη φάση επεξεργασίας όπου θα επιτραπεί η χρήση του οξέως. Από ό,τι κατάλαβα είχατε μία απόφαση α, αλλά μετά την αλλάξατε και τώρα έχετε μία άλλη απόφαση. Ε, στην αρχή είπατε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, τώρα λέτε μόνο στη φάση. Πού ακριβώς λοιπόν, στην τελευταία φάση. Και εν συνεχεία, αυτά που ρώτησε ε, ο κύριος Ντέιβιτ, εάν είναι τόσο καλή ιδέα, γιατί δεν γίνεται υποχρεωτική η χρήση. Ο κύριος Βον Γκόταμ μπορεί να απαντήσει παρακαλώ. Ευχαριστώ. Όπως σας είπα, η πρόταση χρήσης του γαλακτικού οξέως δεν αντικαθιστά τίποτα, είναι μία ε, προσθήκη και μία προϋπόθεση εφαρμογής του γαλακτικού οξέως είναι ότι γίνεται υπολεγόμενες ελεγχόμενες συνθήκες ε, όπως διαβλέπει το σύστημα ε, EHCCP, το σύστημα αυτό διαχείρισης. Όπως σας είπα, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σφαγής, οι αρμόδιες αρχές, οι επισερωτές θα πρέπει να κάνουν δειγματοληψία και αυτή η δειγματοληψία ε, είναι ακριβώς αυτή την κρίσιμη φάση, την κρίσιμη στιγμή και δεν θα με αλλάξει. Έτσι ώστε η αρμόδια αρχή θα είναι σε θέση να δώσει το έχει καλός για τη χρήση του αξέως στην κατάλληλη στιγμή. Θα πρέπει βεβαίως να υπάρχει η ευκαιρία όταν διαπιστωθεί ο κίνδυνος επιμόλυνσης. Δεν λέω ορατής μόλυνσης, ε, αυτή διαπιστώνεται στο σφαγείο και δεν επηρεάζει το γαλακτικό οξύ αν υπάρχει ορατή επιμόλυνση. Αλλά όταν υπάρχει ο κίνδυνος μη ορατής, τότε θα πρέπει να δοθεί το πράσινο φως και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί το γαλακτικό οξύ. You talked about some... Μιλήσατε για τη δειγματοληψία σφαγίων αλλά από ό,τι ξέρω εγώ για την αρμόδια νομοθεσία, θα πρέπει να υπάρχει τυχαία δειγματοληψία του κρέατος ε, στο τέλος της ε, γραμμής επεξεργασίας. Ενώ η Κομισιόν τώρα προτείνει και λέει ότι ε, το κρέας το οποίο έχει τύχει επεξεργασίας με το γαλακτικό οξύ δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο δειγματοληψίας. Άρα λοιπόν στην αρχή της διαδικασίας η μονάδα ε, σφαγίου θα πρέπει να διαπιστώσει ποια σφάγια ε, σε ποια σφάγια θα χρησιμοποιηθεί γαλακτικό οξύ και σε ποια όχι, εφόσον δεν μπορεί πλέον στα σφάγια με γαλακτικό οξύ να γίνει δειγματοληψία στο τέλος. Άρα λοιπόν ποιο το νόημα πλέον της διάταξης που λέει ότι θα πρέπει να γίνουν τυχαίοι δειγματοληψίες, να επιτρέπεται δηλαδή η Τυχαία δειγματοληψία. Άρα καταργείται αυτή η διάταξη. Ο πρόεδρος. Παρακαλώ απαντήστε σύντομα, στα αγγλικά. Yes, thank you. <clears throat> Very short. So, so there is an χωρίς, χωρίς διερμηνία. Θα σταματήσει η διερμηνία. per week. Soldiers are not obliged to use lactic acid. They may choose to work half a day